Buenos días. Si les Καλή σας μέρα. Εάν συμφωνείτε μπορούμε να ξαναρχίσουμε έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη χθεσινή μας συνεδρίαση και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ε, ακρόασή μας σχετικά με την αξιολόγηση. Το θέμα μας ε, είναι ένα θέμα το οποίο ήδη συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, όπου συζητήσαμε με τον κύριο Νταρή αυτή η ακρόαση βασίζεται και σε σχέση με τις, ε, τους οίκους αξιολόγησης ε, πιστοληπτικής φερεγγιότητας. Αν συμφωνείτε, ξεκινάμε με την κυρία Ελένα Ρώσα, ε, εκτελεστική διευθύντρια του της Μονάδας για τις Ευρωπαϊκές Αγορές. Έχετε, καλώς ήρθατε, έχετε τον λόγο σας. Υπενθυμίζω, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα πρώτα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα για να σκιαγραφίσω τις απόψεις της ΕΣΜΑ σε σχέση με τους οίκους αξιολόγησης ε, φερεγγιότητας. Θα ξεκινήσω τις σύντομες παρατηρήσεις μου λέγοντας δύο λόγια για το έργο όπως ε, βρίσκεται σήμερα της ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην φάση της υλοποίησης ε, των διατάξεων των τροποποιήσεων και τροπολογιών της ε, TRA2. Ιδιαίτερα από την 1η Ιουλίου 2011 η ΕΣΜΑ έχει ευθύνες για την καθημερινή εποπτεία των, των οίκων αξιολόγησης με την καταχώρηση των κυριότερων CRA από τον Οκτώβριο πέρσι η ΕΣΜΑ ξεκίνησε άμεσα τα εποπτικά βήματα. Είχαμε μία πρώτη εποπτεία των CRA στον Δεκέμβριο 2011 και αναμένεται ότι θα δημοσιευθεί κατά το, τους πρώτους μήνες ε, φέτος ε, το, η έκθεση αυτή. Επίσης ε, θα έχουμε και τα στοιχεία εκείνα τα οποία εμπεριέχονται στα εργαλεία του κανονισμού ε, με την βάση δεδομένων που είναι ένα ε, σημαντικό μέσο. Επίσης βρισκόμαστε στην διαδικασία της αξιολόγησης του ρυθμιστικού πλαισίου κάποιων μη ευρωπαϊκών χωρών και για την πιο εύλογη συνεργασία όσον αφορά τα εποπτικά σώματα, κάτι το οποίο θα διασφαλίσει ότι η υιοθέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αξιολογήσεων των τρίτων χωρών για αριθμιστικούς σκοπούς θα είναι εφικτό να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας προχωρήσω τώρα και ας κάνω λόγο για τις προτάσεις CRA3 που βρίσκονται επί Έχουμε αρκετές από αυτές τις διατάξεις που ε, δημιουργούν ένα υποπτικό πλαίσιο Ξεκινούμε πρώτα με τις ε, διατάξεις, ε, με τις ρήτρες ε, για την δημοσίευση και αποκάλυψη στοιχείων όσον αφορά τα μέσα τα οποία θα πρέπει να υποχρεώνουν τις τους εμπλεκόμενους να αποκαλύπτουν στοιχεία και δεδομένα τα οποία είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Επιπλέον θα πρέπει να αποκαλύπτεται στην ΕΣΜΑ το τέλος ή τα τέλη τα οποία έχουν καταβληθεί για τις πολιτικές αυτές. Μια άλλη σημαντική συνεισφορά στην νέα αυτή πρόταση αφορά την πρόληψη συγκρούσεων ε, συμφερόντων. Αυτή η διάταξη προβλέπει ότι δεν θα υπάρχουν αξιολογήσεις όταν ο κυριότερος μεριδιούχος θα έχει συμφέροντα στον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης ή όταν υπάρχουν μεριδιούχοι με τέτοια συμφέροντα. Επίσης θα περιορίζονται στις δυνατότητες που θα έχουν για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Με ενδιαφέρον εξετάζουμε την πρόταση σε σχέση με την CRA. Ενώ είναι σημαντικό να έχουμε σωστές διατάξεις σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση των συγκρούσεων ε, συμφερόντων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Ένας άλλος τομέας που θεωρώ εγώ είναι θετικός είναι η πρόταση που απαιτεί μια ε, εναρμονισμένη κλίμακα αξιολόγησης ε, σε σχέση με την CRA μελλοντικά μπορεί να υπάρχει ένα όριο στην δυνατότητα της συμμετοχής στην αγορά και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων. Η ενιαία κλίμακα αξιολόγησης θα δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για όλες αυτές τις αξιολογήσεις. Τέτοιου είδου μέτρα θα συνεισφέρουν για τη διαφάνεια, τη διαλειτουργικότητα και την συγκρισιμότητα των αξιολογήσεων και θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό. Επιπλέον, η πρόταση αυτή είναι επικοδομητικό ότι προτείνει ότι ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να ε, αντιμετωπίζουν θέματα ευθυνών και ε, προσφυγών. Ένα σύστημα ρύθμιση των, ε, ευθυνών, αυτών θα συνεισφέρει ώστε η CRA να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με τα όσα γινόντουσαν στο παρελθόν. Επιπλέον, η πρόταση θα διασφαλίσει αξιόπιστες αξιολογήσεις από όλες τις ε, CRA που όπως υστερότερα ε, θα επεξηγήσω θα μπορέσει να οδηγήσει σε ωφέλη Παρότι συμφωνούμε με την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχουν αξιόπιστοι κανονισμοί στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την διαλειτουργικότητα και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ εθνικών συστημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κίνητρα που απορρέουν από την μερική ε, εφαρμογή, ώστε να υπάρχει μια ε, εξισορροπημένη μέθοδος ε, εφαρμογής. Επιτρέψτε μου τώρα, έχοντας αναφέρει κάποιες από τις προτάσεις που θα είναι επωφελής να προχωρήσω και να αναφέρω κάποια πράγματα στα οποία πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις προτάσεις CRA3 για τις επιπτώσεις που πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να εξεταστούν. Πρώτα απ' όλα η πρόταση εισάγει απαιτήσει για την ΕΣΜΑ να αξιολογεί σχέδια μεθοδολογικά, μεθοδολογικής προσέγγισης. Η πρόταση σωστά αναφέρει ότι η ΕΣΜΑ θα συνεχίσει να αναφέρεται στα ίδια κριτήρια για την αξιολόγηση, όπως υπό τον υφιστάμενο ενισχύ κανονισμό, που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει ανάμειξη τρίτων σε αυτές τις διεργασίες. Επειδή όμως ε, η νέα αυτή πρόταση για τον ρόλο της ΕΣΜΑ θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές εντάσεις ε, με τις απαιτήσει της μη ανάμειξης και της ανεξαρτησίας, μία πιθανή εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η ε, τα πρότυπα να θα μπορούσαν να είναι τα πρότυπα ε, βιομηχανικής ε, εφαρμογής και εποπτείας ώστε να διασφαλιστεί ότι μέσω των CRA θα γίνεται σεβαστή αυτή η προσέγγιση. Δεύτερον, η προσέγγιση CRA 3 έχει και τις, ε, τα στοιχεία για την, ε, τις αναλύσεις ε, υποχρεωτικής ανακύκλωσης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός στον τομέα CRA που μπορεί να έχει περιοριστεί μέσω των προσεγγίσεων, των αξιολογήσεων κατά το παρελθόν. Τούτου λεχθέντος, τουλάχιστον βράχει πρόθεσμα, υπάρχει ένας κίνδυνος ότι θα μπορούσε να υπάρχει ανταγωνισμός με την προσφορά υψηλότερων αξιολογήσεων ή με την μείωση τιμών. Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις. Γι' αυτό ε, εφόσον ε, μικρότερες ε, CRAs θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία ανακύκλωσης θα έχουν όλη την αναγκαία πραγματογνωμοσύνη όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του έργου. Πράγμα το οποίο θα τους δώσει την ευκαιρία να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων που είναι ιδιαίτερα απαιτητικέ. Και ίσως αυτό μεσοπρόθεσμα να μπορεί να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες, ωστόσο μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν ωφέλη. Πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αυτοί οι κίνδυνοι για αυτή την ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την αξιολόγηση αγορών. Επίση, θα ήθελα να αναφέρω μια άλλη πρόταση που θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΣΜΑ να δράσει όσον αφορά την επικέντρωση των σχετικών κινδύνων. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επικέντρωση ε, στην αγορά και οι κίνδυνοι που απορρέουν. Αυτό αναφέρεται στο έργο των εποπτικών αρχών για τον ανταγωνισμό. Ενώ φυσικά η ΕΣΜΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το έργο το οποίο έχει επομιστεί από τους νομοθέτες, θα πρέπει με ιδιαίτερο τρόπο να αναπτυχθεί μεθοδολογία για την αντιμετώπιση των συμπυκνώσεων στις αγορές. Πέρα από αυτό θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ΕΣΜΑ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το δύσκολο έργο του, τον, της αντιμετώπισης διαφορετικών α, αντικρουόμενων στόχων Αφενός δηλαδή την ε, συμβατότητα και από την άλλη πλευρά την, ε, τα θέματα ανταγωνισμού. Έχοντας ε, άμεση αναφορά στις διαδικασίες της ΕΣΜΑ, που βρίσκονται υπό εξέταση υπό τα στελέχη της ΕΣΜΑ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η πρόταση απαιτεί από την ΕΣΜΑ την αναθεώρηση μέχρι την 1η Ιουνίου 2014 της συμμόρφωσης των τρίτων χωρών όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν εισαχθεί μέσω του CRA3. Ο κανονισμός ο οποίος βρίσκεται ενισχύει ήδη απαιτεί από την ΕΣΜΑ να προβεί σε ένα τέτοιο ενεξελίξη έργο όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα όσον αφορά το νομικό πλαίσιο τρίτων ε, χωρών που ε, επιτυγχάνει ε, συγκρίσιμους στόχους ή συμμορφώνεται με τους στόχους αυτούς. Με τις προτάσεις CRE3 έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και προβλέπεται σε σχέση με τις τροπολογίες η αξιολόγηση που όχι μόνο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες, μια και αυτή τη στιγμή πολλές από αυτές τις προτάσεις δεν αποτελούν τμήμα της, ε, ε, του 20, ε, της λέσχης των 20 και της, του πλαισίου ΑΙΟΣΚΟ. Επίσης θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης τρίτων χωρών, διεργασία στην οποία εμπλεκόμεθα, εμπλεκόμεθα υπό τον υφιστάμενο κανονισμό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι πρέπει να επαναλάβω το μήνυμα το οποίο διατύπωσα στο παρελθόν Πρέπει να δοθεί επαρκή χρόνο στην ΕΣΠΑ ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στι τεχνικέ προδιαγραφέ και πρότυπα. Η προθεσμία είναι η 1η Ιανουαρίου 2013 και είναι πολύ στενό και πιεστικό αυτό το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την τελική έγκριση του κανονισμού. Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει επαρκές χρονικό διάστημα για αυτό το στόχο. Ιδανικό θα ήταν να έχει ένα χρόνο στη διάθεσή τη ώστε να συμφωνηθούν και να διατυπωθούν οι τεχνικέ αυτέ προδιαγραφέ ώστε να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα που εσεί και οι άλλοι νομοθέτε απαιτούν θα μπορέσει να είναι ένα εφικτό έργο για μα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρος και ευχαριστούμε πολύ για το ότι προσαρμοστήκατε στο χρονικό όριο της παρεμβασή σας. Ο επόμενος θα έχει πέντε λεπτά. Είναι ο κύριος Γκάλιαρ που είναι οικονομολόγος. έχει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που παρίσταστε. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας εδώ θα ασχοληθώ στην παρουσίασή μου με τρία συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν την αρχή της εκπεριτροπής αξιολόγησης και τον ανταγωνισμό στον κλάδο των οίκων αξιολόγησης. Δεύτερον την ποιότητα των αξιολογήσεων και τρίτον την υπερβολική εξάρτηση από αξιολογήσεις. Με συγχωρείτε. Αν μπορείτε με λίγο βραδύτερο ρυθμό για να μπορούν οι διερμηνείς να σας παρακολουθήσουν, για να μπορέσουν να διερμηνεύουν αυτά τα οποία λέτε. Um, Το πρώτο θέμα είναι η αρχή της εκπεριτροπής αξιολόγησης και ο ανταγωνισμός τον κλάδο των οίκων αξιολόγηση. Νομίζω ότι υπάρχουν βεβαιότητε σχετικά με τι στρατηγικέ των οίκων αξιολόγηση, εάν υιοθετηθεί ο κανόνα τη εκπεριτροπή αξιολόγηση. Εάν ε, ε, ε, υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις. Θα σταματήσει ο οίκος αξιολόγηση να αξιολογεί τον εκδότη μετά την τριετή περίοδο ή θα συνεχίσει την αξιολόγηση χωρίς να του έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Αν σταματήσει την αξιολόγηση ε, μόλις τελειώσει η τριετής περίοδος, υπάρχει κίνδυνος ε, η νέα αξιολόγηση που θα δοθεί στον εκδότη να είναι σημαντικά υψηλότερη ή χαμηλότερη από την προηγούμενη. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ξεκινήσει μια τεχνητή αναβάθμιση ή υποβάθμιση της αξιολόγησης ε, της διαβάθμισης του εκδότη. Αν αξιολογηθεί από κάποιον άλλον, οίκοαξιολόγησης ε, θα μετριαστεί αυτή η επίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο οίκος αξιολόγησης δώσει ε, αξιολόγηση χωρίς να του ζητηθεί όταν τελειώσει η τριετής περίοδος, ε, δεν θα έχει μεγάλη επίπτωση αυτός ο κανόνας, γιατί πολλοί οίκοι αξιολόγησης, οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης μπορούν να συνεχίσουν να αξιολογούν τον εκδότη χωρίς να του έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Και ως αποτέλεσμα, όταν περάσει η τριετή περίοδος, ο οίκος αξιολόγηση θα έπρεπε να απαγορεύει απαγορεύεται να παρέχει αξιολόγηση ε, για τον εκδότη, είτε του ζητηθεί είτε όχι. Παρ' όλα αυτά, αυτή η αρχή τη εκπεριτροπή αξιολόγηση μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, διότι θα εμποδίζει τη σύγκριση των αποδόσεων των οίκων αξιολόγηση, διότι η περίοδο κατά την οποία ένα εκδότη αξιολογείται ταυτόχρονα από διάφορου οίκου αξιολόγηση θα είναι μικρότερη διάρκεια. Επομένως, εγώ έχω μια εναλλακτική λύση προς την αρχή της εκπεριτροπής ε, αξιολόγησης και η πρότασή μου είναι η εξής. Για κάθε ε, περιοχή αξιολόγησης, ε, ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα πρέπει να υπολογίζει ένα κατόφλι, ένα ανώτατο ποσοστό, πέραν του οποίου θα πρέπει να απαγορεύεται για τους, στους οίκους αξιολόγησης να αυξάνουν την κάλυψη αξιολογήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ε, οι εκδότες στους οποίους δεν παρέχεται αξιολόγηση και οι εκδότες που ήδη έχουν αξιολόγηση αλλά που θέλουν και μία πρόσθετη αξιολόγηση θα πρέπει να ζητούν αξιολόγηση από ένα μικρό οίκο αξιολόγηση και όχι από αυτούς που ξεπερνάνε το κατόφλι. Αυτό είναι ένα μέτρο αντιτράστ κατά κάποιο τρόπο που θα, δώσει, ε, που θα προωθήσει τον ανταγωνισμό. Τώρα, δεύτερο σημείο, η ποιότητα των ε, αξιολογήσεων. Αξιολογήσεις είναι αξιόπιστες εάν οι οι αξιολόγηση έχουν μεγάλο αριθμό προσωπικού. Εάν ε, οι αξιολογήσει είναι συνεπεί προβλέψιμε και σταθερές, αν είναι ακριβεί και αν οι οίκοι αξιολόγηση επιβλέπονται στενά από, το, από την ΕΣΜΑ. Ε, υποστηρίζω την, το σχέδιο πρόταση της Επιτροπής που λέει ότι η οίκη αξιολόγησης πρέπει να είναι διαφανής όσον αφορά το προσωπικό στο οποίο αναθέτουν την αξιολόγηση διαφόρων κινήτων αξιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο αυτός ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός. Σήμερα ένας αναλυτής μπορεί να παρακολουθεί μέχρι και 30 εκδότες ομολόγων ως πρωτεύων ή δευτερεύων αναλυτής. Αυτός ο ρυθμός δεν είναι λογικό, διότι δεν έχει χρόνο ένα αναλυτή για να παρακολουθεί κάθε εκδότη. Προτείνω λοιπόν ένας αναλυτής να μπορεί να παρακολουθεί μέχρι 15 εκδότες ως πρωτεύων και δευτερεύων αναλυτής. Μια πρόταση που θα οδηγήσει σε αύξηση του προσωπικού των οίκων αξιολόγησης. Δεύτερον, για την προβλεψιμότητα και σταθερότητα των αξιολογήσεων πρέπει να βελτιωθεί ε, ε, και θα βελτιωθεί εάν πριν από οποιαδήποτε υποβάθμιση δοθεί μια αρνητική προοπτική ή αρνητική παρακολούθηση και πριν από την ε, αύξηση της αξιολόγησης μια θετική προοπτική. Κατά αυτόν τον τρόπο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 θα ε, ε, υπάρχει καλύτερη προετοιμασία και γι' αυτό είμαι κάπως διστακτικός για την πρόταση της Επιτροπής που λέει ότι θα πρέπει να δίδονται αξιολογήσεις στις πιστοληπτικές ικανότητες πιο συχνά, κάθε 6 μήνες αντί κάθε 12 μήνες. Τρίτον, οι προτάσεις μου για την ποιότητα και ακρίβεια των αξιολογήσεων ε, είναι οι εξή. Θα πρέπει να εξετάζουν οι ρυθμιστικές αρχές την απόλυτη ποιότητα των αξιολογήσεων και την σχετική τους ποιότητα. Κάθε αξιολόγηση θα πρέπει να δημοσιεύει τον κίνδυνο κίνδυνο χρεοκοπίας για κάθε τομέα και τα ποσοστά ακρίβειας για κάθε τομέα. Οι μεγάλοι οργανισμοί αξιολόγησης ε, ε, επί χρόνια δημοσιεύουν ε, τα ποσοστά κινδύνου χρεοκοπία, αλλά όχι τα ποσοστά ακρίβεια. Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχόλια για αυτά τα αποτελέσματα και να τονίζει τι αδυναμίες κάθε οίκου αξιολόγηση. Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί την απόδοση κάθε οίκου αξιολόγηση, συγκρίνοντα τα ποσοστά τα οποία δημοσιεύουν. Πρέπει να υπάρχει κοινή περίοδο αναφορά, ένα κοινό δείγμα και σύγκριση αυτών των δικτών. Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει σχόλια σχετικά με τα ισχυρά και αδύναμα σημεία κάθε οίκου αξιολόγηση. Και τέταρτον, η πρόταση τη Επιτροπή δηλώνει ότι οι οίκοι αξιολόγηση θα πρέπει να υποβάλουν τι μεθοδολογίε του στην ΕΣΜΑ για να αξιολογηθούν. Αυτέ οι νέε μεθοδολογίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν εγκριθεί από την ΕΣΜΑ. Είναι θετική αυτή η πρόταση και θα βελτιώσει τη διαφάνεια. Περνώ τώρα στη μείωση τη εξάρτηση από τι αξιολογήσει των οίκων αξιολόγηση. Η χρήση των αξιολογήσεων ε, πολλές φορές είναι υπερβολική και οι ε, αξιολογήσεις ε, δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τους μικρούς επενδυτές. Ως αποτέλεσμα, οι αξιολογήσεις δεν μπορούν να υποκαθιστούν τη δέουσα επιμέλεια των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και σημαντικά ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να έχουν δικούς τους, δική τους αξιολόγηση, θα πρέπει να ελέγχουν και να διασταυρώνουν αυτές τις εσωτερικές αξιολογήσεις και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές η ΕΣΜΑ θα πρέπει να ελέγχει την απόδοση αυτών των μοντέλων αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα. Η χρήση τέτοιων ε, αξιολογήσεων θα πρέπει να εξαρτάται από τη ρυθμιστική έγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Μακότο Ούτσι και κύριο Σύμβουλο ε, τη Ιαπωνική Υπηρεσία Αξιολόγηση. Πέντε λεπτά έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι και κύριοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχήν θα ήθελα να σας κάνω μια παρουσίαση της δικής μου εταιρεία τη JCR. Η Ιαπωνική εταιρεία αξιολόγηση. Ε, λειτουργούμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια στην Ιαπωνία και έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Καταρχήν για το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων και για το μοντέλο αμοιβή. Όντως, το μοντέλο του ότι πληρώνει ο εκδότης περιέχει ενδεχομένω σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά η εναλλακτική λύση, δηλαδή το μοντέλο του ότι πληρώνει ο επενδυτή, ε, η εξέλιξη ε, ε, του μοντέλου όπου υπάρχει εσωτερική αξιολόγηση στον επενδυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένο συγκρούσεων συμφερόντων. Θα σας πω ότι είπε ο καθηγητής Γκουστάβο Μάνσο του MIT ο οίκο αξιολόγηση θα πρέπει όχι μόνο να δίνει μια ακριβή παρουσίαση τη εταιρεία ή τη χώρα όσον αφορά την επιστολυτική ικανότητα, αλλά πρέπει επίση να λαμβάνει υπόψη το ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η τη χωρα οσον αφορα την πιστοληπτικη ικανοτητα αλλα πρεπει επιση να ή η χώρα η οποία αξιολογείται. Εάν οι οργανισμοί αξιολόγηση δεν ενδιαφέρονται για την επιβίωση των εταιριών ή των χωρών που αξιολογούν, αυτό θα επιφέρει ένα επικίνδυνο αγώνα δρόμου προ την υποβάθμιση και εδώ ακριβώς ε, τονίζεται το πόσο, σημαντική είναι, ε, πόσο σημαντικό είναι το μοντέλο του ότι ο εκδότης πληρώνει. Η ε, μεγάλη αμερικανική οίκη αξιολόγηση φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για την επιβίωση των χωρών ή των εταιριών που αξιολογούνται. Εμείς στη JCR είμαστε πολύ προσεκτικοί στις υποβαθμίσεις των εκδοτών σε περίπτωση που αυτό θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση και αποφεύγουμε πολύ προσεκτικά το απλώς να ακολουθούμε ή να επιταχύνουμε τις Τάσει τη αγορά. Δεύτερον, για να μην υπάρξει η τωρινή κατάσταση ολιγοπολίου που στρεβλώνει την αγορά, ε, υπάρχει ανάγκη ε, αυξημένου ανταγωνισμού στον κλάδο. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Από αυτή την άποψη, η Ιαπωνία νομίζω ότι μπορεί να παρουσιάσει ένα καλό παράδειγμα. Δύο Ιαπωνικοί οίκοι αξιολόγηση ε, ανταγωνίζονται με Αμερικανού γίγαντες και επιτυγχάνουν και έχουν εμπιστοσύνη στην αγορά. Όσον αφορά τα ομόλογα που εκδίδονται από ιαπωνικές εταιρείες στην ιαπωνική αγορά, περίπου 80% αυτών αξιολογούνται από ιαπωνικούς οίκους αξιολόγησης. Και πραγματικά χαιρετίζω την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία να δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί οίκοι αξιολόγησης. Οι οίκοι αξιολόγηση που ασχολούνται με την αξιολόγηση πιστοληπτική ικανότητα σε μια χώρα ή σε μια περιφέρεια θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το πολιτικό και το κοινωνικό περιβάλλον καθώς και την ε, ε, ε, πολιτική, τη φιλοσοφία της εταιρείας ή της χώρας. Για να υλοποιηθούν αυτές οι πρωτοβουλίες ε, η πορεία είναι πολύ δύσκολη και υπάρχουν πολλές προκλήσεις διότι το μέγεθος και η αναγνώριση της αγοράς είναι τα βασικά εμπόδια. Ηρωνικά, το πρόσφατα ενδυναμωθέν ρυθμιστικό πλαίσιο ως αποτέλεσμα των προβληματικών πρακτικών των Αμερικανών γιγάντων μπορεί να είναι το υψηλότερο, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους αλλά και για τους υφιστάμενους μικρούς οίκους αξιολόγησης. Το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να εμποδίζει την είσοδο νέων οίκων ούτε να αποθαρρύνει τη λειτουργία μικρών και μεσαίων οίκων αξιολόγησης. Στην Ευρώπη πιθανόν η του ανταγωνισμού μπορεί να απαιτεί πολιτική σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο για να δημιουργηθούν νέοι οίκοι αξιολόγηση και για να κατευθυνθούν οι δραστηριότητες προς, τις νέες, προς τους νέους με την υποστήριξη της εταιρείας ή της χώρας ή της περιφέρειας. Όσον αφορά το τωρινό υφιστάμενο ολιγοπόλιο, η υποχρεωτική εκπεριτροπής αξιολόγηση δεν θα ε, αυξήσει τον ανταγωνισμό. Αν υπάρξουν όμως ε, οίκοι που ετοιμάζονται να δραστηριοποιηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος να δοκιμάσουμε την εκπεριτροπής αξιολόγηση. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, θα πρέπει ε, να κάνουμε τα εξή δύο σχόλια. Κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και του κινδύνου του δημοσίου χρέους, το πιο σημαντικό είναι η πολιτική ε, και η αποφασιστικότητα των ε, πολιτικών και ηθινόντων, καθώς και η αντοχή του λαού ακριβώς αυτό παραμελείται από τους μεγάλους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης όσον αφορά το δημόσιο χρέος των χωρών της Ευρωζώνης. Το επόμενο σημείο είναι ότι παρότι ένας οίκος αξιολόγησης είναι ιδιωτικός, θα πρέπει να έχει και κάποια δημόσια στοιχεία και ε, ε, κατά αυτόν τον τρόπο να, υπά... και δημόσια υπευθυνότητα, ε, διότι η αξιολόγηση ασκεί κέρια επίπτωση στην αγορά και στην τύχη ενός έθνους και στην τύχη τόσων πολλών ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Τιερή Φιλίππονα, Γενικός Γραμματέας της Finance Watch. Πέντε λεπτά έχετε. Ευχαριστώ. Is it working? Yeah, sorry about that. Thank you very much. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μιλάω σήμερα ε, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μεταξύ των πολλών και διαφόρων ε, υποθεμάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα οποία βρίσκονται στη μέση διάταξή μας σήμερα, θα ήθελα εγώ να ασχοληθώ με το ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ε, την υπερβολική εμπιστοσύνη του συνολικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στις εξωτερικές αξιολογήσεις. Γνωρίζουμε τα λάθη λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. <clears throat> Γνωρίζουμε το τι συμβαίνει σήμερα. Κάθε φορά ε, ανακύπτει το θέμα των οίκων αξιολόγηση και κάθε φορά προσπαθούμε να το λύσουμε. πώ είναι δυνατόν όμω να αντιμετωπίσουμε αυτή ε, την υπερβολική εμπιστοσύνη που έχουμε στου οικού αξιολόγηση. Δύο τρόποι υπάρχουν. Πρώτον, μπορούμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την δυνατότητα λάθους που έχουν ε, οι οίκοι αξιολόγησης. Ε, και ε, μερικές αναφορές πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές αναφέρονται ήδη στην οδηγία και στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως μπορεί κανείς ε, να το συζητήσει, πάντως είναι μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση είναι να οργανωθεί το σύστημα με τρόπο ώστε όταν κάνει λάθος ένας οίκος αξιολόγησης, αυτό το λάθος δεν οδηγεί τελικά σε μία συνολική καταστροφή η πραγματικότητα του κόσμου είναι ότι όλοι κάνουμε λάθη, πάντα θα υπάρχουν λάθη, έστω και αν ε, κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να αποφύγουμε τα λάθη αυτά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα σύστημα όπου μία και μόνη γνώμη δεν θα έχει την δυνατότητα να ε, επηρεάσει τις αποφάσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουν διπλό ρόλο οι εταιρείε αξιολόγηση οι οίκοι αξιολόγηση. Είναι και δικαστές και ένορκοι. Ε, και αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί. Ε, Από την μία πλευρά, σαν δικαστές, ε, κάνουν ανάλυση και αυτό και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, οι fund managers μέχρι ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ε, δεν κάνουν δική τους αξιολόγηση αλλά ήδη μέσα στους εσωτερικούς τους κανονισμούς των funds, της διαχείρισης των funds έχουν ενστερνιστεί την αξιολόγηση των οίκων αξιολόγησης. Ε, ε, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η διαγράμματος αξιολόγηση ε, η οποία τελικά δεν έχει και καμία έννοια αυτός ο τρόπος έκφρασης της αξιολόγησης μπορεί να έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο λεγόμενο cliff effect, την επίπτωση κρυμνού και παρόμοια άλλα ζητήματα. Ας πούμε, εάν βλέπουμε ας πούμε την αξιολόγηση η οποία είναι από ε, investment grade πηγαίνει σε non-investment grade και τότε όλοι ε, σχεδόν υποχρεώνονται να ε, πουλήσουν. Με αυτόν τον τρόπο τελικά δίνεται τόσο μεγάλη πίεση στην αγορά που οι ψυχολογικές επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Όσον αφορά τον κανονισμό, ε, ε, στην ε, τροποποιημένη πρόταση της Κομισιόν υπάρχουν κάποια, του περασμένου Νοεμβρίου υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία όσον αφορά την έκφραση του τρόπου αξιολόγησης. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ο τρόπος αξιολόγησης των οίκων τον έχουν ενστερνιστεί όλες οι διαχειριστικές αρχές. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι fund managers θα πρέπει ε, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό γίνεται και στην ε, ε, οδηγία. Οι fund managers δεν θα, πρέπει όχι μόνο να μην έχουν αλλά να υποχρεωθούν να αφαιρέσουν οποιαδήποτε αναφορά σε εξωτερική βαθμολόγηση ή αξιολόγηση που περιέχεται στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, λειτουργίας τους. Ε, θα πρέπει η έκφραση της αξιολόγησης να μην γίνεται πλέον με γράμματα της αλφαβήτου αλλά να εκφράζεται μία γνωμοδότηση βάσει ενός ε, ε, γραπτού κειμένου με επιχειρηματολογία η οποία θα καταλήγει στο ενδεχόμενο χρεοκοπίας probability of default ε, γιατί αυτό χρειάζεται η αγορά. Ένα γραπτό κείμενο που λέει η γνώμη μου είναι ότι έτσι και έτσι και έτσι και ότι πιστεύω ότι ενδεχομένως βάσει των επιχειρημάτων μου υπάρχει πιθανότητα χρεοκοπίας. Τότε ε, ε, μπορούμε να έχουμε ένα καλό σύστημα και αυτό θα πρέπει να φαίνεται και στην ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και βεβαίως θα πρέπει να περιληφθεί η τυποποιημένη μεθοδολογία η οποία θα αφορά τον τρόπο αξιολόγησης. Η ΕΣΜΑ λοιπόν λαμβάνοντας... Ε, ε, και η ΕΣΜΑ θα πρέπει λαμβάνοντας σε τέσσερις ή πέντε ε, τέτοιες εκτιμήσεις να εκτιμά πλέον η ίδια βάση αυτών και λοιπόν παραμέτρων το ενδεχόμενο αθέτησης με τον τρόπο αυτό και οι οίκοι αξιολόγηση θα παίξουν ε, τον ρόλο τους, δηλαδή να κάνουν αξιολόγηση, αλλά δεν θα είναι και σε θέση να επηρεάσουν με τόσο μεγάλο βαθμό ε, το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει η κυρία Βαντόρν, η οποία είναι ε, υπεύθυνη για τις σχέσεις με τους οίκους αξιολόγησης στην Société Générale και εκπροσωπεί και την EBF. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία να εκφράσουμε τι απόψει τη Société Générale και τη Ομοσπονδία Τραπεζών ως αφορά τη CRA. Χαιρετίζουμε την πρόταση να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των οίκων πιστοληπτική αξιολόγηση και τη αύξηση του ανταγωνισμού. Θεωρεί ότι η ανακύκλωση, η κυκλική εξέταση, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να τύχει περαιτέρω εξέταση. Ο τραπεζικό τομέα είναι ο μεγαλύτερο χρήστη αυτών των αξιολογήσεων και ακόμα και των ε, ρυθμιστικών ε, ε, διατάξεων. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε σχέση με την έκδοση 1,5 εκατομμυρίων ομολόγων ετήσια, η αρχή της ανακύκλωσης έχει το θέμα των κινδύνων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας στο πλαίσιο αυτό. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη ότι είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πλαίσια και να έχουμε διαφορετικέ περιόδου για την εκδοσή ομολόγων. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι υπάρχουν ε, οι αναλογίε ε, και σε σχέση με την διαφορετική αξιολόγηση του ιδίου ομολόγου ετήσια θα δημιουργήσει ένα κίνδυνο να, να γίνουν μη ε, ελκυστικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα μακροπρόθεσμα επειδή οι επενδυτές έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, ε, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν τουλάχιστον ε, τρεις ε, αξιολογήσεις. Στη ΣΥΠΑ οι διαχειριστές απαιτούν αξιολογήσεις από τρεις διαφορετικές υπηρεσίες αξιολόγησης και δεδομένου ότι το ίμιση των ανώτερων 100 επιχειρήσεων στη παγκόσμια δεν έχουν την έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν περιορισμένη ελαστικότητα οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Γι' αυτό είναι σαφές για μας ε, ότι η ταχύτερη εφαρμογή αυτών των διατάξεων για την ανακύκλωση θα μπορούσε να θέσει εν κινδύνο τις ε, δυνατότητες των τραπεζών δεδομένων των πιέσεων που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά ωστόσο, οι ευρωπαϊκέ τράπεζε δεν έχουν καταλήξει όμω σε συνενετική άποψη όσον αφορά την πρόταση για την υποχρεωτική αυτή ε, κυκλική αξιολόγηση. Και επειδή αυτή η πρόταση είναι καινούργια σχετικά για μα, όσον αφορά το CRA, γι' αυτό ω Societe Générale θεωρούμε και επίση ε, και άλλε ευρωπαϊκέ τράπεζε θεωρούν ότι οι ε, προτάσει που θα δώσουν τη δυνατότητα τη κυκλικής αξιολόγηση θα πρέπει να εξεταστούν παρότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα επί πολλά έτη τώρα η σχέση, ο συσχετισμός μεταξύ τραπεζών και ε, οίκων αξιολόγησης ε, δεν έχει ε, ανάλογη και ισόρροπη σχέση. Έχουμε και τα θέματα των αγορών και των ρυθμιστών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και η αξιολόγηση είναι σημαντική πτυχή της καθημερινής δραστηριότητας των τραπεζών θα πρέπει να δούμε εδώ ότι υπάρχει και σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεγάλο τμήμα ή η η και εκδίδουν ε, γνωμοδοτήσεις ε, οι απόψεις και από τις ε, ΗΠΑ προστατεύονται από την πρώτη τροπολογία του συντάγματός τους. Ωστόσο στην καθημερινή μας πρακτική η συμπεριφορά τους και οι απαιτήσει τους δημιουργούν ένα πλαίσιο έντασης για τους ρυθμιστές. Θα πρέπει να δούμε ότι σημαντικά θέματα περιορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και υπάρχει σημαντική η πίεση την οποία υφίστανται. Εμείς ως Societe General θεωρούμε ότι η αποκάλυψη πληροφοριών θα πρέπει να ρυθμίζεται με αυστηρό πλαίσιο, ώστε όλοι να αντιμετωπίζουν το ίδιο πλαίσιο και όλοι να έχουν το ίδιο ε, μέγεθος πληροφοριών που θα τους διατίθεται αν αυτό ε, θεωρηθεί επιτρεπτό. Θα πρέπει επίσης σε σχέση με, τον, ε, με τη δημοσίευση εκθέσεων να ε, εμπεριέχονται τυποποιημένες πληροφορίες και να μπορούν να ρυθμίζονται οι οίκοι αξιολόγηση χωρίς ε, ε, αντιφατικές πληροφορίες, χωρίς ε, αντιφατικές και πρακτικές που δημιουργούν τριβέ και να υπάρχει έτσι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Εμεί ω Societe General θεωρούμε ότι οι μεθοδολογίε όχι μόνο θα πρέπει να εξετάζονται, θα πρέπει και να εναρμονίζονται ή τουλάχιστον να βασίζονται σε κάποιο είδου κοινό πλαίσιο. Μόνο τότε και μέσα σε ένα πλαίσιο ε, ρύθμισης ε, κοινή αξιολόγησης ε, θα έχει αξία η αρχή τη ε, κυκλική αξιολόγησης. Δεν είναι πεισμένε όλε οι τράπεζε ότι είναι η καλύτερη χρονική συγκυρία για να εξεταστεί μια τέτοια πρόταση και θα πρέπει να ληφθεί επαρκή πρόληψη και προστασία των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ωστόσο, η Ευρώπη πάντα μάθαινε μέσα από κρίσει. Εμεί ω Societe Generale είμαστε πεισμένοι ότι προτού εισαχθεί η υποχρεωτική αρχή τη κυκλική αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο στοιχείων και μεθοδολογιών για του οίκου αξιολόγηση που θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Είναι μια ευκαιρία η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο, να μειωθούν οι μη ισόρροπες σχέσει μεταξύ των υπηρεσιών, των εκδοτών και να διασφαλιστεί ο ρόλο ε, των Ευρωπαϊκών Τραπεζών στην οικονομία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φαντόρ. Τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος επαϊών πραγματογνώμων. Έχετε πέντε λεπτά και εσείς στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία που δίνετε να παρέμβω σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Θα ήθελα να παρουσιάσω κάποια στοιχεία τα οποία δεν καλύφθηκαν από ακόμη. Πρώτα, θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω όσον αφορά τα προβλήματα σε σχέση με την αξιολόγηση που ξεκινούν με τη σύγκρουση συμφερόντων ιδιαίτερα όσον αφορά την κάλυψη των ε, εξόδων ε, από τους ε, εκδότες και τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό. Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι δημιουργεί μια μονοπωλιακή θέση στην αγορά, όπου οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης ελέγχουν ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, πράγμα το οποίο δεν δίνει κανένα κίνητρο για ανταγωνισμό και προσαρμογή των ε, αξιολογήσεων. Και τρίτον, ε, οι λόγοι που προαναφέρθηκαν πριν ε, ως αρνητικά στοιχεία. Ανακεφαλαιώνοντας, θα θέλαμε να πούμε ότι η σύγκρουση συμφερόντων, ιδιαίτερα η σύγκρουση συμφερόντων που θα πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με την κυκλική αξιολόγηση, δεν νομίζουμε ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί. Θα υπήρχε τεμαχισμό τεμαχισμός ε, της αγοράς ε, και θα είχαμε σε σχέση με τις επιστροφές ένα επίπεδο κερδοφορίας το οποίο δεν υπάρχει και σε καμία άλλη υπηρεσία ε, παροχής υπηρεσιών. Βλέπουμε ότι θα ε, πρέπει να ανταμυφθούν όσοι συμμετέχουν στην αγορά σε σχέση με τα ε, προτερήματά τους όσον αφορά προτερήματα τιμών ή προσφοράς. Θα πρέπει να υπάρχει ωστόσο ένα ισοδίκαιο πλαίσιο ε, στην αγορά όπου οι ίδιοι επενδυτές θα επιλέγουν το τι θα επιλέγεται. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει μεγαλύτερη ένταξη της έννοιας ε, του ο επενδυτής ε, πληρώνει, ε, ο επενδυτής καλύπτει εντός εισαγωγικών ώστε να υπάρχει ένα πιο ισοδίκαιο πλαίσιο. Η ανακύκλωση αυτή, η, κυκλική αξιολόγηση δεν θα πρέπει να μας κάνει να αγνοήσουμε αυτές τις ελλείψεις αυτής της πρότασης όσον αφορά μια πολιτική που θα στοχεύει στην οικονομία της αγοράς. Το επίπεδο της, των κινδύνων των προϊόντων δεν μπορεί να αρθεί ή να αντιμετωπιστεί λέγοντα λέγοντας ότι οι αξιολογήσεις ε, μπορεί απλά και μόνο να ε, συνεπάγονται μια γνωμοδότηση. Η μείωση των κινδύνων είναι πολύ θετική πτυχή. Καλωσορίζουμε αυτή την ε, πρόταση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή σχέση μεταξύ οίκων αξιολόγηση και επενδυτών. Διότι οι επενδυτέ είναι εκείνοι που θα χάσουν χρήματα αν η αξιολόγηση δεν είναι σωστή και αν παραπλανήθηκαν από κάποια αξιολόγηση. Και όχι ότι μια πολύ καλή αξιολόγηση δεν μπορεί ε, να οδηγήσει σε κάποια αθέτηση, διότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός κίνδυνος. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει σωστή αναλογία μεταξύ ποιότητας και ε, προσπάθειας ε, ή επένδυσης που έχει γίνει. Το τρίτο που πρέπει να, ρωτήσουμε, να ζητήσουμε είναι σε σχέση με τους ρυθμιστές που θα πρέπει να εγκρίνουν μεθοδολογικά τις προσεγγίσεις αυτές. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΣΜΑ, γιατί θεωρούμε ότι θα ε, υπάρχει δυνατότητα για την ε, αύξηση του ανταγωνισμού και θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια ε, ενιαία διαμόρφωση των αξιολογήσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και την δυνατότητα αντιμετώπισης της παραπλάνησης. Διότι αν υπάρχει κίνδυνος επικέντρωσης θα μπορούσε να υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος στρέβλωσης στη συνέχεια. Αυτό όσον αφορά την φούσκα στην αμερικανική αγορά, όπου η μεθοδολογία οδήγησε στο να υπάρχει παραπλάνηση και τέτοιου είδους κίνδυνοι ε, συμπίκνωση ε, επικέντρωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Μακροπρόθεσμα τα αριθμιστικά ε, σώματα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλιστούν, να καλύψουν αυτή την πτυχή και γι' αυτό θεωρούμε ότι οι, Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας και ρύθμισης θα πρέπει να δράσουν. Έχουμε αναπτύξει μια πρόταση πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό σε σχέση με την αγορά. Μία πρόταση σε σχέση με την οικονομία της αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία αγορά για τις αξιολογήσεις όπου οι εκδότες θα δημοσιεύουν τις ε, σημαντικές για τις αξιολογήσεις ε, πληροφορίες θεωρούμε ότι τα απόρριτα στοιχεία δεν βελτιώνουν ε, την αξιολόγηση, δεν υπάρχει κάποια απόλυτη ένδειξη γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και καλωσορίζουμε αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Δεν πρέπει να υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος ούτε κανενός. Θα πρέπει όλοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία και να χρησιμοποιούν και την αξιολόγηση ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε σχέση με τις, τους οίκους αξιολόγησης όσον αφορά το συσχετισμό και των επενδυτών σε σχέση με τα όσα προσφέρονται. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω ε, δεν θεωρούμε ότι το θέμα της κρατικής υπερχρέωσης είναι το ε, κυριότερο θέμα όταν ε, έχουμε την αντιμετώπιση της δράσης της των οίκων αξιολόγησης στις αγορές. Με τις υποβαθμίσεις αντανακλώνται κίνδυνοι σε σχέση με τους όσους συμμετέχουν στις αγορές και μια αναθεώρηση της αγοράς δεν θα έπρεπε μόνο να οδηγήσει σε καλύτερες αξιολογήσεις αλλά και σε δημιουργία μεγαλύτερης διαφάνειας. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κράτ. Τώρα θα λάβει τον λόγο τελευταία η κυρία Σούσαν Λόνι, ανώτερη σύμβουλος για ευρωπαϊκές ε, ε, υποθέσεις της Feed Ratings. Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ. Mr. Vice Chair distinguished... Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείτε να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι η οίκη αξιολόγηση ε, είναι το επίκεντρο της προσοχής των ρυθμιστικών αρχών. Καταλαβαίνουμε τις ελλείψεις των, ε, των αξιολογήσεων ε, των, της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ και την τυπλοποίηση αυτών των αξιών στη συνέχεια. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι είναι σημαντική και αξιολόγηση για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο προσκήνιο. Γι' αυτό έχουμε κάνει και πολλές αλλαγές στη μεθοδολογία μας και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και σχετικές προτάσεις. Καταλήτη για τη σημερινή ακρόαση είναι η πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής να τροποποιηθεί ο κανονισμό CRA. Η Fitch συμφωνεί με τους στόχους της πρότασης ε, σε γενικές γραμμές να αυξηθεί ο ανταγωνισμό και η διαφάνεια στην αγορά αξιολόγηση. Πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Fitch έχει συνεισφέρει και στα δύο αυτά θέματα. Τι τελευταίε δύο δεκαετίε εμεί είμαστε η μοναδική εταιρεία που μπορεί να ανταγωνιστεί τη Moody's και την SP, παρότι είμαστε ακόμη πολύ μικρότεροι. Επίση, υποστηρίζουμε τι προσπάθειε να μην υπάρχει μια μηχανιστική αντιμετώπιση στο πώ εξατόμεθα από τι αξιολογήσει. Πιστεύω, ωστόσο, ότι πολλέ από τι πρόσφατε προτάσει τη Επιτροπή θα καταλήξουν σε λιγότερο ανταγωνισμό, λιγότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις αξιολογήσεις. Όπως έχει συνταχθεί τώρα η πρόταση της Επιτροπής, το δυναμικό για συνέπειες από αυτές τις βιαστικές προτάσεις ε, είναι μάλλον αρνητικό. Επίσης υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι προτάσεις αυτές να αυξήσουν την αναταραχή που υπάρχει στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Γι' αυτό θα ασχοληθώ μόνο με ένα θέμα, την εκπεριτροπής αξιολόγηση. Θα ήθελα όμω να δείτε το πλήρε κείμενό μου για να συζητήσουμε τα σχετικά θέματα. Στρέφομαι τώρα στι προτάσει για την εκπεριτροπή αξιολόγηση. Η Fitch πάντοτε ήταν υπέρ του ανταγωνισμού και πάντοτε καταπολεμούσαμε το διοπόλιο τη Moody's και τη S&P. Τα τελευταία 20 χρόνια αυτό κάναμε και μπορέσαμε να αυξήσουμε το μείδιο αγορά μα κατά 17% σε σχέση με 37% τη Moody's και 43% τη Standard Poor's. Θέλουμε να σπάσει αυτό το δύο πόλιο. Ανησυχούμε όμω ότι κάποιε από τι προτάσει ε, μπορεί να ενισχύσουν περισσότερο τη Moody's και την S&P ιδίω. Όσον αφορά τον προτινόμενο κανόνα ότι ένα οίκο αξιολόγηση μπορεί να αξιολογεί μόνο 10 εκδόσει ενό εκδότου πριν από την ε, εκπεριτροπή ε, εναλλαγή, με ελάχιστο χρόνο ενό έτου. Παρακαλούμε, αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο σιγά, γιατί δεν σα καταλαβαίνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Να ξεκινήσω από κάπου αλλού ή να συνεχίσω. Θέλετε να, ξα... να επανελάβω κάποια από αυτά που είπα. Λοιπόν, αυτό ακριβώ είναι το θέμα για τον προτινόμενο κανόνα ότι ένα οίκο αξιολόγηση μπορεί να αξιολογεί 10 εκδόσει ενό εκδότου πριν πρέπει να υπάρξει αναλλαγή με ελάχιστο χρόνο ένα έτο πριν την αναλλαγή. Ωστόσο, ένα δεύτερο οίκο για τον ίδιο εκδότη μπορεί να συνεχίσει να αξιολογεί αυτόν τον εκδότη και του τίτλου για 6 χρόνια. Δεδομένης τη δύναμη τη αγορά ε, τη Moody's και τη ε, S&P, πιστεύουμε ότι οι εκδότε θα πρέπει να υποχρεώνονται ε, να ζητούν αξιολόγηση από έναν από του δύο δύο οίκου αυτού, οποιαδήποτε στιγμή και ένα από του δύο αυτού μεγάλου θα πρέπει να είναι ο οίκο αξιολόγηση για τα έξι χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 τράπεζε αναγκάστηκαν να αλλάξουν οίκο αξιολόγηση μετά από ένα χρόνο σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα των 10 ε, ε, εκδόσεων. Το ίδιο ισχύει για 25 μεγάλε εταιρείε τη Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η France Telecom, η Deutsche Bahn, η Volkswagen, η EDF, BP και η Volvo για να πληρούνται οι απαιτήσει αυτών των διατάξεων για την περιτροπή, οι εκδότε ε, μάλλον θα χρησιμοποιήσουν κατά μέγιστο δύο οίκου αξιολόγηση κάθε στιγμή. Αυτό είναι αντίθετο με την εκπεφρασμένη επιθυμία των ε, επενδυτών και ρυθμιστικών αρχών να υπάρχουν περισσότερε απόψει στην αγορά εργασία και εκτιμούμε ότι το 55% των ε, τραπεζών εκδοτών στη Δυτική Ευρώπη έχουν τρει ή περισσότερε αξιολογήσει σε κάθε μία. Και αυτό το κάνουν διότι οι επενδυτέ που αγοράζουν τα ομόλογά του αξιολογούν ένα μεγάλο φάσμα γνωμοδοτήσεων για την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότου. Κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι επενδυτέ να αξιολογήσουν τον πιστοτικό κίνδυνο των ομολόγων, αυξάνεται η ζήτηση και μειώνεται το επιτόκιο που καταβάλει ο εκδότη. Το αποτέλεσμα μια πρόσφατη μελέτη 3.000 τίτλους στις Ηνωμένες Πολιτείες αξίας 1,63 εκατομμυρίου δολαρίων ήταν ότι οι τίτλοι με τρεις αξιολογήσεις ε, είναι περίπου 40 BPS ε, καλύτερα από ότι τίτλοι με δύο αξιολογήσεις μόνο. Η πραγματικότητα της αγοράς είναι ότι υπάρχουν ε, ε, τρεις ε, οίκοι αξιολόγηση σε παγκόσμια βάση, η Fitch, η Moody's και η S&P. Χρειάστηκαν δύο δεκαετίες ε, και επενδύσεις πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να μπορέσει η Fitch να ανταγωνιστεί με τη Moody's και την S&P σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης ανταγωνίζονται για χρηματοδότηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Volkswagen, παραδείγματο χάρη, αν θα έπρεπε να έχει μόνο μία αξιολόγηση για ολόκληρο τον κόσμο, θα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση γιατί θα προσπαθούσε να αντλήσει κεφάλαια στι ΗΠΑ και αλλού εκτό τη Ευρώπη. Αυτό τονίζει επίση και το ότι σύμφωνα με τι προτάσει αυτέ, οι οίκοι αξιολόγηση μπορεί να επιλεγούν για λόγου διαφορετικού και όχι για την ποιότητα των αξιολογήσεών του. Παραδείγματο χάρη δεδομένου του μικρού αριθμού οίκων αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του μεγάλου χρονικού διαστήματο που χρειάζεται για να αποκτήσει κανεί την εμπειρία, οι εκδότε μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα οίκο αξιολόγηση, μόνο και μόνο διότι όλοι οι άλλοι είναι σε περίοδο που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι μπορεί να χρησιμοποιήσουν δεύτερο οίκο αξιολόγηση, δίπλα στου δύο μεγάλου, μόνο και μόνο διότι οι αξιολογήσει του δεύτερου οίκου είναι υψηλότεροι από ό,τι τη Moody's ή τη S&P. Δεδομένων αυτών των συνεπειών που δεν είναι αυτέ οι οποίε θα επιθυμούσε η Επιτροπή, δεν ξέρουμε αν ο πραγματικό σκοπό των, διατάξεων για την σε αξιολόγηση δεν είναι να ε, ενταθεί ο ανταγωνισμό, αλλά να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συγκεκριμένων οίκων αξιολόγηση, ε, όπου ο συνδρομητής θα πληρώνει και όχι ο εκδότη θα πληρώνει ε, δεδομένου του πού θα εφαρμόζονται οι κανόνες για του οίκου αξιολόγηση. κάτι το οποίο είναι μια ε, ανεπιθύμητη συνέπεια. Πολλοί από αυτούς που απάντησαν στη διαβούλευση τη Επιτροπής είπαν ότι συγκρούσει συμφερόντων θα υπάρχουν σε όλα τα μοντέλα. Η Fitch πιστεύει, χωρί μικρόφωνο η ομιλήτρια. Η Fitch πιστεύει ότι η αγορά θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα μοντέλα, δεδομένου ότι συγκρούσει συμφερόντων θα πρέπει να εντοπίζονται και στο μέτρο του δυνατού να εξαλείφονται. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται το μοντέλο του ότι ο εκδότης πληρώνει, πιστεύουμε ότι είναι καλώς κατανοητές οι συγκρούσεις συμφερόντων και δημοσιοποιούνται. Το ότι έχουμε υποβαθμίσει πρόσφατα 8 από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες είναι ένα αντεπιχείρημα στο ότι οι αξιολογήσεις μας κινούνται από το ότι μας πληρώνουν οι εκδότες. Με βάση την εμπειρία μας, οι υπηρεσίες που, πληρών, που παρέχουν οι και αξιολόγηση που πληρώνονται από τον εκδότη δεν μπορούν να παρασχεθούν από ένα μοντέλο που πληρώνει ο επενδυτής. Τώρα θα αρχίσει ο γύρος ε, παρεμβάσεων ξεκινώντας ε, από τον εισηγητή και από τους δύο εισηγητές όσον αφορά τις υπηρεσίες αξιολόγησης. Ε, θα σας ευχαριστούσα αν λέγατε προς ποιον στοχεύει η ερώτησή σας ή η παρέμβασή σας. Ο κύριος Ντομινίτσι πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Ντομινίτσι. Στο τέλος, εντάξει. Κύριος Γκοζές, σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΑ και συντονιστής ε, του ΕΛΚΟ. Κύριος Γκοζές, παρακαλώ, έχει τον... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρουν, όπως ξέρετε, η, η, η, μου και η εισηγητής των δύο πρώτων εκθέσεων. Θέλω να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι είναι πιο έξυπνο να δίνει κανείς συγκεκριμένα μηνύματα και όχι σύντομα ε, και όχι γρήγορα παρά επί 7 λεπτά να μας κατακλίζουν σε γλώσσες περίεργες ε, και που οι διερμηνείς προσπαθούν ε, και του συμπονώ για το έργο τους προσπαθούν να μεταφράσουν. Εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι, ότι υπάρχουν πολλές κάμερες και γιατί αυτό, μα γιατί οίκη αξιολόγηση ε, που δεν ήξεραν ούτε καν ότι υπάρχουν οι πολίτε τη Ευρώπη πριν από μερικού μήνε. Τώρα είναι στα χείλη όλων. Πρώτε σελίδε τη εφημερίδε, όλοι μα λένε για θέτηση όρων, όλοι μα μιλάνε για δημόσιο χρέο. Δεν θέλω να υπεραμεινθώ των οίκων αξιολόγηση, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μα. Θεωρώ ότι τα δύο κείμενα τα οποία έχουν εγκριθεί είναι ήδη ε, κείμενα καλά τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Η εκπρόσωπος της ΕΣΜΑ γνωρίζει πολύ καλά πόσο αγωνίστηκα έτσι ώστε οι τρεις κύριοι ήξοι αξιολόγησης να αποκτήσουν πιστοποίηση ε, ενώ έχουν υποβάλει, ε, τα, είχαν υποβάλει τους φακέλους τους τον Νοέμβριο του 10 πιστοποιήθηκαν τελικά το Δεκέμβριο του 11. Βεβαίως δεν ήταν ευθύνη της ΕΣΜΑ αλλά του, της εποπτικής, της ρυθμιστικής αρχής όμως αυτό καταδεικνύει τη δυσκολία του πράγματος, πόσο δύσκολο δηλαδή είναι να προχωρήσει ε, η νομοθεσία για ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε στρώματα επιστρωμάτων κανόνων και κανονισμών που δεν θα ε, υλοποιηθούν ποτέ. Ε, εγώ που έχω μάθει να βασίζομαι στα οικονομικά στους μαθηματικούς κανόνες ε, πραγματικά βρίσκω παράλογη όλη τη φιλολογία και τη συζήτηση που γίνεται για όλα αυτά τα θέματα. Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ε, να επισφραγίσει, να εγγυηθεί και να δώσει μία βαθμολόγηση στους οίκους αξιολόγησης έτσι ώστε να βοηθηθεί η αγορά και οι επενδυτές. Εμείς φταίμε εάν οι οικοί κατέλαβαν τόσο μεγάλη θέση στις ε, ε, χώρες μας. Πρώτο, το, το ίδιο το, σύστημα ε, των ε, funds και οι ίδιες οι τράπεζες, όπως υπόθηκε προηγουμένες, προηγουμένως, έχουν ενσωματώσει τους κανόνες των οίκων αξιολόγησης ε, στα, συστήματά τους. Και από την άλλη μεριά, ενώ λέγαμε ότι η οίκοι αξιολόγηση είναι σημαντική όταν χάσαμε το τριπλό α, είπαμε εντάξει δεν έγινε και τίποτα, επομένως μπερδεύονται οι πολίτες μας. Ε, είναι γεγονός ότι ε, σε σχέση με το δημόσιο χρέος κάθε ε, υποβάθμιση υποτίθεται ότι θα πρέπει να αυξάνει το επιτόκιο δανεισμού. Είδαμε όμως ότι και στη Γαλλία και σε άλλες περιπτώσεις χάνει η Γαλλία το, το, το τριπλό α αλλά δανείζεται με καλύτερες συνθήκες. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι πλέον η αγορά έχει αποσυνδεθεί. Εν πάση περιπτώσει το σημαντικό είναι ε, ότι όλοι λένε ότι ο ανταγωνισμός ε, είναι ο κυρίαρχος ε, στόχος και επομένως για να έχουμε καλύτερες συνθήκες θα έχουμε μεγαλύτερη, μεγαλύτερο ανταγωνισμό μέσω της περιτροπής. Ναι, αλλά λυπούμε το θέμα της περιτροπής δεν είναι τόσο εύκολο. Είδαμε, ακούσαμε και την εκπρόσωπο της Φίτς. Η Φίτς κουράστηκε πάρα πολύ και χρειάστηκε πολύ χρόνο ε, για να μπορέσει να καταλάβει τη θέση που καταλαμβάνει στην αγορά, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τους άλλους δύο, το ακούσαμε προηγουμένως. Επομένως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι προτάσεις περιτροπής ε, στην ουσία θα ενδυναμώσουν έτσι περαιτέρω τη θέση το, της διαρχίας των δύο οίκων αξιολόγησης και θα αποκλείσει την εισαγωγή στην αγορά άλλων οίκων. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν μια χώρα χρειάζεται αξιολόγηση, δεν επιλέγει μια μέσου μεγέθους, ένα μέσου μεγέθους εθνικό οίκο αξιολόγηση, επιλέγει έναν από τους ε, μεγάλους ε, οίκους ε, αξιολόγησης. Ε, και όπως είπε και ο Ζωαμπιέρ Ζουγέ που λυπάμαι που δεν είναι στην ΕΣΜΑ θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε ε, να ζούμε χωρίς ε, τις, να κάνουμε αποτοξίνωση κατά κάποιο τρόπο από τους οίκου αξιολόγηση. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που δεν θα είναι ακριβώς ένα θερμόμετρο το οποίο θα μεγαλώνει από μόνο του, θα τροφοδοτεί από μόνο του τον πυρετό και όταν ας πούμε ανακοινώνει κάποια αθέτηση οι επιπτώσεις ε, για την ε, ε, αφορόμενη χώρα να είναι δραματικές. Το ερώτημα το οποίο τίθεται σήμερα για τον τρίτο κανονισμό το είχαμε θέσει και πριν από πολλά χρόνια και το 1999 και το, το 2010 και το δεύτερο κανονισμό και δεν είχαμε βρει καλό τρόπο αντιμετώπισης. Το σχήμα του ε, issuer payer είναι ένα πρόβλημα και ο Ιάπωνας παρεμβαίνω σήμερα το πρωί το είπε. Ε, όταν πληρώνει ο επενδυτής θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι να μην ξεκινήσουμε νομοθεσία η οποία δεν θα έχει καμία πρακτική επίπτωση και που μονάχα θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αναταραχή. Ε, αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η φυστάμενη νομοθεσία. Όσον αφορά το ρόλο της ΕΣΜΑ, η ΕΣΜΑ οπωσδήποτε θα υποπτεύσει τις πιστοποιημένες υφιστάμενες εταιρείε αξιολόγησης έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι λειτουργούν αυτή η εποπτεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να ζητάμε όμως και να περιμένουμε από την ΕΣΜΑ πέρα ε, και παραπάνω από αυτά που μπορεί να κάνει μια ρυθμιστική αρχή. Δεν μπορεί να ε, ε, είναι υπεύθυνη η ΕΣΜΑ για τον τρόπο εργασίας ή για την ποιότητα του αποτελέσματος. Η ΕΣΜΑ πρέπει να εποπτεύει έτσι ώστε να ξέρει ότι λειτουργούν βάσει των κανόνων οι οίκοι αυτής και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να σταματήσει είναι μια αδιάφανη λειτουργία των ε, οίκων αυτών που δίνουν περίεργες αξιολογήσεις στην αγορά. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, υπάρχουν πολλά στοιχεία υπολογισμού, το είπε ο Ιάπωνας παρεμβαίνουν τα κράτη ε, είναι γεγονός ότι ε, ε, μέσω, της, μέσω των δημοσιονομικών αρχών και μέσω της, των φόρων τα κράτη μπορούν να ανανεώσουν τα κεφάλαιά τους ενώ οι εταιρείε και οι επιχειρήσεις θα βρεθούν χωρίς καθόλου κεφάλαια και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριο Σουβάρτ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πρέπει νομίζω το συνολικό αυτό θέμα με ψυχραιμία να το αντιμετωπίσουμε, χωρίς υπερβολική συναισθηματική φόρτιση. Το θέμα των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης τις τελευταίες εβδομάδες πιστεύω εγώ ότι για όλη αυτή τη συζήτηση πήρε μια τέτοια μορφή και ένταση που μάλλον μας παρακολεί στην αναζήτηση μιας σωστής λύσης από ό,τι θα μας ευνοούσε. Γίνεται λόγος για μια θεωρία συνωμοσία ήδη Κάποιοι δημοσιογράφοι πάνε και τόσο μακριά και λένε ότι επειδή οι Αμερικανοί μέσω των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης προσπαθούν να παρέμουν λέει, στην ευρωπαϊκή οικονομία με αυτόν τον τρόπο και εδώ θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και πάλι και να είμαστε ψύχρεμοι και νυφάλιοι. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει καλές προθέσεις, όμως σε πολλά επιμέρους ε, σημεία αγνοεί το πρόβλημα και ο ίδιος Ζαν Πολ Γκοζές το προανέφερε. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι βιώσιμες προτάσεις ε, και εφικτές προτάσεις και πού λείπουν και προτάσεις για την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι δεδομένο ότι οι οίκοι αξιολόγηση έχουν δυσανάλογη σημασία σε σχέση με τα όσα λένε οι ίδιοι οι οίκοι αυτοί για τον εαυτό τους. Όταν λένε ότι εκδίδουν μια γνωμοδότηση, αυτό είναι εφημισμός. Ε, έχει τεράστιες επιπτώσεις αυτή η εισαγωγικά γνωμοδότηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την κρατική υπεχρέωση κάποιων χωρών και ομόλογα αυτών των χωρών που εκδίδονται. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ να μεριμνήσουμε για τη σωστή θέση των πραγμάτων. Η πρώτη παρατήρηση που ήδη από κάποιους προαναφέρθηκε είναι το ότι έχουμε υπερβολικά μεγάλη, δυσανάλογη εξάρτηση από αυτούς τους οίκους ε, ε, αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κρατικά ομόλογα. Και δεν μπορούμε αυτό να το κατανοήσουμε. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται. Διότι όλα όσα χρειάζεται για να αξιολογήσει κανείς την ποιότητα τέτοιων προϊόντων μιας χώρας είναι από πολλές πηγές ε, μηνιαία όλα διαθέσιμα. Όσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όλα αυτά τα όργανα δημοσιεύουν μηνιαία πληθώρα πληροφοριών που είναι αναγκαίες ε, για την αξιολόγηση αυτών των χωρών και πτυχών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιδοτικά ταμεία ή επενδυτικά κεφάλαια για ποιο λόγο αυτά θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε μια αξιολόγηση ενός των οίκων αξιολόγησης και να μην λαμβάνουν τις αποφάσεις ιδία ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν εμεί οι ίδιοι να μεριμνήσουμε για αυτήν την αλλαγή. Εμεί οι νομοθέτε. Και εμεί όμω οι ίδιοι μπορούμε με νομοθετικέ προτάσει και τροποποιήσει να μεριμνήσουμε να απελευθερωθούμε από την ε, ας το πω έτσι, δεσμευτική πρόταση μιας ή αξιολόγηση ενός οίκου αξιολόγησης. Πρέπει να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και πρέπει να γίνει άμεσα η ευθύνη για την αξιολόγηση, δηλαδή η ευθύνη για το προϊόν είναι κάτι το οποίο συμμερίζομαι, διότι έχω και την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία που συνέταξα. Πρέπει όμως εδώ ωστόσο να δούμε και τους κινδύνους που ελοχεύουν. Αυτή τη στιγμή σε 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 27 διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο αστικού κώδικα, αστικής νομοθεσίας για αυτά τα θέματα στην Ευρώπη. 27 διαφορετικά συστήματα έχουμε. Αν θέλουμε να εισαχθεί η ρήτρα για την ευθύνη υπευθυνότητα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε 27 διαφορετικά τέτοια καθεστώτα για αυτή την ευθύνη, την αστική ευθύνη. Και έτσι ανοίγουμε πόρτα και παράθυρο ώστε να υπάρχει εδώ legal arbitrage. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε φυσικά. Και γι' αυτό καλείται εδώ ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει και να διασφαλίσει ότι αυτό ο κίνδυνο θα αντιμετωπιστεί και δεν θα υπάρχει πλέον για μα. Η ΕΣΜΑ έχει ένα σημαντικό ρόλο. Όμω δεν πρέπει να ζητάμε υπερβολικά πράγματα από την ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ μπορεί, όπω πιστεύω εγώ, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για τι μεθοδολογίε των οίκων πιστοληπτική αξιολόγηση ώστε για την ποιότητα και την ε, αποτελεσματικότητα των αξιολογήσεων είναι υπεύθυνοι. Είναι πολύ περίπλοκες τεχνικές διεργασίες. Για να τις κατανοήσει κανείς απαιτείται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ενασχόληση. Και πραγματική αντιμετώπιση σε βάθο όλων αυτών. Αυτά δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα η ΕΣΜΑ. Αυτό που θα μπορούσε να προσπαθήσει η ΕΣΜΑ και ίσω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να έχει ευθύνη είναι να μεριμνήσει ώστε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, των οίκων αξιολόγηση, να είναι καλύτερα συγκρίσιμα στο μέλλον από ό,τι σήμερα. Περισσότερα δεν μπορούμε να αναμένουμε ή να απαιτούμε. Η αρχή της κυκλικής ε, ε, αξιολόγηση αναφέρθηκε από τον Ζαν Πολ και από, εκπροσώπους, ε, από τον εκπρόσωπο της ε, Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Συμμερίζομαι την επιφύλαξη ότι με τέτοιου είδους ε, ανακύκλωση ενισχύουμε το διπολικό σύστημα. Θέλουμε όμως να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και γι' αυτό θλίβομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της δεν συμπεριέλαβε τη δική μας ιδέα και πρόταση. Τουλάχιστον να γίνει προσπάθεια και να αναλυφθεί ε, το διάφημα, μια ευρωπαϊκή, ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης υπομορφήν ιδρύματος να μπορέσει να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει. Καλό θα ήταν αν παράλληλα με τους τρεις μεγάλους οίκους θα είχαμε εμείς ως Ευρώπη μια δική μας ξεχωριστή τέτοια ε, οργάνωση ως ε, οίκο αξιολόγησης. Εν τω μεταξύ πάνω από 90% της αγοράς παγκόσμια ε, αξιολογείται από αυτούς τους τρεις οίκους. Και αυτό είναι ίσως μάλιστα θα έλεγα μια μονοπωλιακή θέση για αυτές. Ε, και με πάνω από 40% όσον αφορά τις ε, επιστροφές μετά την ε, χρεοκοπία της, ε, του οίκου Lehman Brothers και αυτά τα οποία συνέβαιναν και πιο πριν δείχνουν ότι υπάρχει μονοπωλιακή θέση από πλευρά τους. Χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Ασία, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, παντού. Και δεν πρέπει να υπάρχει πρόημα κάποια δράση, αλλά να κάνουμε κάτι αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα. Με ενοχλεί ένα πράγμα και το οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι η χρονική συγκυρία, το timing της έκδοσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης τώρα. Τι διαπιστώνουμε. Μπορεί ίσως να ήταν μια τυπική σύμπτωση, αλλά ε, φταίχτης είναι εκείνος ο οποίος ε, ενδίδει στον πειρασμό και σκέφτεται πιο πονηρά. Ίσως θα μπορούσε σε σχέση με την Σύνοδο Εκοφήν, ίσως σε σχέση και με την έκδοση νέων τέτοιων ομολόγων, να βλέπουμε ότι αλλάζουν τέτοιες αξιολογήσεις. Κάποιες λίγες μέρες ε, ή και λίγο πιο πριν συμβαίνουν τέτοιες αλλαγές αξιολόγησης. Τι συμβαίνει εδώ. Στις περισσότερε περιπτώσεις η αλλαγή αξιολόγησης έρχεται καθυστερημένα. Ωστόσο όμως ξέρει κανείς ότι το παιδί έπεσε στο πηγάδι και υπάρχει εδώ ε, κίνδυνος και μετά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή αξιολόγησης και σε σχέση και με πριν από δύο εβδομάδες πότε έγινε αυτό αυτά έγιναν όταν πλέον ήταν σαφές ότι θα ε, συνέβαινε κάτι τέτοιο ως προοπτική. Πώς μπορούμε λοιπόν να μεριμνήσουμε η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης να ανταποκρίνεται περισσότερο στην, πραγματικότητα και όχι να υπάρχει κάποια ε, πολιτική σε εισαγωγικά πρόθεση. Επαρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, ε, βλέπω τον σκιώδη εισηγητή της ΣΕΚ. Δεν ξέρω, κύριο Στρέτσεκ θέλει να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, εσείς θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ πολύ δεν είμαι ο Γιώργης εισηγητής της ECR, δεν είμαι πραγματογνώμων σε σχέση με τα θέματα εικοναξιολόγησης. Ωστόσο με μεγάλη προσοχή άκουσα και παρακολούθησα αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν και θα ήθελα και εγώ να κάνω δυο, να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, από πλευράς μου. Συμφωνώ με τον κύριο Κλίντς πρέπει να πω ότι στην σημερινή κατάσταση και συγκυρία αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια νυφάλια, μια ψύχρεμη, μια όρημη, ήρεμη συζήτηση που θα επικεντρώνεται στα θέματα ουσίας. Και θα έπρεπε να στοχεύουμε με ψύχρεμο τρόπο να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, η έκβαση η τελική. Ίσως αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της ε, ενίσχυσης, ενδυνάμωσης ε, ανταγωνισμού μεταξύ των CRAs. Μου φαίνεται ότι αυτούς τους τελευταίους μήνες οι ε, CRA από πλευρά τους δημοσίευαν πληροφορίες σε σχέση με τις εταιρείες, ε, κοινωνίες μας ε, που ε, ήταν ίσως ανησυχητικά τα στοιχεία αυτά για πολλού. και είναι πράγματα τα οποία πολλέ φορέ πολιτικοί εκπρόσωποι τη πολιτική ζωή δεν θέλουν και δεν του αρέσει να ακούν. Υπάρχει εδώ η τάση να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για να ενθαρρύνονται οι υπηρεσίε αυτές μελλοντικά να δημοσιεύουν τέτοιου είδου στοιχεία όπω αυτά τα οποία θα ήθελαν να λαμβάνουν υπόψη και να ακούουν οι πολιτικοί. Ωστόσο, πρέπει εδώ να δούμε ότι υπάρχει επικέντρωση γύρω από το θέμα του ανταγωνισμού. Ανταγωνισμού μεταξύ οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ακούγοντας ε, τους διάφορους εισηγητές, ε, αναγνωρίζω ότι και οι ίδιοι αυτοί από πλευρά τους ε, οι εισηγητές δεν έχουν μια ενιαία προσέγγιση ή άποψη για το τι θα έπρεπε να γίνει για την ενίσχυση αυτού του ανταγωνισμού μεταξύ οίκων αξιολόγησης. Και το επαναλαμβάνω δεν είμαι εμπειρογνώμων. Ωστόσο όμως ε, μου αρέσουν πολλές από τις προτάσεις ε, που έγιναν από τον κύριο Γκοζές και για διαφορετικούς ε, λόγους ακούγοντας αυτά τα οποία είπε νομίζω με σοφό και συνετό τρόπο τοποθετήθηκε δεν είμαι όμως εμπειρογνώμων και περιρίζομαι εδώ τώρα στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο εκπροσωπώντας τους πρασίνους ο κύριος Πασκάρ Καφάν παρακαλώ ε, Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στους πανελίστες, ε, γιατί θέλουν να ακούσουν τις ερωτήσεις μας, όχι να ακούσουν τη συζήτηση που κάνουμε μεταξύ μας, που μπορούμε να την κάνουμε και αργότερα. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν ε, μια παρατήρηση σχετικά με αυτά που είπε ο Ζαν Πολ Γκοζές, όχι κατά την έννοια του συναδέλφου των συντηρητικών, ε, ο Μισελ ε, Γκοζές, ήταν παλιά πιο φιλικός προς τις προτάσεις της Κομισιόν και του Μισελ Μπαρνιέ συγκεκριμένα. Ε, είπες ότι μία από τις προκλήσεις ήταν ε, να μην ανατροφοδοτείται το σύστημα από τις αξιολογήσεις των οίκων ε, θα ήθελα να επιστήσω προσοχή μας σε αυτά που ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του Finance Watch ε, γιατί, και τις προτάσεις ε, γιατί πραγματικά μας δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει να βγαίνει ένας μέσος όρος και επομένως να μην ενθαρρύνεται η αστάθεια και να μην υπάρχει αυτή η έννοια του marketing από κάποιους οίκους αξιολόγησης και κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αποτελέσει το χρυσό κανόνα ανάμεσα ε, και τον σωστό μέσο όρο ανάμεσα στον ανταγωνισμό και τα όρια του ανταγωνισμού έτσι ώστε ε, να ε, μην ενθαρρύνεται η αστάθεια των αγορών. Η πρόταση λοιπόν που έγινε από το Finance Watch πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα ο εκπρόσωπος του Finance Watch να μας δώσει την άποψή του σχετικά με ένα θέμα το οποίο αποτελεί επίκεντρο των συζητήσεων και των επικρίσεων. Το θέμα δηλαδή της εκπεριτροπής. Ο κύριος Φιλιππονά δεν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ήθελα την άποψή του. Και δύο ακόμα στοιχεία. Μία ερώτηση στην εκπρόσωπο της Société Générale γιατί ε, σαν να κατάλαβα ότι δεν συμφωνούσε με, ε, με το αντεπιχείρημα ε, ε, σχετικά με τον ανταγωνισμό των μοντέλων. Ο Στέφανο Κλίντ λέει είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα μοντέλα αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο περίπλοκα. Είναι ε, μοντέλα α πούμε τύπου μακροοικονομικών μοντέλων. Γιατί λοιπόν από τη στιγμή που αξιολογούμε τα μακροοικονομικά μοντέλα, γιατί να μην αξιολογούμε και τα μοντέλα των οίκων αξιολόγηση, ενδεχομένω χωρί μια τελική επιβεβαιωτική σφραγίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει χωρί εναρμόνιση να υπάρχει τουλάχιστον συνέχεια και συνέπεια ε, στα μοντέλα. Θα ήθελα την ε, άποψη της εκπροσώπου του Σοσιατέ Γενεράλ και, εν πάση περιπτώσει, να απαντήσει στα αντεπιχειρήματα που ακούστηκαν. Τελευταίο σημείο αφορά την πρόταση που έγινε από τον κύριο Κράλ και που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της γραπτής του παρέμβασης. Εάν κατάλαβα καλά, ε, ε, να γίνει μια προσπάθεια επίλυσης των... των Σύγκρουση συμφερόντων που φαίνεται ότι δεν λύνονται τελικά. Ε, εγώ θα μπορούσα να προτείνω και ένα τρίτο δρόμο. δεν, γιατί, ξέρετε, η τελευταία παράγραφος του γραπτού σας κειμένου δεν είναι πάρα πολύ σαφής. Έχω λίγο χρόνο ακόμα, επομένως ακόμα ένα σημείο. Ε, λέμε συχνά ότι είναι θερμόμετρα η οικοί αξιολόγηση. Όχι, δεν είναι θερμόμετρα. Είναι γιατροί που χρησιμοποιούν δείκτε. Οι δείκτε είναι τα θερμόμετρα. Ε, ε, και επομένω είναι γιατροί οι οποίοι κάνουν διάγνωση και μετά προτείνουν, κάνουν προτάσει. Οι γιατροί κάνουν τι προτάσει. Ε, Όμω, γιατροί, εάν είχαν κάνει τόσα λάθη όσον αφορά την Ισλανδία, όσον αφορά την Ελλάδα, όσον αφορά τα subprimes, προ τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τα λάθη, τέτοιοι γιατροί, αλίμονο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν. Θα πρέπει να μειωθεί λοιπόν ε, ε, το βάρος της αξιολόγησης των οίκων και ελπίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ε, ρωτώ λοιπόν πώς είναι δυνατόν να περιορίσουμε αυτήν την πλευρά της ιατρικής διάγνωσης των οίκων αξιολόγησης και να περιοριστούν σε ένα ρόλο αξιολόγησης κινδύνων. Ε, ας πούμε ε, να μας πούν εάν ναι να κάνετε αξιολόγηση κινδύνου πολύ ωραία αλλά να μην κάνετε συστάσεις είτε οι συστάσεις μου αρέσουν είτε δεν μου αρέσουν ε, αυτό ρώτησα και η πρώτη αντίδραση του εκπροσώπου της Μούντις όταν είπα την πρόταση αυτή με κατέπληξε γιατί είπε ναι γιατί όχι Μία από τις συστάσεις ας πούμε για την ε, Γαλλία ήταν να γίνει πιο ευέλικτη η αγορά εργασίας. Ε, η Standard Poor's ενδεχομένως μπορεί να έχει ε, γνώσεις όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί οι αναλυτές της Standard Poor's έχουν την ικανότητα να πούν ε, η συνταγή είναι να κάνετε πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας. Αυτό πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και επομένως θα, θα πρέπει να μας δώσετε, αυτό θα ήθελα από τους εμπειρογνώμονες, να μας δώσουν την αξιολόγησή τους, εάν πρέπει να μείνουν στην αξιολόγηση κινδύνου ή να κάνουν και συστάσεις ευχαριστώ πολύ. Ο Πόρτας, ε, εξ ονόματος Ενωτικής Αριστεράς, παρακαλώ, κύριε Πόρτας. Ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις και μετά κάποιες ερωτήσεις ε, για αποσαφήνιση κάποιων πραγμάτων. Πρώτο, πρώτη παρατήρηση για το κρατικό χρέος που νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο καθιστά απόλυτα αναγκαία και επίγουσα αυτή τη συζήτηση γι' αυτό. Από όσα άκουσα, συνεχίζετε να σκέφτεστε ότι δεν υπάρχει λύση για την αντιμετώπιση της κρατικής υπερχρέωσης που να μην είναι το να εξεταστεί το κρατικό χρέος ως προϊόν, χρηματοοικονομικό προϊόν που θα πρέπει να αξιολογείται ή όσον έχουμε εδώ και αλλαγή αξιολόγησης ή προφανώς όλες οι άλλες λύσεις δεν επιλύουν, λένε, ε, ουσιαστικά το πρόβλημα. Ισχύει αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτό σε σχέση με όσα ανέφερε ο κύριος από τον Ιαπωνικό οργανισμό. Θα ήταν αναγκαία λοιπόν η ύπαρξη μιας δημόσιας συνιστώσας, μιας, ενός, μιας δημόσιας υπηρεσίας σε σχέση με τις, κρατικές, με τις ιδιωτικές μας συγχωρείτε, υπηρεσίες αξιολόγησης. Θα ήθελα να διευκρινιστεί. Περί πρόκειται για συμμετοχή στο κεφάλαιο είναι η αναφορά αυτή ή πρόκειται για οποιοδήποτε τρόπο ουσιαστικά με την ε, ε ανάμιξη σε σχέση με την ε, έδρα ή τη δημόσια αρχή του κράτους ε, στην οποία θα βρίσκεται μια τέτοια υπηρεσία. Ερωτώ όλα αυτά, επειδή στη συζήτηση για το θέμα για το θέμα της ύπαρξης μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας αξιολόγησης έχω τις μεγαλύτερες αμφιβολίες <clears throat> για το αν θα πρέπει να προαχθεί με δημόσια κονδύλια. Διότι διήθατερον ένα από τα δύο θα γίνει. Ή θα υπάρχει μια δημόσια αρχή ευρωπαϊκή αξιολόγησης και τότε δεν ξέρω πώς θα μπορεί να βρει ή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην αγορά σε σχέση με, την, ε, ε, με ένα ε, χρονικό διάστημα 20 30 ετών ή μια ιδιωτική υπηρεσία όπου θα πρέπει να υπάρχει ο συνεισφέρον. Εκεί τι θα γίνει. Ε, το δημόσιο θα συνεισφέρει σε σχέση και με την δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας. Διότι εδώ ε, έχουμε πολύ παρόμοια, έχουμε συγκρίσιμα πρότυπα μαθηματικά όσον αφορά την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Θα ήθελα λοιπόν ο υπεύθυνο από τον Ιαπωνικό οργανισμό να επεξηγήσει καλύτερα τι θα είναι αυτό το οποίο εννοεί ως δημόσια συνιστόσα ή δημόσιος οργανισμός, κρατικός οργανισμός σε σχέση με υπηρεσία αξιολόγησης. Μια τρίτη ερώτηση στη συνέχεια. η δημοσιος οργανισμος κρατικος οργανισμος σε σχεση με υπηρεσια αξιολογησης μια τριτη ερωτηση στη συνεχεια δεύτερη, δεύτερη ερώτηση προς τον την εκπρόσωπο της Société Générale που ήταν σαφέστατη στις παρατηρήσεις που έκανε και είπε ότι οι οίκοι αξιολόγηση μεροληπτούν υπέρ κάποιων κρατών. Θα ήθελα να μου πει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι εννοεί αυτή την τοπο, με αυτή την τοποθέτησή της. Τι ήθελε να πει, τι εννοεί με αυτή. Και τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Finance Watch τι είναι εκείνο το οποίο ήθελε ακριβώς να πει. Ακριβώς να πει. Με μια γνωμοδότηση λέει που δεν θα επηρεάζει. Διότι περί τίνος πρόκειται. Είναι σαφές πιστεύω ότι σήμερα η οίκη αξιολόγηση είναι ρυθμιστικές αρχές σχεδόν. Καθορίζουν τους όρους και τις συνθήκες της αγοράς ε, με αυτές τις ε, δράσεις τους. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αποσυρθεί, να αφαιρεθεί αυτή η εξουσία επηρεασμού και επιρροή σε σχέση με μια τέτοια αξιολόγηση από πλευρά σου. Δεν το κατάλαβα καλά από τα όσα είπατε. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε ε, Πόρτας. Πιέζει πολύ ο χρόνο, είναι πολύ περιορισμένο. Θα δώσουμε τον λόγο σε εκείνου που ζήτησαν τον λόγο. Ο κατάλογο είναι. Φιρμάντα Μπαλθίτη, el señor el señor Diego Follo, el señor Peter Simon, la señora Podimata, el señor Langen y el señor Κάποιο άλλο επιπλέον. Εδώ λοιπόν κλείνει ο πίνακα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Τόμα Μαν και θα σα ζητούσα παρακαλώ να προσαρμοστείτε στα δύο λεπτά ω όριο στι παρεμβάσει σα. Δύο λεπτά στην παρέμβασή σα, διότι πιέζει πολύ ο χρόνο. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Μαν λοιπόν έχει τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ έχω το ρολόι, θα το λάβω υπόψη τον χρόνο, δεν θα ξεπεράσω το όριο. Βρήκα ενδιαφέρον αυτό το οποίο αναφέρθηκε από την κυρία Λόνη ότι υπάρχει λέει εξαιρετικό ανταγωνισμό. Όχι για του μεγάλου τρει οίκου αξιολόγηση, αλλά οι του Φιτς εργάστηκαν λέει και συνεισέφεραν για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ε, ύπαρξή τους. Για μένα ήταν μια ομάδα αυτοί οι τρεις. Αυτό είναι κάτι λοιπόν αξιόλογο. Ζωάν Πολγκοζές έχεις δίκιο. Οι υπηρεσίε αυτέ συντάσσουν κάποιε γνωμοδοτήσει και επηρεάζουν τα πράγματα. Στην πολιτική έχουμε ένα τεράστιο χώρο. Με κάθε υποβάθμιση κρατών έχουμε κάποια σύνοδο κορυφή στη συνέχεια, έχουμε ε, προσπάθειες που γίνονται για να βρεθεί λέει, μια λύση. Έτσι όμω δεν μπορούμε να εργαζόμαστε. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριο Κλίντ. Πρέπει να δούμε με ηρεμία και νυφαλιότητα να πετύχουμε, να δαμάσουμε, να τυθασέψουμε την επιρροή αυτή των οίκων αξιολόγηση. Μία πρόταση είναι η ανακύκλωση, η ανακυκλούμενη αξιολόγηση. Έχω επιφυλάξει. Εσεί προτείνατε μια ε, εναλλακτική λύση. Ο Βόρκαν Σόιμπλε είπε το 2009 ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία αξιολόγηση και όχι μία που θα δίνει ε, απλά και μόνο κάποια καλύτερα αποτελέσματα αλλά που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Πραγματικά σύμφωνη λοιπόν για την ανεξαρτησία. Και σε σχέση με την προέλευση αυτής της πρότασης έχουμε και την πρόταση ενός ιδρύματος που θα δημιουργηθεί 300 εκατομμύρια ευρώ Θέλετε λέει με διαφορετικό τρόπο να δράσετε. Τι θα γίνει διαφορετικά όταν δεν θα υπάρχει επηρεασμό. Αν μπορείτε να διασφαλίσετε αυτή την ανεξαρτησία, θα είσαστε πρόθυμοι να είσαστε υπεύθυνοι για τι επιπτώσει των αξιολογήσεών σα και μέχρι πού θα φτάνετε. Τι θα γίνει με τη διαφάνεια. Τι θα γίνει διαφορετικά από ό,τι μέχρι σήμερα σε σχέση με του τρει μεγάλου οίκου αξιολόγηση. Είπατε ότι πιθανώ λέει θα πρέπει να αποκαλυφθούν κάποιε μεθοδολογικέ προσεγγίσεις και μέθοδοι. Πώ θα γίνει αυτό, ποιε μέθοδοι θα όταν έχουμε αποτελέσματα τα οποία σίγουρα μπορεί να έχουν κάποιο αρνητικό χαρακτήρα σε επιπτώσεις τους, θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα με τη διασφάλιση λέει, τον της ανεξαρτησίας. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει δεν θα είχα πρόβλημα, αλλά πρέπει από κοινού να ρυθμίσουμε τους κανόνες. Πρέπει με τον ίδιο τρόπο να μπορούμε να δράσουμε. Χρειαζόμαστε όμως όρους και προϋποθέσεις για να υπάρξουν αποτελέσματα. Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει δράση όπως μέχρι σήμερα, αλλά θα ξεκινάμε από αξιόπιστα σαφή στοιχεία. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Πραγματικά δημορώ να ακούσω τι θα μας προσφέρετε ως απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Μάν. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρονικό όριο. Τώρα ο κύριος Μπαλφίτης. Παρακαλώ δύο λεπτά. Ačiū Ευχαριστώ. πρόεδρε, e, συνάδελφοι. Μία προοπτική σε σχέση με αυτά τα θέματα και ως υπουργό ε, Οικονομικών ε, θυμάμαι ότι σε σχέση με την αξιολόγηση της χώρας μας ε, από πλευράς των οίκων αξιολόγησης και αξιολόγησης δεν είναι μόνο απλά μια εταιρεία οι αξιολογήσεις αυτές έχουν τεράστιες επιπτώσεις, πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση οποιασδήποτε αξιολογούμενης χώρας. Υπάρχει μεγάλη επίπτωση όσον αφορά και τις ίδιες τις τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης επηρεάζουν αυτές οι αξιολογήσεις το διεθνές κύρος ή την διεθνή θέση μιας τέτοιας χώρας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 2008 και σε μεγάλο όγκο κιόλας έχει παρέμβει επειδή οι αξιολογήσεις κάποιων χωρών υποβαθμίστηκαν. Καλωσορίζουμε λοιπόν την πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκροτηθεί μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία ως Ευρωπαϊκός Οίκος Αξιολόγησης και υποστηρίζουμε επίσης και τον ε, φίλο από την Ιαπωνία στα όσα προτείνει. Και θεωρώ ότι όσοι εργάζονται για την συγκρότηση αυτού του οικοαξιολόγησης θα πρέπει να εργάζονται και να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εργασία τους, το έργο τους θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οίκοι αξιολόγηση όχι μόνο έχουν μεγάλο βάρο παγκόσμια, αλλά έχουν και πρόσβαση σε πάρα πολύ σημαντικέ πληροφορίε ω στοιχεία. Είναι λοιπόν η χρονική στιγμή να αντιληφθούμε ότι πρέπει να ανταγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε στη διεθνή αγορά και η οίκοι αξιολόγηση είναι ένα από τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο να αυξηθεί, να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά μα παγκόσμια. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιε ίσονο σημασία επιφυλάξει για τεχνικά θέματα, όπω θέματα εποπτεία για παράδειγμα, ή την ε, ε, συγκέντρωση, ε, συμπίκνωση στι αγορέ. Γενικά όμω έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία και αυτή πρέπει να δράξουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπαρφίτη. Στη συνέχεια ο κύριο Μιγόλ παρακαλώ. Δύο λεπτά. Μάλιστα, ευχαριστώ. Καταρχήν πρώτα ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Και ευχαριστώ πολύ και για το μεγάλο ταξίδι που κάνατε από την Ιαπωνία μέχρι εδώ στην Ευρώπη στις Βρυξέλλες. Δεν το κάνει κανείς καθημερινά αυτό. Κάποιες σύντομες ερωτήσεις προς εσάς πρώτα κυρία Ρώσα. Δεν ήμουν σίγουρος όσα είπατε για, τις, για τις, ε, τους ελέγχους ε, όσον αφορά τις, τους οίκους αξιολόγησης και για την έκθεση. Τον κύριο Μαγιόρ τον κατάλαβα τότε ότι μια μεγάλη λέει έκθεση ε, διακρύβωση θα γινόταν και όχι μόνο γιατί της στους συγκεκριμένους ελέγχους. Για την ίδια την αγορά. Θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχει μια συνολικότερη έκθεση από πλευρά τη ΕΣΜΑ για την αγορά αξιολογήσεων με περιπτώσεις συγκρουόμενων συμφερόντων, με τριβές που υπάρχουν και πιθανά προβλήματα που υφίστανται σε αυτό το πεδίο. Θα ήθελα από εσά να μου πείτε σε ποιο πλαίσιο ε, θα γίνει αυτή η μελέτη, αυτή η έκθεση, πότε θα δημοσιευτεί, πότε θα είναι διαθέσιμη. Η δεύτερη ερώτηση την οποία έχω να διατυπώσω επανειλημμένα αναφέρθηκε αφενός λόγω της μεγάλης συμπίκνωσης στις αγορές και από την άλλη πλευρά λόγω πιθανών αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων που με κανένα πρότυπο όμως δεν μπορούν να αποφευθούν σήμερα. Θα συμφωνούσα λοιπόν. Ταυτόχρονα είναι σαφέ ότι δεδομένη της υψηλή συμπίκνωση στις αγορές θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μεγαλύτερο πλουραλισμό, ένα πιο πλουραλιστικό πρότυπο. Και πράγματι το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεση του Wolfgang Klintz τοποθετήθηκε υπέρ τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγηση, που σαφώ θα είναι υπέρ του κοινού συμφέροντο, του συμφέροντο δηλαδή της κατά δύναμη, της ε, δυνατής αξιολόγησης Τώρα στη δική σας πρόταση ε, από πλευράς Μπέργκερ και ε, άλλων θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Σημαντικά κονδύλια ε, πρόκειται να αναλωθούν ώστε οι χρηματοοικονομικοί παράγοντες να μην έχουν δυνατότητες ε, τέτοιας παρέμβασης και επιρροής. Και δεδομένο, δεδομένης της κερδοφορίας που υπάρχει στην αγορά αξιολογήσεων, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα τέλος το οποίο θα επιβάλλεται, ώστε να δημιουργηθεί ένα ταμείο για αυτό το ίδρυμα. Διότι όταν έχουμε 40% κερδοφορία, κάτι θα έπρεπε να λειτουργήσει υπέρ του κοινού συμφέροντος. Και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του Ιδρύματος, το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σβέν. Στη συνέχεια ο κύριος Φεγιό παρακαλώ δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα περάσω αμέσως ε, στις ερωτήσεις που έχω. Ένα από τα θέματα που δεν καλύπτεται στην πρόταση που έχουμε εδώ επί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συσχετίζεται με τη χρηματοδότηση των ε, οίκων αξιολόγησης. Όπως ε, πολύ καλά ανέφερε πριν από λίγο ο συνάδελφος Ζαν Πολ δεν είναι απλό αυτό το θέμα καθόλου. Η συγκεκριμενοποίηση, η εξειδίκευση αυτού του θέματος ε, δεν έχει προφανή ακόμα αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να μου πείτε εσείς από πλευρά σας είναι αν συμφωνείτε σε σχέση με τη σημερινή χρηματοδότηση όσοι υπάρχει σήμερα ή μήπως θα ήταν σημαντικό να πορευτούμε να πορευτούμε προς μια χρηματοδότηση που θα γίνεται από τους ίδιους τους επενδυτές και πώς αυτή η χρηματοδότηση θα μπορούσε να διαμορφωθεί συγκεκριμένα. Το δεύτερο θέμα σε σχέση με την αναφορά από πλευράς ΡΟΣ όσον αφορά την λειτουργία της αγοράς διότι εφιστώ την προσοχή για την ανάγκη, την ανάγκη αξιοπιστίας για τους οίκους αξιολόγησης και από την άλλη πλευρά για την σωστή λειτουργία της αγοράς με περισσότερες, περισσότερους εμπλεκόμενους στην αξιολόγηση από όσους υπάρχουν σήμερα. Να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν ήδη κάποιες πιστοποιήσεις από διάφορους οίκους αξιολόγησης πέρα από αυτούς τους τρεις μεγάλους οίκους. Πώς θα βλέπατε την δυνατότητα να λειτουργήσουν από κοινού σαν ένα σύνολο, διαδικτυωμένοι όλοι αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης και να δημιουργηθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά. Τρίτον, και ολοκληρώνω, υπάρχουν διάφορες αναφορές ε, στην ρυθμιστική και νομοθετική λειτουργία όσον αφορά τις αξιολογήσεις, χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις. Οι ίδιοι εδώ οι νομοθέτε θα πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη. Είναι δυνατόν να τροποποιηθούν αυτές οι νομοθετικέ ρυθμίσει, οι ρυθμιστικέ αυτέ διατάξει, σε μια πρώτη φάση να έχουμε αυτή την τροποποίηση, α το πω έτσι, ώστε να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση τη αγοράς, μια και υπάρχει εξάρτηση σε σχέση με του οίκου αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριο Σάιμον. Πείτε δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση στον κύριο Κράλη και μετά προς τον Φιλίπ. Κύριε Κράλ, στο δικό σας έγγραφο αναφερθήκατε στην κατάσταση της δομής ε, ιδιοκτησίας ή κυριότητας σε σχέση με τους οίκους αξιολόγησης και για τον μονοπωλιακό ρόλο τους. Προφορικά όμως ε, αναφερθήκατε και είπατε ότι υπάρχουν λέει συγκρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τους οίκους αξιολόγησης. Με βάση τη δομή κυριότητας ή ιδιοκτησίας. Ίσως θα μου ευγνώμων αν θα μπορούσατε αυτά να τα επεξηγήσετε ε, περαιτέρω και θα ήθελα να πω ότι θα ήμουν ευγνώμων για την αξιολόγησή σα, αν με βάση τη δομή κυριότητα ή αξιολόγηση των οίκων αξιολόγηση, υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα ίσω που μπορεί να ε, ελοχεύουν που για τον χρήστη θα μπορούσε να είναι βλαπτικά ε, για τη μία ή άλλη συγκυρία αξιολογηση οπω συμβαίνει. Ευχαριστώ. Yes. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σάιμον. Στη συνέχεια η κυρία Ποδηματά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπήρξε μια ε, φράση στην ε, ήταν εξαιρετικές και πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι εισηγήσεις υπήρξε μια φράση στην παρουσίαση του κυρίου Ουτσούμη που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Ουτσούμη παρέπεμψε σε μια φράση του καθηγητή του του MIT, του κυρίου Γκουστάβο Μάνσο, την οποία την επαναλαμβάνω διότι θεωρώ ότι έχει τεράστια σημασία. Είπε λοιπόν ότι The rating agency Ο οίκος αξιολόγησης θα πρέπει αφενός να, αποτυπώνει ένα έναν ακριβή πίνακα της ε, κατάστασης αλλά και την, ε, το γενικότερο πλαίσιο ε, ύπαρξης της εταιρείας ή του κράτους στην οποία λειτουργεί η εταιρεία αυτή. Γιατί Ε, εάν δεν αξιολογηθούν ε, σωστά αυτά τα πράγματα ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε ανακρίβεια. Τι αφορά τι αξιολογήσει του δημόσιου χρέου, τι αξιολογήσει χωρών, πολύ περισσότερο ε, από ότι όταν μιλάμε για τις αξιολογήσεις εταιριών. Και πάλι παραπέμποντας στην παρέμβαση του κυρίου Ουτσούμη και το ερώτημά μου απευθύνεται προς την ΕΣΜΑ ε, ο κύριος Τσούμι είπε ότι ε, μιλώντας για τις αξιολογήσεις του δημόσιου χρέους έχει πολύ μεγάλη σημασία να λαμβάνεται υπόψη ε, ο δημόσιος χαρακτήρας της αξιολογήσης η διάσταση δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος ακριβώς επειδή οι αξιολογήσεις επηρεάζουν έχουν επίπτωση στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων εκατομμυρίων πολιτών επειδή αυτό είναι ένα ζήτημα κεφαλαιόδου σημασία, πολύ επίκαιρο στι μέρες μας ήθελα να ρωτήσω πρωτίστω εσάς αλλά και όποιον άλλον από τους ε, ομιλητές που συμμετείχαν στο πάνελ ε, πρώτα απ' όλα αν συμμερίζεστε την αναγκαιότητα να διασφαλίσουμε αυτή την αρχή τη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι αξιολογήσει χωρών πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό ε, μπορούμε να το κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μέσω της δημιουργίας ενός δημόσιου οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπως συζητάγαμε στην ευρώπη. μία λύση θα ήταν αυτό που πρότεινε ο επίτροπος μπαρνιέ και δεν υιοθετήθηκε να αναστέλλεται προσωρινά η αξιολόγηση των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε κυρία Ποδηματά. Ο κύριος Λάγκε, δύο λεπτά παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Τα επιχειρήματα δεν θέλω να τα επαναλάβω. Όμως πιστεύω ότι η υπερβολική εξάρτηση από αξιολογήσεις των οίκων αξιολογήσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεκινώντα όσον αφορά την αναχρηματοδότηση μέσω τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που προϋποθέτει κάποια αξιολόγηση από οίκους αξιολόγηση. Είναι απόφαση λοιπόν των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μπορεί να απαγκιστρωθούμε από αυτή την κατάσταση. Ερωτώ τους συμμετέχοντες, εισηγητές, πώς κρίνεται την ε, ε, δράση στη ΣΥΠΑ που απαγορεύει ρητά στην αξιολόγηση και εποπτεία τραπεζών να έχουμε εξωτερικά ratings, εξωτερικές δηλαδή αξιολογήσεις. Το αντίστροφο έγινε σε σχέση λοιπόν με τους Lehman Brothers. Δεν γίνεται όμως συζήτηση γι' αυτό. Το δεύτερο ερώτηση, μεγαλύτερη διαφάνεια που πρέπει να διασφαλιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ενιαία κριτήρια πρέπει να υπάρξουν. Η κυρία Ρος, βλέπετε να είσαστε σε θέση κάπως να δημιουργηθούν ενιαία κριτήρια. Σε αυτά δεν θα έπρεπε να ανήκει και μια επισκόπηση μια επισκόψη για τα τέλη ή τις δομές ε, χρηματοδότησης ε, και εισφορές. Ε. Ανήκει υποχρεωτικά νομίζω στο ότι για ένα κράτος ένας οίκος αξιολόγησης μπορεί να είναι πιο φθηνός εντός εισαγωγικών από ότι σε σχέση με κάποιον επενδυτή. Και τρίτον, ο κύριος Κράλ μίλησε στο τέλος της εισήγησής του ότι ανεξάρτητες πλατφόρμες πρέπει να δημιουργηθούν και μέσω της ε, δράσης των οίκων αξιολόγησης μέσω μιας τέτοιας κεντρικής πλατφόρμας. Τι εννοούσε ο κύριος Κράλ με αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος Νιόκ παρακαλώ δύο λεπτά. Merci. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κάποιε ερωτήσει και δύο παράδοξα. Πρώτη ερώτηση. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι σε μια χρηματοπιστωτική αγορά μπορούμε να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτήν την αγορά είναι η αβεβαιότητα και οι οίκοι αξιολόγηση υποτίμησαν του κινδύνου των subprimes και τώρα υπερτιμούν τον κίνδυνο του δημοσίου χρέου. Όσον αφορά το δημόσιο χρέο, μια δεύτερη ερώτηση. Αρκετοί παρεμβαίνοντε μίλησαν για τα συγκρουόμενα συμφέροντα στο μοντέλο που πληρώνει ο εκδότης. Όμως ε, το μοντέλο που είναι ακόμη χειρότερο από το μοντέλο του ότι ο εκδότης πληρώνει είναι ο προσυπογράφων, αυτός που αγοράζει που πληρώνει. για να μπορούν να ζητήσουν ε, ε, πολύ υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου. Άλλη μια ερώτηση. Μπορούν οι οίκοι αξιολόγηση να είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένοι από τα ελεγκτικά συνέδρια για να αξιολογούν το δημόσιο χρέο. Και τέταρτη ερώτηση σχετικά με τις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Σε ποιο μακροοικονομικό μοντέλο βασίζεστε για να κάνετε τις προβλέψεις σας μακροοικονομικά μοντέλα και μοντέλα αξιολόγηση κινδύνου δεν είναι τα ίδια, θα ήθελα να πω και προ τον φίλο Ζαν Πολ Μακροοικονομικά μοντέλα μπορεί να χρησιμοποιούνται βασιζόμενα σε επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία. Εσεί σε τι μοντέλα στηρίζεστε και ως προς τι είναι καλύτερα από τα μοντέλα που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οίκοι αξιολόγηση ε, θέλουν να κάνουν συστάσεις. Βλέπουμε όμως τις συστάσεις που κάνουν και εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένα παράδοξο. Δεν νομίζετε ότι υπάρχει ένα παράδοξο σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι είναι σε ύφεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο το χειρισμό των χρεών και ταυτόχρονα υποχρεώνονται τα κράτη σε πολιτικές λιτότητας. Άλλο ένα παράδοξο είναι ότι Μιλάμε για ανταγωνισμό, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο ανταγωνισμός ωφελεί τα μονοπόλια. Και μια τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα να μου πείτε το μοντέλο του ότι ο ιδιώτης εκδότης πληρώνει, γιατί να μην επιφέρει και το ότι ο δημόσιος εκδότης πληρώνει έχοντας έναν δημόσιο οργανισμό αξιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πιστεύω ότι τα δύο προβλήματά μας, τα, τουλάχιστον τα δικά μου δύο μεγαλύτερα προβλήματα, είναι το πρόβλημα της υπερβολικής συγκέντρωσης ή συμπίκνωσης στις αγορές και το πρόβλημα που συνεπάγεται το πώς μπορεί να υπάρχει ένα αποτελεσματικό ανταγωνιστικό κλίμα ε, περισσότερος ανταγωνισμός ε, από πλευράς ε, αναφοράς θα ήθελα να μας αναφερθεί πόσες αυτές τις υπηρεσίες αξιολόγησης υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν καταχωρηθεί. Ποια είναι τα κύρια εμπόδια για την πρόσβαση και πώς μπορούν να μειωθούν αυτά τα εμπόδια. Και αν δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει εδώ αυτό το οποίο λειτουργεί στην διαχείριση ανταγωνισμού ουσιαστικά. Δηλαδή περιορισμός όσον αφορά ποσοστώσεις στην αγορά. Δηλαδή, ρύθμιση όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχή στην αγορά, όσον αφορά τα όρια πρόσβασης. Το δεύτερο θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί είναι το θέμα της αξιολόγησης του εθνικού χρέους το εθνικό κρατικό χρέος και όσον αφορά τη δράση των υπηρεσιών αξιολόγησης δημιουργούνται προβλήματα τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ την αξιολόγηση ιδιωτών και διαρωτώ με αν μήπως εδώ έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του εκδότη και του πληρώνοντας ε, Στο κρατικό χρέος υπάρχουν δράσεις στην αγορά που απαιτούν και ε, εξαρτώνται από την αξιολόγηση τα CDS, Credit Default ε, Swaps ε, και τα θέματα υπερχρέωσης ε, κάποιων κρατών βρίσκονται ως λόγοι πίσω από αυτές τις αξιολογήσεις ως εξηγήσεις. Και έχουμε εδώ και το θέμα και της συγκυρίας, χρονικής συγκυρίας και την ίδια την αξιολόγηση. Πρέπει να δούμε αν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει παρέμβαση για τέτοιου είδου αξιολογήσει γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φεραίρα. Τώρα θα ήθελα να δώσουμε τον λόγο στους ε, πραγματογνώμονες. Πρώτα για τις αναφορές που έγιναν στην ίδια την κυρία Ρος. Πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θα δώσω δύο λεπτά. Δύο λεπτά σε καθέναν από εσάς και μετά θα ολοκληρώσει ο εισηγητής για την έκθεση αυτή, ο κύριος Ντομινίτσι. Κυρία Ρο, δύο λεπτά παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο γίνεται περισσότερε ερωτήσει, αλλά βεβαίω δημερό μπορώ να απαντήσω σε οποιονδήποτε ε, δεν έχει πάρει απάντηση, γιατί σε δύο λεπτά δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Συμφωνώ απολύτω ότι η σημασία των οίκων αξιολόγηση έχει ξεπεράσει κάθε ε, προσδοκία ή επιθυμία ή λογική. Είναι, θα πρέπει λοιπόν σιγά σιγά βαθμιαία να αντιστρέψουμε την τάση αυτή. Είναι δύο οι τρόποι και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να δει του δύο αυτού δρόμου όμως τι δύο δυνατότητε. Η μία είναι αύξηση τη ανταγωνιστικότητας και δεύτερον είναι η μείωση τη ε, ε, ε, βάση τη εμπιστοσύνη που δίνεται εις στην αξιολόγηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή πολλέ καταγραμμένε εταιρείε αξιολόγηση. αλλά οι περισσότερε είναι οι οικοί οι οποίοι βασίζονται και δρούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. σαφε είναι πολύ λίγοι οι κυρίαρχοι τη παγκόσμια αγοράς είναι δυνατόν να υπάρχει δίκτυο ε, ε, ε, αξιολόγηση, ή θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να δουλέψουν πολύ οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί η βάση, η αξιοπιστία που δίνεται στην αξιολόγηση των οίκων. Ε, Βεβαίω, κοινό παρονομαστή όλων είναι η αύξηση τη διαφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να δούμε πώ είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι υφιστάμενε προτάσει, τι οποίε αναφέρθηκαν πολύ, αλλά ε, ποιε είναι και οι επιπλέον ε, διαδικασίε, επιπλέον μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμό στην αγορά και να μειωθεί η βάση που δίνεται σε αυτά τα ε, στοιχεία και σε αυτή την αξιολόγηση. Εμείς ε, ε, κάνουμε βάση και του κανονισμού ήδη από την αρχή Ιανουαρίου του 2011 πληθώρα εκθέσεων. Εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως στο αποτέλεσμα της έρευνας που κάναμε τον Δεκέμβριο και θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα στο τέλος του πρώτου τετραμήνου του 2011. Για τα υπόλοιπα θα απαντήσω Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο ε, Γκαγιό. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Oui, ε, je... Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Φερέιρα όσον αφορά το ζήτημα των περιορισμών των τμήματων ε, της αγοράς, τα μερίδια αγοράς δηλαδή νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε κάποια μέτρα ε, ή τέλος πάντων κάποιους τρόπους ε, που θα αναφέρονται στο νέο κανονισμό ε, έτσι ώστε να περιοριστούν τα μερίδια της αγοράς. Μπορούμε διμερώς περαιτέρω να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Όμως πιστεύω ότι αυτό είναι ένας δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι ένα καλό ενδεχόμενο. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω. Μετά από την ε, παρατήρηση ενός παρεμβαίνοντος βουλευτού σχετικά με το θερμόμετρο και τον ε, γιατρό, είναι πολύ σωστή η εκτίμηση που έκανε. Και νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ότι κάνουν συστάσεις οι οίκοι αξιολόγησης από πολιτικής απόψεως. Βεβαίως αυτό είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ε, και θα πρέπει οι συστάσεις των ε, ε, οίκων αξιολόγησης ε, να αφορούν μονάχα κάποιες εσωτερικές κοινοποιήσεις στα εμπλεκόμενα μέρη κυρίως όταν μιλάμε για θέτηση ή για χρεοκοπία και για δημόσιο χρέος ακόμα περισσότερο και να μην κοινοποιούνται. Ε, ε, γιατί βεβαίως ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να σοκάρει. Από τη στιγμή που πρόσφατα είδαμε ας πούμε πράξεις της Άντερεν που μπορούν να θεωρηθούν ανάμεξη στις ιστορικά των χωρών. Επίσης, όσον αφορά την αξιολόγηση ε, με γράμματα της αλφαβήτου. Ε, ναι, οι πρώτες ε, αξιολογήσεις είχαν γίνει έτσι, γιατί θέλαμε αρχικά και αυτό ξεκίνησε στις ΗΠΑ με τρόπο έτσι λίγο πιο χαλαρό ε, και ο νομοθέτης ε, τότε στην αρχή των οίκων αξιολόγηση, ο νομοθέτης της ΗΠΑ ε, είχε προβλέψει ότι θα υπήρχε και ένα περιθώριο όσον αφορά την αξιολόγηση των οίκων. Αλλά έκτοτε προσκοληθήκαμε στο γράμμα και όχι στο πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσούνη, έχετε τον, Τσούμι, έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Uh, Άκουσα τα σχόλια σε σχέση με αυτό το οποίο ανέφερα, ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα πρέπει να έχουν και κάποια πτυχή που να σχετίζεται με το δημόσιο. Όταν λέω με το δημόσιο, δεν, λέω ότι θα πρέπει να ε, διαβουλεύονται με το δημόσιο. Θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι και επιμένω στην ανεξαρτησία. Αλλά το πνεύμα και η, βασική αρχή της ε, αξιολόγησης ε, είναι αυτή. Ο οίκος αξιολόγησης πρέπει να εμπεριέχει και μια πτυχή δημοσίων στοιχείων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στον τραπεζικό τομέα, ο τραπεζικός τομέας είναι ιδιωτικός. Πολλοί λένε όμως ότι υπάρχει και μια πτυχή δημοσίου τομέα στις τράπεζες και η φούσκα των ακινήτων που δημιουργήθηκε από τραπεζική συμπεριφορά στην ε, Ιαπωνία και η κρίση των subprime των ακινήτων ε, στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες πάλι από τον τραπεζικό τομέα προκλήθηκε. Τράπεζες που λησμόνησαν εντελώς το δημόσιο αγαθό, το δημόσιο τη δημόσια πτυχή που θα έπρεπε να έχουν. Αυτό εννοώ όταν λέω θα πρέπει να υπάρχει και μια δημόσια πτυχή στους οίκους αξιολόγησης. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσόμη. Ο κύριος Φιλιππονά, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, okay. Is this good now? Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω στα δύο λεπτά τις απαντήσεις μου για όλες τις ερωτήσεις. Κάτι φαίνεται να προκύπτει αυτά που λέμε. Μιλάμε για το δημόσιο όφελος, για το δημόσιο συμφέρον και γι' αυτό υπάρχει συνένεση. Και αυτό μας οδηγεί στο θέμα της εκπεριτροπής αξιολόγησης. Μας φέρνει στο θέμα των ολιγοπολίων και μας φέρνει και στο θέμα του πώς θα δίδεται μια γνώμη, μια αξιολόγηση που δεν θα έχει επίπτωση στην αγορά. Για το θέμα της εκπεριτροπής αξιολόγησης είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε την κριτική κατά της αρχής της εκπεριτροπής αξιολόγησης. Η αγορά της αξιολόγησης είναι ολιγοπόλιο, όπως είπαμε. Επομένως, αν υπάρχει εκπεριτροπής αξιολόγηση, ανοίγουμε την αγορά σε οίκους εκτός του ολιγοπολίου, που εξορισμού δεν έχουν την ίδια φήμη και το ίδιο κύρος και επομένως είναι λιγότερο αξιόπιστη και άρα δεν είναι ε, σωστή η τακτική αυτή. Ε, τεχνικά λοιπόν υπάρχει τεκμηρίωση για, αυτή, για αυτές τις κριτικές κατά της εκπεριτροπής ε, αξιολόγησης αλλά δεν είναι μια επιστολή αξιολόγησης είναι κάτι σαν δικαστική απόφαση. Όταν δώσουμε σε κάποιον την εξουσία να δίνει ετοιμιγορία ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει ε, χειραγώγηση ή ε, ε, σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι κανείς δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να δίνει ετοιμιγορία. Θα πρέπει να έχουμε κάτι τεχνικό, αλλά όχι τόσο συγκινησιακό, όπως λέμε πιθανότητα θέτησης. Ένας αριθμός θα μπορούσε να δίδεται. ώστε να έχει τελικά το αποτέλεσμα που θέλουμε. Υπήρξε και μια ερώτηση σχετικά με τα χρονικά περιθώρια. Δεν υπάρχει καμία θεωρία συνωμοσία για το αν ε, έγιναν επίτηδες ή όχι. Δεν γνωρίζω Πάντως η χρονική στιγμή που γίνεται κάποια υποβάθμιση ή γίνονται κάποια σχόλια από οίκους αξιολόγησης ήταν ατυχής. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Πάντως ήταν ατυχής η στιγμή των σχολείων αν έγιναν πριν ή μετά κάποιες συναντήσεις Ευρωπαίων ηγετών κλπ. Οι επιστολές ε, που εκφράζουν τη γνωμοδότηση μπορεί να ε, να εκφράζονται με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται το σύστημα από ένα και μόνο στοιχείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φαντόρ. Καλό δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. στι δύο ερωτήσει που μου είχαν διατυπωθεί για την κοινή κλίμακα αξιολόγηση και για, μετά για την ε, υπηρεσία αυτή Δύο σχόλια. Η μεθοδολογία πέρα από τα διαθρωμένα προϊόντα δεν βασίζονται ουσιαστικά σε μαθηματικά πρότυπα. Είναι υποκειμενικού χαρακτήρα και να θυμόμαστε το θέμα των εκδοτών όσον αφορά την έκδοση μια ε, ολόκληρη επιτροπή αξιολόγηση. Ε, και είναι υποκειμενικές βασίε Έχουμε και τα θέματα μεθοδολογία ε, και εδώ το θέμα του μη εναρμονισμένου συστήματο προστίθεται. Οι μεθοδολογίε μπορεί να είναι αντιφατικές η μία έναντι τη άλλη. Και εδώ έχουμε το θέμα και της ανταγωνιστικής ε, συμπεριφοράς και στάσης. Ε, έχουμε και ε, τον υποχρετικό χαρακτήρα όσον αφορά ε, την απέτηση μιας υπηρεσίας τα προϊόντα αυτά να αξιολογούνται αποκλειστικά από αυτή την ίδια υπηρεσία. Ενδιαφέρον αυτό. Και βλέπουμε και το θέμα της ε, αναλογίας μεταξύ φερεγγιότητας όσον αφορά τις, τα διάφορα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Όλοι οι οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν αυτά τα ποσοστά και έχουμε εδώ και το πλαίσιο της Βασιλείας 3 και πολλές φορές αυτό ακριβώς ε, είναι ε, το σημείο αναφοράς ε και έχουμε μια μεθοδολογία που βασίζεται συγκυριακά υπό τα πρότυπα του αμερικανικού προτύπου ε, αξιολόγησης χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Και πρέπει εδώ να δούμε και τα θέματα των ε, ενυπόθηκων δανείων. Έχουμε και τις ε, επιδοτούμενες τράπεζες από πλευράς της Ευρώπης. Με αυτή τη βάση οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν χαμηλότερο ποσοστό κεφαλαιοποίησης και έχουμε εδώ και το πρόβλημα που τίθεται από αυτές τις αναλογίες. Θα πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα της ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ε, έχουμε και την ένταξή τους στην μεθοδολογία της στρατηγική από πλευρά των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτά να λυθούν υπόψη. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κράλ, έχετε τώρα δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. I will focus my answer on... Θα επικεντρώσω την απάντησή μου στις δύο ερωτήσεις και θα απαντήσω τα υπόλοιπα μερός. Μία ερώτηση. Πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα χρηματοδοτείται από τους επενδυτές ως πλατφόρμα. Δεύτερον, τι θα γίνει σε σχέση με την υπηρεσία αξιολόγησης όπως προτείνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αξιολόγησης που θέλουμε να δημιουργηθεί θα ε, καλύπτεται από ιδιωτικά κεφάλαια που θα συνεισφέρονται ιδιωτικά και θα είναι μη κερδοφόρο ίδρυμα. Εδώ σε σχέση και με το, την έννοια του δημόσιου αγαθού που μπορεί να ε, υποστεί πολύ αρνητικές ε, ή και αντίστοιχα και θετικές επιπτώσεις από μια αξιολόγηση. Το πρότυπο λειτουργία μια τέτοια ε, ε, υπηρεσία αξιολόγηση θα είναι τελείω διαφορετικό από τον τρόπο που λειτουργούν οι σημερινοί αξιολόγηση αξιολόγηση. Θα βασίζεται στο ε, πρότυπο Βασιλεία 2, συν επιπλέον μια υπηρεσία ε, για τις, ε, τα δάνεια και πιστώσει. Αυτό το σύστημα θα είναι από το σχεδιασμό του πιο διαφανέ. Θα μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα και θα είναι και πολύ φθηνότερο όσον αφορά τα κόστη που θα συνεπάγεται. Τρίτον, θα υπάρχει ένα υψηλό βαθμό διαφάνεια. Αυτό που ζητούμε να επιτευχθεί είναι η υπερδιαφάνεια. Ό,τι θα κάνει αυτή η υπηρεσία θα είναι προσπελάσιμο στο διαδίκτυο. Όποιος οποιοδήποτε θα μπορεί να ξέρει ε, τα στοιχεία λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας όπως ο κεντρικά υπεύθυνο ε, για την διαχείριση αυτού του οίκου. Θα γνωρίζουν όλοι με ποια βήματα, διαβήματα και μεθοδολογίες λειτουργεί αυτή η υπηρεσία θα δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο όχι μόνο τα αποτελέσματα αλλά και τα ενδιάμεσα διαβήματα για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Όλοι θα μπορούν στο διαδίκτυο να παρακολουθήσουν αυτές τις εργασίες. Δεύτερον, πόσα έχει αυτή η πλατφόρμα. Η πρότασή μας είναι πάγεται δύο τροποποιήσεις στην νομοθεσία. Κάθε εκδότης θα πρέπει όλα τα στοιχεία να τα δημοσιεύει σε αυτή την πλατφόρμα. Δεύτερον, όταν θα υπάρχουν ε, κάποιες ε, δράσεις ε, θα είναι η θα υπάρχει υποχρέωση είτε συμμόρφωση ε, είτε με την εφαρμογή των ίδιων των διατάξεων Βασιλεία 2. Αυτή είναι η πρότασή μας. Αφενό ε, θα μειώσει την ε, απουσία υπευθυνότητας ή λογοδεσίας και θα υπάρξει από την άλλη πλευρά ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και κατά τη διάρκεια δύο λεπτών τώρα η κυρία Λαουνή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη στι απαντήσει μου. Συμφωνούμε με την υπερβολική εξάρτηση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από τι αξιολογήσει και θα πρέπει οι αξιολογήσει να βασίζονται σε κανονισμού. Δεν σημαίνει ότι θα αντικαταστήσουμε τι αξιολογήσει με κάτι άλλο, γιατί οτιδήποτε και αν είναι αυτό με το οποίο θα τι υποκαταστήσουμε θα έχει κάποια... κάτι το μαγικό στο όνομά του. Αυτό που θέλουμε, θέλουμε να υπάρχουν διάφορε μορφέ αξιολόγηση και εξορισμού οι εταιρείε ε, να ασκούν τη δική τους δέουσα επιμέλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, δεύτερον, ε, η διαφάνεια γύρω από τις αξιολογήσεις είναι σημαντική. Δημοσιεύουμε τη μεθοδολογία μας, τα μοντέλα μας, τις αξιολογήσεις μας, το σκεπτικό και Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν όλοι να δουν πώς καταλήξαμε στο συμπέρασμά μας και να αποφασίσουν αν διαφωνούν μαζί, με εμά ή όχι. Είναι ελεύθεροι να διαφωνούν με τις απόψεις μας όσοι διαβάζουν τις εκθέσεις μας. Η διαφάνεια λοιπόν είναι ένα σημείο κλειδί. Από την πλευρά της Fitch ε, πρέπει να πούμε ότι δεν δίνουμε συμβουλές από τον κανονισμό. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να εξηγούμε ε, το σκεπτικό που μας οδήγησε στην αξιολόγηση. Για ποιο λόγο υποβαθμίσαμε ή δώσαμε υψηλότερο βαθμό σε κάποιον. Δεν έχει διαφορά αν είναι εταιρεία ή κράτος ή δημόσιο χρέος. Αυτά τα στοιχεία για μας είναι απαραίτητα. Το θέμα ε, της, ε, του ποσοστού αθέτησης, ε, πρέπει να πούμε ότι οι αξιολογήσεις δεν δίνουν πιθανότητα αθέτησης. Μέσω του χαρτοφυλακίου βλέπουμε την πιθανότητα αθέτησης και μπορεί να βγαίνει ένας αριθμός. Αν θα είναι μέσος όρος ή αν θα είναι ένας και μόνος αριθμός, ένα, μία θα είναι η επίπτωση. Εμείς προσπαθούμε να μην βασιζόμαστε σε μία πληροφορία και μόνο, αλλά να καταλαβαίνουμε καλύτερα όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις πληροφορίες για να μπορεί ο καθένας να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάουνη. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή και στον κύριο Ντομινίτσι. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στο πάνελ, κυρίως δε τους συναδέλφους που έδωσαν ιδέες, έκαναν προτάσεις. Να πω το εξής μονάχα. Η δουλειά που μας περιμένει, που έχουμε μπροστά μας, είναι δύσκολη και περίπλοκη. Ε, γιατί θα πρέπει να μεταφράσουμε τις ιδέες αυτές σε τροπολογίες στην πρόταση νέου κανονισμού που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό δεν θα είναι εύκολο. Ε, συζητούμε το θέμα αυτό γιατί οι οίκοι αξιολόγηση διάπραξαν πολλά σφάλματα. Ε, σήμερα όμως συζητούμε εδώ και γιατί ε, υπήρξε και αποτυχία της ισχύουσας νομοθεσίας, γιατί διαφορετικά ε, δεν είναι δυνατόν σε, ένα, σε αυτό το μικρό διάστημα μεταξύ ε, του πρώτου κανονισμού Σεπτέμβριο 2009 για τους οίκους αξιολόγησης ε, και το γεγονός ότι χρειάζεται πλέον αναθεώρηση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του σε ορισμένα στοιχεία. Πρώτον, αναθεώρηση των κανόνων. Εάν πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή της εξαίρεσης που αναφέρεται σε μεμονωμένες πρόνοιες, δηλαδή ή αν θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε μια γενικότερη γραμμή όπως στην Αμερικανική νομοθεσία που υπενθύμισε ο κ. Λάγκε. Δεύτερον, ε, για το, δημόσια, ε, για το δημόσιο χρέος θα πρέπει οι κανόνες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Τρίτον, θα πρέπει να σταματήσει το ολιγοπόλιο, να υπάρξει καλύτερος ανταγωνισμός. Εδώ έχουμε την πρόταση της εκπεριτροπής αξιολόγησης λειτουργεί αυτό και εναλλακτικέ προτάσεις. Ε, επόμενο σημείο. Δεν γίνεται λόγο στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή ε, ε, στον κανονισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτό το θέμα αυτό. Δεν θέλω να παρέμβω επί άλλων σημείων γιατί όπω είπαμε δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Εγώ υπενθυμίζω μονάχα ένα στοιχείο. Χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή νομική βάση για τι αποφάσει που λαμβάνουμε γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα στοιχεία τα οποία μπορεί να δυναμητήσει ε, όλο το σύστημα και επομένως να προκαλέσει κατάρρευση των ε, προτάσεων που κάνουμε. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με τη συνεργασία όλων ε, να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά για να αποδείξουμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί και πρέπει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομινίτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ την κυρία Ρώσ και ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές που εξέφρασαν τις απόψει τους. Ε, σας υπενθυμίζω ότι στις 28 ε, Φεβρουαρίου <clears throat> θα παρουσιάσει ε, η έκθεση και 22 Μαρτίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Παρακαλώ όσοι πρόκειται να αποχωρήσουν ε, να μας βοηθήσουν για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ βγείτε έξω όσοι θέλετε να έχετε συζητήσεις. This one? Is this one any better? Could those who are leaving please go? Παρακαλώ πολύ όσοι θέλουν να φύγουν να φύγουν. Δεν θέλω να γίνονται πηγαδάκια και συζητήσεις μέσα στην αίθουσα. Where's the rapporteur? I wish to give the floor to Otmar θα δώσω το λόγο άμεσα στον Ότμαρ Κάρα, στον εισηγητή. Yes, hello, Otmar. If you start... Ότμαρ, ίσω αν αρχίσει να μιλά, ενδεχομένω ε, θα δείξουν κάποια ευγένεια. Εάν δεν δείξουν την απαραίτητη ευγένεια, θα κατεβώ και θα σα πιάσω από τα αυτή να σα βγάλω από την αίθουσα. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν. Να μην παραμένουν στην αίθουσα. Ο Ότμαρ Κάρα θα παρουσιάσει την έκθεσή του όσοι συζητούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Λυπούμε, ήδη βρισκόμαστε 20 λεπτά πίσω από το χρονοδιάγραμμα, πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος Κάρας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πορεία από την συζήτηση και τους οίκους αξιολόγησης στη διαδικασία της Βασιλείας δεν ε, είναι μεγάλη η απόσταση αυτή. Σε κάποια ζητήματα άμεσα έχουμε και σύνδεση θεμάτων Βασιλείας 2 με τα όσα προσυζητήθηκαν. Ξεκινούμε με τη σημερινή παρουσίαση της έκθεσης και τονίζω από κοινού, από κοινού εξετάζουμε το νομοθετικό έργο το οποίο ξεκινάμε. Αυτό το νομοθετικό έργο έχει ε, θεμελιωθεί όπως σπάνια στο παρελθόν μέσω της κοινή προσπάθειας. Τον Οκτώβριο 2010 με την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας εμείς και το λέω συνειδητά, εμείς εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξ ονόματος αυτής της Επιτροπής θέσαμε τα θεμέλια για την πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής της Βασιλείας. Και τα θεμέλια τέθησαν επίσης ε, για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν αυτές οι δράσεις και τα θεμέλια. Και η πρόταση τώρα που έχουμε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την αξιολογούμε με αυτή την έκθεση κάνει ένα βήμα αποφασιστικής σημασίας προς την κατεύθυνση των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι εχθές και η, Προεδρία, η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου εχθές στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας η πρόταση ακριβώς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό αυτό το πνεύμα εξετάζεται και είναι μια αξιόλογη, μια αξιόπιστη βάση για τις εργασίες μας. Για μένα και επιτρέψτε μου να πω για εμάς όλους είναι αδιαμφισβήτητο ότι έτσι οι στόχοι της απόφασης αυτής οι στόχοι της, ε, των αποφάσεων της Λέσχης των 20 θέλουμε να επιτευχθούν και να εφαρμοστούν. Και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όχι μόνο επιθυμούμε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να το πράξουμε και αυτό θα πράξουμε. Πάντα είμαστε υπέρ ότι όταν ερχόταν, θα ερχόταν η ώρα της υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ενδοευρωπαϊκά ιδιόμορφα στοιχεία όσον αφορά την οικονομική δομή, τη χρηματοδότηση της ίδιας οικονομίας και το αποκεντρωμένο, το αποκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα που πολυσχηδώς πρέπει να λειτουργεί, όλες αυτές οι διομορφίες στην ενδοευρωπαϊκή εφαρμογή τους πρέπει όλες αυτές οι πτυχές να επιτεθούν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θέλουμε να λαμβάνετε υπόψη και έτσι να δρούμε. Από τις, ε, την έγκριση της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας ε, υπήρξαν εξελίξεις ε, που το πλαίσιο επιπλέον το διευρύνουν σε σχέση με τις δικές μας προτάσεις. προτάσεις. Αφενός έχουμε και την ε, απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για το 9% επανακεφαλοποίηση. Το αναφέρω αυτό επειδή αυτό ως ποσοστό είχαμε αναφέρει εμείς και πολλές τράπεζες, όχι όμως όλες οι τράπεζες, μόνο οι τράπεζες που υπέστησαν δοκιμασία, τα τεστ μέχρι την 30 Ιουνίου 2012 πρέπει να έχουν επιτύχει και να έχουν πάρει πιστοποιητικό. 9% όχι για όλες λοιπόν τις τράπεζες αλλά για κάποιες από αυτές και 9% με διαφορετική γενικούς ε, ορισμούς και προσδιορισμούς ιδίου κεφαλαίου όσον αφορά τις διεργασίες της ε, Συμφωνίας της Βασιλείας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεύτερον, έχουμε κάποια κράτη-μέλη και αναφέρω τη Σουηδία και την Αυστρία που την επισπεσμένη εφαρμογή της φάσης Βασιλείας 3 από την 1η 2013 άσχετα από τις μεταβατικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν έχουν ήδη αποφασίσει. Τρίτον, σε αντίθεση με όλα αυτά έχουμε πρώιμη εφαρμογή ή επισπεσμένη εφαρμογή του 9% ή και όσον αφορά την ίδια την εφαρμογή των διεργασιών της Συμφωνίας Βασιλείας. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, έχουμε μια αντίστοιχη ε, ε, εξέλιξη όπου ούτε ε, τα θέματα βασιλείας ούτε τα CRI 3 ούτε και η βασιλεία 2 επαρκώς εφαρμόζονται αυτή τη χρονική στιγμή ως παράλληλη έκβαση. Παρότι έχουμε την, τα διεθνή θεμέλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για κάτι τέτοιο, τα οποία έχουν ήδη τεθεί. Αυτές οι διαφορετικές συνθήκες πλαίσιο λοιπόν που ισχύουν έχουν και διαφορετική νομική βάση που δημιουργούν. Έχουν μια διαφορετική, αν θέλετε, προσέγγιση των ιδίων κεφαλαίων. Αλλά αν εμείς πολιτικά δεν καταλήξουμε σε μια αλληλουχία και αλληλεξάρτηση αυτών των θεμάτων, θα έχουμε συσσόρευση μεν αθρηστικά υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που θα έχουν επιπτώσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση και της ανάπτυξης και των επενδύσεων και της ε, ε, ανάπτυξης ε, που θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι στη διεργασία της Βασιλείας εμείς νομοθετικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε επανορθώσεις ή διορθωτικές κινήσεις. Όμως έχουμε την υποχρέωση να λάβουμε υπόψη το πολιτικό πλαίσιο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Και έτσι η έκθεσή μου όχι μόνο τροπολογίες και τροποποιήσεις εμπεριέχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχει επίσης ε, και κάποιες, ε, κάποια αιτήματα ή απαιτήσει έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτή τη διεργασία και εξέταση και τροπολογιών, ώστε κάποια θέματα να αποσαφινιστούν, ώστε μέσα στο πλαίσιο τη της προθεσμίας τροπολογιών να μπορέσουν να εξεταστούν. Παράδειγμα, στρέβλωση ανταγωνισμού έναντι των ΗΠΑ, αλληλουχία σε σχέση με το 9% για τις τράπεζες. Όλα αυτά ζητούν απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εμείς εδώ λοιπόν προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη και αξιολογήσεις που πρέπει να γίνουν και να ληφθούν επίσης υπόψη σε σχέση με τα κράτη-μέλη κάποιες δράσεις που αν δεν έχουν συντονιστεί οι βλάβες, οι ζημιές στο τραπεζικό τομέα ή σε σχέση με άλλες ε, ε, χώρες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε 27 διαφορετικές ρυθμίσεις που αποδυναμώνουν ένα συνολικό πλαίσιο, ενιαίο πλαίσιο και οδηγούν σε στρεβλώσεις και εντάσεις. Και σε αυτό προβλέπει η έκθεση και στοχεύει σε μία ε, εναρμόνιση και μεγιστοποίηση, όχι ελαχιστοποίηση, αλλά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εναρμονισμό και συντονισμό. Και τελευταία παρατήρηση. Έχουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι, όπου βραχυπρόθεσμες ε, κινήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα υψηλότατο επίπεδο όπως ποτέ στο παρελθόν παρατηρούνται η εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών ε, ακόμα δεν είναι δεδομένη. Και λέγω ότι ο στόχος πρέπει να ληφθεί υπόψη ενωμένο το Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν στην οικονομία και θα απελευθερωθούν προς όφελος της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Αυτές τις συνθήκες πλαίσιου έχω λάβει υπόψη και προτείνω σε σχέση με την έκθεσή μου. Δεν είναι όμως η τελική έκθεση αυτή με αυτόν τον τρόπο. Προσπάθησα από τις διάφορες συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο να καταλήξω σε θεμέλια, σε μια βάση για την κοινοβουλευτική μας εργασία, για το κοινοβουλευτικό μας έργο και να αναφερθώ στα κυριότερα ζητήματα και από κοινού μαζί με εσάς τώρα να καταλήξουμε στη διατύπωση τροπολογιών που θα δώσουν τη δυνατότητα μέχρι την τελική έγκριση, ψήφιση και έγκριση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή που προβλέπεται για τον Απρίλιο, να καταλήξουμε σε μια κοινή έγκριση αυτών των προτάσεων όπως ε, ως ήθιστε, ώστε να καταλήξουμε σε ε, κοινέ αποφάσεις. Όμως αυτή η έκθεση είναι ένα σαφές μήνυμα προς ποια κατεύθυνση θέλουμε με συνέπεια να κινηθούμε ώστε να εγκριθεί αυτό το εγχείρημα. Χαίρομαι ότι το Συμβούλιο, το Συμβούλιο μέχρι στιγμής ε, ε, προβλέπει αυτή την κοινή θέση και την πρόθεσή του, ώστε μετά την συνεδρίαση και λήψη απόφασης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εμπλακεί πλήρως σε αυτές τις διεργασίες. διεργασίες. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των διαβουλεύσεων στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή τώρα, από τώρα μέχρι τον Απρίλιο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την δυνατότητα παραλληλισμού των ε, ε, προτάσεων των δικών μας ώστε να καταλήξουμε στο ρυθμιστικό πλαίσιο που παράλληλα θα πρέπει να μπορέσει να αναπτυχθεί, ώστε να μην είναι το ένα σκέλος κατά του άλλου. Κατά του άλλου. Εμείς είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι και δεν απεμπολούμε ως Ευρωκοινοβούλιο ε, για λόγους ε, ε, που ίσως θα μπορούσαν να εξυπηρετούν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν απεμπολούμε αυτό το δικαίωμα. Το πρώτο θέμα όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιο είναι. Είναι το ότι απορρέουν όλα αυτά από την συζήτηση σε σχέση με τα όσα ε, εξετάζουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τον, τη ρήτρα των 9%. Θα ήθελα επ' να πω ότι η αύξηση του ιδίου κεφαλαίου των τραπεζών θα πρέπει το δυνατόν ταχύτερα να επιτευχθεί, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν τα πλήγματα ή τις διακυμάνσεις να τις αντιμετωπίσουν ή να τα αντιμετωπίσουν έγκαιρα. Δηλαδή, μεταξύ του 2013 ή 2014, μεταξύ του 3,4 και του 5,4% του κεφαλαίου που θα πρέπει να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ προτείνω από την 1η του 2013 ήδη 4,5% του ε, ιδίου κεφαλαίου να αυξηθεί σε 6% ώστε να έχουμε την διασφάλιση αυτού του ποσοστού ως κεφαλαίου, ώστε να έχουμε την αντιμετώπιση του ζητήματος της ελαστικότητας. Γιατί διαφορετικά θα είχαμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις που δεν θα συνεισέφεραν στην ε, αποσαφήνιση των πραγμάτων η υψηλότερη δηλαδή ε, το υψηλότερο ποσοστό και όχι το χαμηλότερο που θα έπρεπε να ισχύσει κατά αυτή τη χρονική στιγμή. Δεύτερον, η άρση των ανισορροπιών όσον αφορά τα ε, δάνεια και τις πιστώσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το τονίζω αυτό. Πάντα από κοινού συζητείται αυτό το θέμα και, στο, και στους πολίτες μας σε σχέση με το ESFS ή το, ε, ε, τις διάφορες άλλες ρυθμίσεις ε, παρόλα αυτά όμως ε, και καταλήγουμε σε αυτή την κατάσταση έχουμε μέτρα με διαφορετικές επιπτώσεις εκάστοτε. Πρέπει όμως να εξισορροπήσουμε τα πράγματα, να σταθεί η ισορροπία, να πούμε τι θα γίνει με την μηδενική αυτή δράση ή τοποθέτηση σε σχέση με την κρίση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και τις επιπτώσεις της. Πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Γι' αυτό έχουμε το κυριότερο αίτημα χωρίς ε, να έχουμε εδώ την ε, πρόθεση να αγνοηθούν τα θέματα του δημοσίου, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι, είναι μια σαφής τοποθέτηση αυτή από πλευρά μας ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα. Εδώ από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια δηλαδή της προθεσμίας εξέτασης των τροπολογιών να μας δώσει την αξιολόγηση της ομάδας εργασίας και των προτάσεων του Συμβουλίου. Τρίτη, ε, τρίτος τομέας είναι οι διατάξεις για την ρευστότητα. Πιθανότατα είναι το πιο σημαντικό τμήμα των νέων ρυθμίσεων, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε ε, κυριότατα ένα θέμα ρευστότητας ε, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Δηλαδή, είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε προτάσεις της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει όμως να επανεξεταστούν σε σχέση με τη ρευστότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει επαρκώς καθοριστεί, δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς. Ποιες επιπτώσεις ε, εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Για παράδειγμα το θέμα του χρυσού, των ε, δανείων, όπου σε σχέση με την ρευστότητα μπορεί να επηρεάζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ασάφεια και θέλουμε να υπάρχει μια δράση παράλληλα προς τις ε, προτάσεις για, την, ε, για τις τράπεζες και τη Βασιλεία ώστε μέχρι το 2015 να είναι δεσμευτικές και αυτές οι προσεγγίσεις. Χρειάζονται λοιπόν σαφέστεροι ορισμοί. Τέταρτο σημείο, αναλογία leverage, μοχλική αναλογία. Εδώ χρειάζεται αξιολόγηση των πραγμάτων. Αν θα μπορούσε νωρίτερα να δημοσιευθεί αυτή, τότε δεν θα ήταν πλέον ε, χωρίς επιπτώσεις. Μια και υπάρχει μεγάλη πίεση των αγορών. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι οι σημερινές διατυπώσεις ε, όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργούν ασάφειες Μία σημαντική ασάφεια είναι εκείνη που στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορούμε να άρουμε εμείς. Δηλαδή, διεθνώς να δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι χαρακτηρισμού ή ε, αναφοράς ε, με, ε, στην, ε, στις διεθνείς δράσεις. Πρέπει όμως να υπάρχει συγκρισιμότητα των ψηφίων ή των τρόπων αξιολόγησης. Τέταρτο σημείο, ΕΠΑ. Ξέρουμε ότι έχουμε 170 διασταυρούμενες αναφορές. Όλοι νομίζω έχουμε το στόχο, κοινό στόχο να μειώσουμε αυτές τις πολυάριθμες αναφορές. Στη σημερινή πρόταση έχουμε τρία σημεία. Πρώτον, ένα πίνακα προτεραιότητας για αυτέ τι διαφορετικέ αναφορέ με 12 συγκεκριμένε προτεραιότητε να ξεκινήσει το έργο τη ΕΠΑ παράλληλα με το έργο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. και πρέπει να διεξαχθεί διάλογο μεταξύ μα. Δεύτερον, μία διαγραφή 10 διασταυρούμενων διαφορετικών αναφορών. Έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα με την ΕΠΑ και 17 σημεία με αναβολή όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, με χρονική αναβολή. Έχουμε ένα πακέτο λοιπόν 40 συνολικά τέτοιων ε, προτάσεων που διαφοροποιούμε το τι πρέπει να γίνει και αυτό θα ήθελα να σας το αναφέρω να το λάβετε υπόψη. Το επόμενο σημείο είναι στην οδηγία έχουμε την corporate governance ε, όσον αφορά τον τίτλο και τις δυνατότητες ε, των δυνατοτήτων παρέμβασης. Σε σχέση με τα κράτη-μέλη υπάρχει μια σχετική, τροποποι... μια σχετική προσαρμογή. Έβδομο σημείο. Ο υπολογισμός ε, των ε, μη κυκλικών ή κυκλικών και μη κυκλικών δράσεων είναι αυτή τη στιγμή εξατομικευμένος. Χρειαζόμαστε όμως μια κοινή βάση για όλους για αυτή τη διαμόρφωση αυτού του περιθωρίου. Θα πρέπει λοιπόν ε, εδώ να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή βάση των αντικυκλικών αυτών ε, ε, χαρακτηριστικών που θα λαμβάνονται υπόψη από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Τε, τελευταίο σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ έχουμε δύο αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια τμήματα από όλα αυτά δεν μπορούν όπως θεωρούμε εμείς αν οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν συμμορφωθούν ταυτόχρονα και δεν υλοποιήσουν ταυτόχρονα αυτές τις προτάσεις. Διότι διαφορετικά θα καταλήξουμε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά. Παρακαλώ λοιπόν <clears throat> οι διαφορετικές αυτές, ε, οι διαφορές αυτές ε, μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ να μην χρησιμοποιηθούν ως ένασμα ή ε, άλοθη για να πούμε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εμείς η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να αναλάβει και να προχωρήσει με το νομοθετικό έργο. Κατά τη διάρκεια όμως αυτών των ε, διεργασιών να ξέρουμε ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν για την Ευρώπη αν θα υπάρξει άνισο ή διαφορετικό χρονικό διάστημα εφαρμογής αυτών και οι ΙΠΑ δεν τηρήσουν τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις τους θα πρέπει έτσι πολιτικά να αξιολογηθούν αυτά τα θέματα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Το τελευταίο σημείο είναι μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων ρυθμίσεων όσον αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το δυνατόν ταχύτερα πρέπει να διευθετηθεί αυτό, διότι αφενός πρέπει να συμφωνήσουμε στους κανόνες και κανονισμούς και να συναγάγουμε τα συμπεράσματα από την κρίση. Όμως να μην παρακολήσουμε την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης <clears throat> Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτών των ε, υποχρεωτικών σημείων αναφοράς ε, συνέταξα την έκθεσή μου εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Προσβλέπω στην ενδιαφέρουσα συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Καθένας από εμά ζητείτε να συμμετάσχει, όχι μόνο η συγητή. Σας ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές για την ομάδα των σοσιαλιστών. Ούντο Μπούλμαν. Ο κύριος Ούντο Μπούλμαν, ευχαριστώ Σάραν, ευχαριστώ τον Ότμαρ Κάρας για την κατάθεση, την παρουσίαση αυτών των προτάσεων και την κίνηση της συζήτησης. Εμείς στη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή ότι σε τέτοια περίοδο κρίσης η καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά βοηθά περισσότερο και όχι η αναμονή ή η αναβολή. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή ε, συνεργασία και κοινό έργο. Έχει δίκιο ο εισηγητή όταν λέει ότι όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε και να εμπλακούμε. Εδώ έχουμε ένα στοιχείο πυρήνα της νομοθεσία που βρίσκεται επί τραπέζης ε, και πρέπει να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν η συζήτηση από πλευρά τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα έχει πάρει την εξή τροπή. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια από τι μεγάλε ευκαιρίε εδώ μπροστά μα. ώστε η αναγκαία αναδιάρθρωση και προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος να επιτευχθεί και να επηρεάσουμε τα πράγματα σε σημαντικό βαθμό με αυτόν τον τρόπο. Να μην χάσουμε την ευκαιρία για την αναπροσαρμογή αν θέλουμε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση και να εξέλθει νικήτρια. Έτσι λοιπόν με φιλόδοξους αυτούς στόχους πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να επινοήσουμε τον τροχό εκ νέου βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στην προσαρμογή και αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είναι το benchmark αυτή είναι η πρόκληση όταν θέλουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να δραχτώ της ευκαιρίας και κάποια σημεία να αναφέρω, όχι όλα βέβαια, διότι ο εισηγητής έχει και το δικαίωμα με μια τέτοια ευκαιρία να γνωρίζει προς ποια κατεύθυνση επιθυμούν οι σκιώδεις εισηγητές να πορευθούν, προς ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να μεταξελιχθεί η συζήτηση από πλευρά των εμπλεκόμενων κοινοβουλευτικών ομάδων όσο αφορά το νομοθετικό έργο. Καταρχήν πρώτα, ποια είναι η γενική ρήτρα, ποιο είναι το γενικότερο σκεπτικό είναι το ότι το σύστημα πρέπει να μειώσει τους κινδύνους πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των κινδύνων. Δεν επιτρέπεται να ξανακαταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίζουν ανεξέλεγκτους ε, κινδύνους ε, από πλευρά του χρηματοοικονομικού συστήματος και από τις τράπεζες που στο παρελθόν οδήγησε στην κατάρρευση και δεν θα είναι δυνατό να υποστούμε μια νέα τέτοια κατάσταση έκθεση σε τέτοιους κινδύνους. Αυτό πρέπει να μας κάνει να ξεχωρίζουμε μεταξύ φορεί κινδύνων και επικίνδυνων επισφαλών προϊόντων και πρέπει να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την πτυχή των δανείων, ιδιαίτερα για εκείνους που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ιδιαίτερα στον, τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν λοιπόν προτείνει ο εισηγητής εδώ να προσέξουμε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρξει σωστή στάθμιση κινδύνων, έχει δίκιο και θα βοηθήσουμε και θα προχωρήσουμε και εμείς με συγκεκριμένες προτάσεις που θα υποβάλουμε για να βοηθήσουμε για να δούμε πού βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος και πού βρίσκονται οι καθημερινοί κίνδυνοι της καθημερινής εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε δυσανάλογη ε, επιβάρυνση που να οδηγήσει στο να μην μπορούν να επενδύσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όταν εμείς λοιπόν θέλουμε τη δομή των κινδύνων να την αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε θέματα ρευστότητας, τότε δεν έχουμε ακόμα πιστεί ότι όλα τα προβλήματα με την liquidity coverage ratio, με την αναλογία κάλυψης ρευστότητας μπορούν να επιληθούν. Πολύ περισσότερο πρέπει να δούμε και την αντιμετώπιση επισφαλιών και κινδύνων. Μακροπρόθεσμα δηλαδή θέματα που αφορούν την δομή, την διάρθρωση της ρευστότητας και μπορούν να την επηρεάσουν. Θα θέλαμε λοιπόν έτσι με τον ίδιο τον εισήγητη να καταλήξουμε σε διαβουλεύσεις, σε συζητήσεις για να δούμε αν το net funding ratios θα μπορούσε να είναι ένα μέσο με το οποίο θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε ή να ε, μειώσουμε τους κινδύνους συστημικά από το ίδιο το σύστημα και μια βραχυπρόθεσμη, ένας βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός να μετατραπεί σε ένα πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τραπεζικά. Αν θυμηθούμε τι έγινε με το ε, προηγούμενο των Lehman Brothers, πρέπει να δούμε ότι διαδραμάτισε ένα ρόλο η βραχυπρό, ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός και αντιμετώπιση των προβλημάτων και είχαμε την κατάρρευση. Ας δούμε λοιπόν την άλλη προοπτική. Μήπως υπάρχουν λειτουργικά κάποια πρότυπα και πρότυπα σχεδιασμού όπου μπορούμε να καταλήξουμε σε μεγαλύτερη ασφάλεια στο σχεδιασμό μας. Επόμενο σημείο είναι το ζήτημα πώς να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν από το θέμα των sovereign bond. Εδώ έχουμε το ζήτημα, όπως λέει ο εισηγητής, ότι πρέπει να υποβάλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρυθμιστεί αυτός ο τομέας. Και εμείς συμφωνούμε. Θα θέλαμε όμως να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, πιο μακριά έχουμε κινδύνους σε σχέση με την διαχείριση αυτού του κινδύνου. Έχουμε κάποια βήματα αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων και ακριβώς έχουμε και την απήχηση των όσων ακούσαμε σήμερα το πρωί. Δηλαδή πώς θέλουμε να τροποποιηθούν οι δράσεις των ε, οίκων αξιολόγησης και να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτήν την επιρροή που ασκούν και να δούμε τι μπορεί να γίνει ώστε να μην υπάρχουν ρήτρε και διατάξεις που δεν είναι απόλυτα αναγκαίες. Αν το θέλουμε όμως αυτό, υπάρχει μια διασύνδεση της έκθεσης ε, του Λεωνάρντο Ντομένιτσι, της έκθεσης του κυρίου Ότμαρ Κάρας ε, και των προτάσεων για τους οίκους αξιολόγησης και πρέπει αυτά να συμπτυχθούν και να γίνουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει αξιοπιστία γιατί λοιπόν εδώ δεν προσεγγίζουμε αυτό το σημείο με τον ίδιο τρόπο και γιατί δεν απαιτούμε από το τραπεζικό σύστημα να δημιουργηθούν δομές τέτοιες με τις οποίες θα μπορούμε καλύτερα να λειτουργήσουμε και να εργαστούμε στο τέλος χωρίς διαρκώς να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες τις κατηγορίες και τα παράπονα για τους οίκους αξιολόγησης. Ένα βήμα προς τα εμπρός δηλαδή θα ήταν ευκταίο. Αυτό θα θέλαμε να το συζητήσουμε λοιπόν με τον εισηγητή το ζήτημα το οποίο ε, ανέφερε ο Ότμα Κάρανς, Κάρας, να υπάρξει ένας ανταγωνισμός, ε, η ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ του καθεστώτος ε, Βασιλείας 3 και του καθεστώτος ΕΠΑ. Πώς θα πρέπει δηλαδή όλα αυτά τα θέματα να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο όσον αφορά και τις απαιτήσει κεφαλαίου. Θα πρέπει εδώ συμβατότητα να ε, εμπνέει το έργο μας ρυθμιστικά και να ξέρει ο τραπεζικός τομέας ότι υπάρχει μακροπρόθεσμα ένα αξιόπιστο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να βασίζεται. Τι θα κάνουμε, μακροπρόθεσμα θα το σχεδιάσουμε ώστε να υπάρχει αξιοπιστία και να υπάρχει η ασφάλεια, η νομική και η βεβαιότητα. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον ως νομοθέτες να έχουμε διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς και μακροπρόθεσμα να μην μπορούν να υπολογιστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια Θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα εδώ είναι ένα θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε να απασχολούμεθα με την έκθεση της συναδέφου Αρλίν Μακάρθη. Corporate Governance, ένα από τα κύρια σημεία επικέντρωσης, εξέτασης στην ε, προηγούμενη αυτή έκθεση. Νομίζω ότι κάποια θέματα ακόμα εκκρεμούν. Εκκρεμούν κάποια θέματα. Πώς ε, η συμπεριφορά στη διαχείριση θα λαμβάνει περισσότερο μακροπρόθεσμους στόχους υπόψη. Τότε στο παρελθόν κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, ό,τι καλύτερο δεν καταλήξαμε σε όλα τα θέματα στην βέλτιστη ρύθμιση. Θα θέλαμε να ξαναξεκινήσουμε τώρα με τον συνάδελφο, τους συναδέλφους του ΕΛΚ και με τους ε, συναδέλφους των φιλελευθέρων να ξανασυζητήσουμε και να δούμε με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά το τελευταίο διάστημα για το ζήτημα της corporate governance αν θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε ένα πακέτο μέτρων που θα να προτείνουμε ένα πακέτο μέτρων που θα εγκρινόταν ώστε να είμαστε μακροπρόθεσμα προετοιμασμένοι για τέτοιες προκλήσεις και να αντιμετωπίσουμε προς όφελος των επενδυτών και των καταναλωτών τέτοιες προκλήσεις. Αυτά ουσιαστικά είναι σε αδρές γραμμές τα ουσιοδέστερα σημεία με τα οποία πρέπει να απασχοληθούμε. Είμαστε σίγουρα, σίγουροι ότι βρίσκεται σε καλά χέρια αυτή η έκθεση και χαιρόμαστε για τη μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώ σα προειδοποιώ ότι ήδη έχουμε 11 ονόματα στον κατάλογο αγορητών, 12 τώρα με την Αλήν. Αν δεν τα καταφέρουμε να τελειώσουμε σήμερα, θα πρέπει να βρούμε κάποια άλλη χρονική στιγμή να το συζητήσουμε. Θα μιλήσω εγώ στη συνέχεια ως σκιώδης εισηγήτρια από την άλλη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι έλαβε υπόψη του πολλά από τα σημεία τα οποία συζητήσαμε στην ανταλλαγή απόψεων και στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Δεν ε, ε, είναι εύκολο να αναφέρω όλα τα σημεία στα οποία ε, συμφωνώ ή διαφωνώ. Μόνο λίγε παρατηρήσει θα κάνω. Καταρχήν θέλω να πω όπως θα περιμένετε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό ε, το ότι προσπαθεί να επιτύχει αυτή η μηδενική ρυθμίση για το δημόσιο χρέος. θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι ε, δυσανάλογο το ποσοστό διατήρησης ε, στοιχείων μηδενικού κινδύνου να μην δημιουργηθούν φιλοκυκλικά φαινόμενα αν προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή πολύ γρήγορα ή χωρίς να το έχουμε σκεφτεί επαρκώς. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από τους κανόνες που θα έχουμε για το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, θα πρέπει κατά παρόμοιο τρόπο να υπάρχουν κανόνες και για τις τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες ε, αντιπροσωπεύουν λιγότερο ονομαστικό δημόσιο κίνδυνο, ε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα όταν μια χώρα ε, ζητήσει κάτι θα πρέπει να γίνει κατόπιν αιτήματος Και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με την τροπολογία ε, για ε, το trade finance. Εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι επιζητούμε επενδύσεις και ανάπτυξη, δεδομένης της κρίσης δημοσίου χρέους στην οποία βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε δημοσιονομική ισορροπία μέσω της λιτότητας. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητά μας. Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι σημαίνει το trade finance. Θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη διατύπωση με πραγματικό ορισμό. Όπως και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το trade finance δεν είναι ένα τομέα όπου θα πρέπει να πειραματιστούμε με το υψηλότερο κεφάλαιο και μετά να επανέλθουμε και να κάνουμε μία ε, ανασκόπηση για να δούμε αν ε, επιφέραμε κάποια ζημία με αυτά τα οποία θεσπίσαμε. Διότι οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες ενδέχεται να υποστούν ζημίες αν εμείς είμαστε πάρα πολύ βιαστικοί. Και σίγουρα στις παρούσες οικονομικές συνθήκες δεν πρέπει να ρισκάρουμε το να δημιουργήσουμε ζημίες. Ε, κάποια στοιχεία για την αναλογικότητα έχετε συμπεριλάβει όπως έχουμε συζητήσει. Μιλήσατε και για τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και υπάρχουν πολλές τέτοιες ε, ιδιαιτερότητες όπως είπε και ο Μάριο Ντράγκη την περασμένη εβδομάδα ως ε, πρόεδρος του ESRB. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μία κοινή λύση για τα πάντα. Είπαμε ότι θα, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη εναρμόνιση από τη μία πλευρά και των πολλών διαφορών από την άλλη πλευρά όταν έχουμε τις ευρωπαϊκές συστημικές ε, ε, τράπεζες και ό,τι υπάρχει από την άλλη πλευρά. Προσπαθούμε να τα επιλύσουμε όλα αυτά, διότι αντί να ασχοληθούμε για το τι γίνεται σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, θα πρέπει να έχουμε διατάξεις που θα εφαρμόζονται κατά οριζόντιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Για τις συστημικές τράπεζες όμως έχω την γενική εντύπωση ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα κριτήρια της Βασιλείας αρκετά στενά, με τη ρήτρα που αναφέρεται σε σχέση στις Ηνωμένες Πολιτείες. κάποια απόκληση από τη Βασιλεία δεν θα είναι ασυνεπής σε διεθνέ επίπεδο, γιατί δεν εφαρμόζουν άλλες χώρες τα κριτήρια της Βασιλείας στα ίδια σημεία. Και θα πρέπει ε, να αποδεχθούμε το ότι ίσως δεν μπορούμε να φτάσουμε το σημείο της μέγιστης εναρμόνισης, αλλά σε ορισμένους τομείς χάρη της αναλογικότητας πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τις Ηνωμένε Πολιτείε και σε αυτό το θέμα και σε άλλα θέματα θα ήθελα ε, να μην πάνε γυμνή στη μάχη οι δικοί μας διαπραγματευτές. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι σκόπιμο να περιμένουμε αμερικανική νομοθεσία. Πρέπει κάποιο άλλο τρόπο να βρούμε ε, για να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Πάντως ε, καταλαβαίνω αυτό που επιθυμεί ο εισηγητής ε, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε ίσως με κάποια άλλη έκθεση στη συνέχεια. Είπαμε ότι μπορούν να εφαρμόζονται οι διατάξει ε, ε, σε κάποια ομάδα τραπεζών, όπως υπάρχει και στην οδηγία. Ε, λέτε επίσης, στην τροπολογία 2 νομίζω, ότι θα πρέπει να ισχύει ενιαίο σύστημα κανόνων σε όλους του συμμετέχοντες στην αγορά. Σύμφωνα με αυτό το οποίο λέτε και για την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να εννοούμε συγκρίσιμους παράγοντες της αγοράς ε, αν κάνετε κάτι για μια ε, τράπεζα αποταμιευτική, δεν είναι το ίδιο αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για μια πολυεθνική συστημική τράπεζα. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες. Χρειάζεται λοιπόν ένα μείγμα επιπέδων και να χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, και την ESRB με προσαρμοσμένο τρόπο, να μην ξεχνάμε δηλαδή τις εξουσίες που έχουμε δώσει σε αυτούς τους οργανισμούς και ως προς αυτό συμφωνώ ότι πρέπει τις δεσμευτικές εξουσίες μεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να τις επεκτείνουμε και σε άλλα σημεία. Αυτό είναι ένα οριζόντιο θέμα για την Επιτροπή μας. Εν γέννη συμφωνούμε με το άρθρο 19β και με την δεσμευτική μεσολάβηση που αναφέρεται εκεί και θα θέλαμε να χρησιμοποιείτε περισσότερο και όχι λιγότερο. Υπάρχει λίγο θόρυβο στην αίθουσα, αλλά συνεχίζω. Στην τροπολογία H προτείνεται ότι άλλοι συστημικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, με προληπτική εποπτεία που μπορεί μακροοικονομικά να αναπτυχθεί Πράγμα το οποίο και συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε ένα, κείμενο, ένα κείμενο που να μας δίνει περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά την ESRB. Ε Προς το παρόν, ο ρόλος που τους ε, έχουμε δώσει ε, δεν ε, πληρεί, δεν φτάνει στο επίπεδο των άρθρων 16 και 17 τους αποδίδουμε ένα ρόλο συμβουλευτικό για την ομοθέσια και έχουν και κάποιο ρόλο συμβουλευτικό στο πλαίσιο των μεμονωμένων κρατών μελών. Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε κάθε φούσκα κινήτων που μπορεί να προκύψει και ένας από τους λόγους που υπάρχει η SRB είναι ακριβώς ε, να αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα και όπως γνωρίζετε στο παρελθόν τα κίνητα στην Ισπανία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάστηκε να τα βάλουμε στο στόχο μας, πράγμα το οποίο δεν χρειάστηκε στη Γαλλία και προειδοποιήσεις από την ESRB θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να το αντιμετωπίσουμε αυτό μπορεί να μην πρόκειται για εναρμόνιση, αλλά μπορεί να, πει σε κάποιο, να μπορούν να πούν σε κάποιο κράτο μέλο ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτή τη φούσκα κινήτων διότι δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία σα. Υπάρχει δηλαδή ε, μια εναρμόνιση, διότι υπάρχει καθοδήγηση από μια ευρωπαϊκή πηγή, από το ESRB, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Δεν γίνεται με βάση 27 διαφορετικούς κανόνες των κρατών μελών αυτό το οποίο προτείνει η SRB δεν θα είναι ε, πάντοτε ακριβώ το ίδιο για κάθε κράτο μέλο. Θα πρέπει να το ακολουθούν όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την, ε, τον κανονισμό ΕΜΗΡ ε, υπάρχουν περισσότερα τα οποία πρέπει να γίνουν και ιδιαίτερα για τα συνταξιδοτικά ταμεία και για τα εταιρικά κεφάλαια. Νομίζω ότι είμαστε στο πλαίσιο των CDA. Το θέμα ε, της διαφάνειας ε, είναι το επόμενο που θα ήθελα να αναφέρουμε. Σε πολλούς τομείς θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερο για το τι συμβαίνει στον ε, τραπεζικό τομέα και στις συναλλαγές γενικότερα. Ίσως υπάρχουν υποχρεώσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε και οι οποίες ισορεύονται. Παραδείγματο χάρη θα πρέπει να υπάρχει κάποια δήλωση των συμφωνιών επαναγοράς μεταξύ τραπεζών όταν υπάρχουν ε, στοιχεία ενεργητικού στα οποία είναι αντικείμενα ανταλλαγών μεταξύ τραπεζών, ε, ε, θα πρέπει να το γνωρίζουμε, θα πρέπει κάπου να καταγράφεται. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε πλήρη εικόνα των όσων γίνονται. Καλύτερα θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτά τα οποία ε, είναι αντικείμενο συναλλαγών και στις συναλλαγές ε, ε, παραγόγων θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρήτρα. Αυτό ήταν και το πρόβλημα με την Lehman Brothers. Κάποια στοιχεία ενεργητικού που νομίζαμε ότι τα έχει μια τράπεζα, ξαφνικά βρίσκονταν στα πλαίσια ενός clawback σε μια διαφορετική κατάσταση. Και τελικά ο καταθέτης ή ο ασφαλιστικός φορέας του καταθέτη θα φέρει το βάρος. Εάν υπάρχει κάποια ρήτρα clawback και δεν είναι καταγεγραμμένο, δεν θα πρέπει να έχει και νομικές επιπτώσεις. Αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη νομική, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ε, ε, σύστημα του σκιώδους τραπεζικού τομέα. Τέλος, σχετικά με τα ε, ε, ρέπος ήδη ε, μίλησα, αλλά και για διαφορετικά προϊόντα, θα πρέπει να βρούμε μία μορφή δημοσιοποίησης που θα δείχνει τι ποσοστό, τι ποσοστό κεφαλαίου καλύπτει τις καταθέσεις. Όταν έχουμε ομόλογα ή άλλες ή άλλα προϊόντα μερικές φορές ε, ε, τίθεται σε ένα κατάλογο προτεραιότητας διαφορετικό από αυτό που θα είχαν επιλέξει οι καταθέτες. Άλλα ε, στοιχεία της δημοσιοποίησης χρειάζονται και για την εποπτεία και γενικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει κάποιο επίπεδο δημοσιοποίησης πιστοποίησης ε, που να καλύπτει τις ανάγκες των καταθετών. Δεν θέλω να καταχραστώ όμως το χρόνο και δίνω το λόγο στην επόμενη σκιώδη εισηγητήρια που είναι η Βίκη Φόρντ. Λέω τον κατάλογο. Cool, Olli Ludvigsen, Wolf Klintz, Pavanche Beres, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Peter Skinner, Arlene McCarthy. Oh. Well, and we won't get δεν θα έχουμε άλλους ομιλητές, ε, γιατί θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο. Πράγμα που το κάναμε και για τη δική σου έκθεση, Βέρνερ. Αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, θα χρειαστούμε και άλλη συνεδρίαση. Βίκη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που γράφει ο εισηγητής και με πολλά από τα σχόλια που έκανε σήμερα. Ε, να τον ευχαριστήσω επίσης ε, γιατί βλέπει και, και το θέμα της ε, ιδιοκτησίας και θα πω δύο λόγια για το trade finance ε, γιατί ε, το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι, ότι μιλάμε για πραγματικά ακίνητα και ότι υπάρχει ασφάλεια των συναλλαγών. Επίσης θα ήθελα να δείξει μεγαλύτερη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, και ότι το ε, άρθρο 129 θα πρέπει ε, ενδεχομένως να προσαρμοστεί αλλά πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούν και άλλοι τρόποι προσαρμογής και μη επιστροφή στη Βασιλεία 1. Συμφωνώ με τον Ούντο, δυστυχώς έφυγε πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και το δημόσιο χρέος εδώ γιατί το να το αφήσουμε στο Συμβούλιο ενδεχομένως εκεί να υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν και αυτό. Επίσης να προσθέσω ότι θα πρέπει να δούμε και το ενδεχόμενο κινδύνου που μπορεί να είναι πολύ χαμηλός όσον αφορά ε, τον κίνδυνο ε, ιδιοκτησίας και ενδεχομένως αυτό να προκαλέσει και αύξηση ε, του, του κόστους δανεισμού. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και κάποια καλύτερη διατύπωση όσον αφορά το επόμενο σημείο. Όσον αφορά τώρα ε, τα hedge funds που χρησιμοποιούν οι εταιρείε, ενδεχομένως αυτό θα πρέπει ε, να μπει στο CVA ε, αν και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό ίσως πάμε πολύ, ε, πολύ μακριά. Ε, στα παράγωγα των επιχειρήσεων πάντα μπορεί να υπάρχει κάποιος ε, κίνδυνος. Λοιπόν, ναι, βεβαίως θα πρέπει να δούμε το συμφέρον των μικρών μετόχων ή των, της μειοψηφίας. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η νομική δυνατότητα απέτησης του κεφαλαίου από άλλες ομάδες, αν και πιστεύω ότι ο εισηγητής ενδεχομένως έδωσε περισσότερη ε, ευελιξία από θα έπρεπε. Συμφωνώ επίσης με την ανησυχία του σχετικά με το πόσο εξουσία έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της διαδικασίας κατεπήγοντος θα πρέπει θα έπρεπε να δοθούν περισσότερες κατεξουσιοδότηση πράξεις και όχι οδός που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει συμφωνώ πάντως ότι θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε, υλοποιήσουμε αυτά που είχαμε βάλει στο πακέτο της ε, εποπτείας. Και όπως είπε και η Σάρον, ε, και εγώ πιστεύω ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε ε, βάσει του κατεπήγοντος. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία με τα οποία δεν συμφωνούμε. Ναι, βεβαίως χρειαζόμαστε ένα single rule book, αλλά ε, η εναρμόνιση και ο τρόπος εναρμόνισης δεν είναι πάντα σωστές. Και κατά αυτή την έννοια εξεφράστηκε ο κύριος Ντράγκη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, ορθολογιστές, να καταλάβουμε ότι οι πιστοτικές πραγματικότητε και ε, η οικονομία των τραπεζών είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διεκδικούν υψηλά πρότυπα ε, όπου είναι απαραίτητο. Ας πούμε, οι τροπολογίες που έχει υποβάλει ο εισηγητής ε, ε, στην ουσία μειώνει την δυνατότητα χρήσης ε, του, του μηχανισμού ε, απόσβεσης κινδύνων του buffer και το ECRB ενδεχομένως θα μπορούσε καλύτερα να ανταποκριθεί σε, αυτά τα, σε αυτές τις απαιτήσεις. Τώρα, εάν αλλάξουμε τον τρόπο ή τους στόχους εφαρμογής, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να μειώσουν το ρυθμό τους και δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι καλό όσον αφορά τη σταθερότητα των αγορών. Αναγνωρίζω πάντως ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο παρουσιάζει κάποιες ε, ε, ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να τις σκεφτεί έτσι η έκθεση Κάρας, αλλά παρόλα αυτά όσον αφορά ε, το μοντέλο ασφάλεια των τραπεζών είναι ε, γεγονός ότι μπορεί να μην ε, καταγράφεται στο ενεργητικό των τραπεζών γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα αλλά παρόλα αυτά ε, ε, εμένα με, ε, με ενδιαφέρει και το θέμα των μετόχων, αλλά με ενδιαφέρει και το θέμα των φορολογούμενων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταγράφονται σαφώς οι κίνδυνοι, έτσι ώστε όλοι να ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο και για την τράπεζα Lloyds αλλά και για άλλες τράπεζες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υποχρεωθούν έτσι ώστε να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους, έτσι ώστε τα στοιχεία όσον αφορά την, ε, τις επενδύσεις και όσον αφορά ε, την αποταμίευση να είναι σαφή. Ε, επίσης θεωρώ ότι η leverage ratio θα πρέπει να είναι, είναι σημαντική και επομένως θα πρέπει να δημοσιοποιείται και συμφωνώ με τον Ούντο ότι ε, όντως χρειαζόμαστε δημοσιοποίηση του stable finance ratio στην ουσία οι τράπεζες το κάνουν, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι ε, ενέχονται στις διαδικασίες αυτές και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της μεταρρύθμισης. Όσον αφορά ε, την ροή, ε, λέμε ότι οι ΗΠΑ δεν εφαρμόζουν τη Βασιλεία 2, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μην ξεχνούμε ότι η Βασιλεία 2 είναι πιο ασθενής από τη Βασιλεία 1 και επομένως ενώ θα πρέπει να επανέλθουμε στις ροές έτσι όπως αυτές προβλέπονται στη Βασιλεία 1. Ε, και μην ξεχνούμε ότι όντω δεν εφαρμόζουν οι ΗΠΑ, αλλά όχι μόνο οι ΗΠΑ ε, την Βασιλεία 2. Υπάρχουν και κάποιε αλλαγέ ε, οι οποίε αφορούν την Βασιλεία. Το Ordner Shares έχει γίνει capital instrument. Έχουν γίνει κάποιε αλλαγέ τέλο πάντων όσον αφορά τι ορολογίε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο άρθρο 25 ε, funds for General Banking Risk. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει εκεί να διορθωθεί λίγο η διατύπωση. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουμε αναφέρει. Ας πούμε όσον αφορά την αγορά κινήτων υπάρχουν μερικές χώρες όπου τα δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια ε, δεν ισχύουν ας πούμε, για το πρώτο τρίμηνο ή για τις 160 πρώτες μέρες. Δηλαδή ενδεχομένως ε, έχω χάσει τη δουλειά μου, αλλά παρόλα αυτά έχω έξι μήνες, δηλαδή δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να πληρώσω το δάνειό μου, αλλά ε, παρόλα αυτά δεν θέλω να πουλήσω το ακίνητο που μου ανήκει. Έχω έξι, έξι μήνες για να ξαναβρω δουλειά και να ξαναμπω στην αγορά. Ενδεχομένως, αν μειώσουμε στις 90 μέρες, στους τρεις μήνες, να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ε, όσον αφορά την τιτλοποίηση, την αγορά ε, θα πρέπει να δούμε ότι ενδεχομένως για κάποιους εκδότες ε, ε, εταιρείε αυτό θα μπορούσε να ε, προκαλέσει πρόβλημα. Βεβαίως, σαφώς δεν θέλω να επανέλθουμε στην κατάσταση αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης που έτσι όπως την έχει καταγράψει και η ΣΥΕΛΟ αλλά νομίζω ότι ε, θα πρέπει να, να, μένουμε σε επαφή και με τους ε, εκδότες ε, για να βλέπουμε ποιες είναι οι ανησυχίε τους. Συμφωνώ με τον Νούντο όσον αφορά την, τον κίνδυνο των, της χρήσης των αξιολογήσεων, αλλά δεν νομίζω ότι η επιστροφή στις εσωτερικές αξιολογήσεις θα μπορέσει να δώσει λύση στο πρόβλημα από τη μία άκρη δεν μπορούμε να πάμε στην άλλη. Βεβαίω λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στις, ε, στα κίνητα τα οποία Whether under covered structure. που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε ε, ε, το σύνολο της αγοράς και των τροπεζών. Με ενδιαφέρει, ένα στιγμή που με ενδιαφέρει με την κρίση αυτή είναι ότι όσο όλο και περισσότερο γίνεται μέσω εκλοπήσεων ε, οι, δανεισμοί και ε, υπάρχουν τράπεζες οι οποίες έχουν καλύτερη, καλύτερα περιουσιακά στοιχεία και άλλες με λιγότερο καλά περιουσιακά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ε, εάν έχουν υγιή ή τοξικά στοιχεία στα χέρια τους. Δηλαδή πρέπει να έχουν στοιχεία όσον αφορά την τράπεζα. και επίσης ε, θα πρέπει να δούμε ε, πώς είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το ποιοτικό ας πούμε ε, βήμα ε, αξιολόγησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Και αναρωτιέμαι μήπως θα πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο το θέμα του κατά πόσον οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ελάχιστες ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω τέλος πάντων ratio σχετικά με τα κεφάλαια τα οποία έχουν γιατί ε, εάν δεν ξέρεις ε, ε, κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία είναι καλά ή όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όταν αποφασίζει κανείς να επενδύσει ή όχι. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και στη συζήτησή μας όσον αφορά τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φιλίπ Λαμπέρ. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Δεν θέλω κι εγώ να αναφέρω όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία συμφωνώ με, τον, με την πρόταση του εισηγητού. Σας ευχαριστώ καταρχήν για, αυτή την για αυτό το πρώτο κείμενο και χαίρομαι που δεν το θεωρείτε τελικό κείμενο, αλλά το θεωρείτε σημείο αφετηρίας για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εκτιμώ ιδιαίτερα λοιπόν την προσπάθειά σας και την προσπάθεια ακριβώς να συνδέσετε αυτό το έργο σας με όλα τα άλλα τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμπστράκτο, ε, ξεκομμένο από όλα τα άλλα ε, προτείνεται. Το εκτιμώ λοιπόν αυτό. Σχετικά με αυτό που είπε η Δίκη για τις αξιολογήσεις και το πιστοτικό κίνδυνο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Είτε θα μιλήσουμε για τους οίκους αξιολόγησης, και δεν, θέλουμε να τους δώσουμε σχεδόν ρυθμιστικό χαρακτήρα ή βασιζόμαστε σε συστήματα εσωτερικής αξιολόγησης που δεν εμπιστευόμαστε. Και πρέπει να δούμε και τον δίκτυ μόχλευσης. Εδώ υποστηρίζουμε το να έχουμε δεσμευτικό δίκτυ μόχλευσης ε, στην νομοθεσία μας. Όχι απλώς διαφάνεια, αλλά δεσμευτικό δίκτυ, δίκτυ γιατί αυτό πραγματικά καλύπτει τον κίνδυνο. Πρέπει να υπάρχει ένα ε, όριο, πραγματικό όριο όμως κινδύνου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε να περιλαμβάνεται στην νομοθεσία. Ένα άλλο σημείο που δεν αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες ε, ε, διμερώς είχα συζητήσει με τον Ότμαρ ότι μετά τους προηγούμενους εισηγητές που έχουν κάνει αντίστοιχες εκθέσεις θέλουμε να έχουμε και ένα κανόνα κάρας με βάση, που θα ξεκινήσει από αυτή την έκθεση. Μου έκανε εντύπωση τις προάλλες που η αυτή αναφέρθηκε στον πλούτο σε σχέση με το City. Γιατί ε, βλέπουμε ότι υπάρχει καλή απόδοση όταν υπάρχει καλή διαχείριση. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε να έχουμε ως αποτέλεσμα και να δώσουμε κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτό το κείμενο μπορεί να αποτελέσει το σημείο στο οποίο θα μπουν αυτά τα θέματα. Για τις συστημικές τράπεζες ε, είπαμε ότι πρέπει να καλυφθούν και τώρα πρέπει να το κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το καθυστερήσουμε. κάποιος που είναι πολύ μεγάλος για να αποτύχει, ίσως είναι πολύ επικίνδυνος στο να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε, δεν ε, έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε. Τράπεζες που υπήρχαν πριν από την κρίση μπορεί να είναι ακόμη πιο συστημικές σήμερα και πιο επικίνδυνες. Δεν πρέπει να περιμένουμε καθόλου λοιπόν. Για τις απαιτήσει κεφαλαίου, Περισσότερο μια γραμμή του Λονδίνου είναι αυτή παρά μια γραμμή της υπόλοιπης Ευρώπης εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ ε, αντίστοιχα στοιχεία πρέπει να έχουμε και ως προς τη συγκέντρωση. Η Financial Times, νομίζω στο χτεσινό της φίλο ήταν, Αναφέρεται ο Wolf που λέει πρέπει να ε, έχουμε δίκτυ μόχλευσης κατά μέγιστον 10. Δεν προχωρούμε εμείς τόσο πολύ στις προτάσεις που κάνουμε αλλά πιστεύω ότι αυτούς τους κινδύνους πρέπει να αποφύγουμε. Μπορεί να είναι κάτι που ξεκίνησε από το Λονδίνο, αλλά και το Λονδίνο έχει πληγεί από την κρίση και επομένως κάποια σημεία τα έχουν καταγράψει ως σημείο πρέπει να εφαρμοστούν για να μην ε, έχουμε νέα κρίση. Για τον κίνδυνο ρευστότητας, άλλο ένα σημείο που υπάρχουν κάποιες δυσκολίες Συμφωνώ με κάποια από αυτά που είπαν ο και η Δίκη. Αλλά και πάλι εδώ είναι ένας τομέας που πρέπει να έχουμε δεσμευτικά μέτρα. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ε, κάποιο μεταβατικό περιθώριο για την εφαρμογή, αλλά δεν πρέπει απλώς να κάτσουμε και να κοιτάζουμε αυτούς τους δείκτες. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, αλλά χρειαζόμαστε και πιο συγκεκριμένα δεσμευτικούς δείκτες. Και το είπε και ο Ότμαρ, νομίζω, ότι το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης ήταν κρίση ρευστότητας και όχι κρίση φερεγγιότητας. Και υπό αυτή την έννοια πιστεύω ότι υπάρχει υπερβολικά μεγάλος κινδύνος ρευστότητας στο σήμερα αυτή τη στιγμή και κάτι πρέπει να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Επανέρχομαι στο μοντέλο εσωτερικής αξιολόγησης. Αν δεν μπορούμε ε, να απαλλαγούμε από αυτά, θα χρειάζεται μεγαλύτερη εποπτεία και benchmarking για τους κανόνες σχετικά με την αμοιβή. Ε, στη CRD3 ήδη κάτι είχαμε ε, ε, κάνει σχετικά με αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, πώς εφαρμόστηκαν αυτοί οι κανόνες, αυτές οι διατάξεις. Θεωρούμε ότι είναι επαρκείς αυτές οι διατάξεις, είναι αρκετά αυστηρές. Δεν είμαι βέβαιος. Αν κοιτάξουμε και πάλι το τι γίνεται στο Λονδίνο, πάλι υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καταλάβει ακόμη. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η παλαιά εποχή. Για, το για τη μέγιστη και ελάχιστη εναρμόνιση τώρα, χρειαζόμαστε κάποια ευελιξία. Συμφωνώ με όσους λένε ότι οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι ακριβώς ίδιες και η δομή της αγοράς δεν είναι ακριβώς ίδια στις διάφορες χώρες. Όμως θέλουμε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να παίζει ένα ε, ισχυρό ρόλο παρακολουθώντας και διαχειριζόμενη τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Δεν θέλουμε να είναι κάτι το οποίο θα είναι ανοιχτό προς όλους και έτσι να πλήττεται η εσωτερική αγορά. Οποιαδήποτε παρέκκληση από τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και θα πρέπει να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας του κοινού μας συμφέροντος εδώ. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα θέματα που θέλουμε να αναφέρονται. Είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ως προς το τι μπορούμε να επιτύχουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι κάτι το οποίο θα έχει και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να δοκιμάσει, να δει πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά το φιλόδοξο κείμενο, αλλά να μην μείνετε σε κάτι ε, μετριοπαθές. Προσπαθήστε να δοκιμάστε τις αντιδράσεις για να δείτε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε και να μην χάσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Ε, ο Ευρωπαίος νομοθέτης δεν θα υποταγεί στις ε, επιθυμίες του Αμερικανικού Κογκρέσου, εμείς θα πρέπει να δούμε τι είναι προς συμφέρον της Ευρώπης. Και πολλές φορές είναι προς συμφέρον μας οι πιο αυστηροί κανόνες. Και αν δείτε τι έχει κάνει το Λονδίνο μετά την κρίση, πώς θέτει δεσμευτικούς κανόνες για τη ρευστότητα κλπ. Βλέπετε το Λονδίνο το είπε ότι το θέλουμε, θέλουμε τις ρυθμίσεις ε, γιατί είναι προς συμφέρον μας. Ίσως υπάρξουν και ανεπιθύμητες ενέργειες, ε, αλλά το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ρυθμιστικές αρχές στο Λονδίνο είναι ότι τελικά η θέση που ακολούθησαν ήταν ε, θετική ως προς τον ανταγωνισμό. Το ότι είχαν αυστηρότερες διατάξεις ήταν θετικό για τον ανταγωνισμό. Θέλουμε κανόνες που θα κάνουν την αγορά μας και τον χρηματοπιστωτικό τομέα περισσότερο ελκυστικό, ε, περισσότερο ανθεκτικό ε, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κεφάλαια. θα είναι ασφαλέστερες οι αποδόσεις μας στην Ευρώπη, ακόμη και αν είναι μικρότερες και οι επενδυτές θα γνωρίζουν ότι σε αυτή την αγορά τουλάχιστον θα είναι ασφαλής. Θα, μπορούν, ε, θα μπορεί η απόδοση την οποία περιμένουν να είναι προβλέψιμη και σταθερή. Και αυτό νομίζω ότι είναι παράγον εμπιστοσύνη. Αυτά λοιπόν ήθελα να σα πω. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα και θα συνεχίσουμε ω συνήθω να δουλεύουμε σκληρά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με τον κατάλογο ώστε να καλύψουμε τους περισσότερους δυνατών αγορητές. Ε, Κόριν, η επόμενη είσαι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Οτμαρ Κάρας για το έργο που επετέλεσε, προετοιμάζοντας το σχέδιο έκθεσης. Έκθεσης που γενικά, σε γενικές γραμμές θα ήθελα να το υποστηρίξω πλήρως και να δούμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερις τομείς όπου νομίζω τουλάχιστον χρειάζεται από αυτόν περισσότερη δουλειά για να εξειδικευθούν. Πρώτον, θα ήθελα να σχολιάσω την πρόσφατη αβεβαιότητα από πλευράς του Συμβουλίου με συγκεχημένα μηνύματα σε σχέση με το ε, σι αντί τέσσερα αν είναι προτεραιότητα ακόμα ή όχι. Δεν ξέρω πώς πρέπει να ερμηνευθούν ε, οι κλήσεις από την Γερμανία και την Γαλλία σε σχέση με την καθυστέρηση αυτού του πακέτου και γι' αυτό δημιουργείται σύγχυση. Αφενός ζητάμε 9% ποσοστό ρευστότητας το δυνατόν πιο γοργά για τις τράπεζες που βρίσκονται υποδοκιμασία υπό διαδικασία δοκιμής. Δεν είναι απόλυτα σαφές πώς αυτό θα υλοποιηθεί όμως ε, σήμερα και γι' αυτό είναι κατεπίγουσα ανάγκη πιστεύω να δώσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια στις αγορές. Ασφάλεια και βεβαιότητα για το πώς αυτό το ποσοστό ρευστότητας θα υλοποιηθεί και θα διαμορφωθεί και αυτό μπορεί να συνεισφέρει για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Βλέπουμε ήδη κάποιες κινήσεις στις αγορές ε, που αφορούν συγκεκριμένα τέτοια ε, κεφάλαια που ίσως δεν θα ε, ελαμβάνονται υπόψη και γι' αυτό αυτές είναι εξελίξεις προς την εσφαλμένη κατεύθυνση αντί προς την ορθή κατεύθυνση. Έχει τεράστια λοιπόν σημασία να διατηρήσουμε την ε, προτεραιότητα για το 4 και να πάμε και ένα βήμα παραπέρα ακόμα αν γίνεται είναι τόσο σημαντική αυτή η προτεραιότητα σε σχέση με την εισφορά των συμμετοχή των τραπεζών. Εκείνοι που θέλουν να καθυστερήσουν την εφαρμογή του CRD4 και θέλουν <clears throat> να υλοποιηθεί ήδη νωρίτερα ένα σύστημα εισφορών των τραπεζών, συμμετοχής των τραπεζών είναι λανθασμένο θα πρέπει να ενισχυθεί ο τραπεζικός τομέας είναι ο καλύτερος τρόπος για να διεξέλθουμε από την χρηματοοικονομική κρίση. Βήμα προς βήμα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Δεν είμαι κατά του banking levy, δεν είναι αυτό εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω. Είναι όμως το ότι είναι ανάγκη να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις προτεραιότητες ε, που θα θέλαμε να επιτευχθούν. Δεύτερο, για το που στοχεύουμε και θα πορευθούμε. Μία ευρωπαϊκή, Μια ευρωπαϊκή, μια παγκόσμια προσέγγιση σε κάποιους τομείς μπορούμε να πάμε παραπέρα. Δεν θα είχα πιο προβλήματα να γινόταν κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να σχολιάσω όμως το, τη γραμμή του μέγιστου εναρμονισμού που πρότεινε στην έκθεσή του Ότμαρ Κάρας. Συμφωνώ με αυτή την πρόταση αυτή τη πορεία μέγιστου εναρμονισμού. Ξέρουμε όμω ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητε και συγκυρίε σε κάποια κράτη και για κάποια είδη τραπεζών που θα πρέπει να λάβουμε τα πράγματα υπόψη και να δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε πιο πέρα. Είναι πολύ σημαντικό το να περιοριστεί το θέμα του να ξεπεράσουμε αυτό το πλαίσιο και να πάμε σε ένα μέγιστο εναρμονισμό. Σε σχέση για παράδειγμα με τις Ολλανδικές τράπεζες, να ξεπεράσουμε τα εσκαμμένα των κριτηρίων του C αντί 4 αν χρειάζεται. Δεν πρέπει να επισέλθουμε σε κάτι τέτοιο τώρα. Χρειάζονται σαφή κριτήρια και ένα σαφής ρόλος ε, για, ε, ε, για να εξεταστεί το θέμα αυτό και η ελαστικότητα που επιτρέπεται και που όχι. Διότι επιθυμούμε η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά να σέβεται αυτές τις προδιαγραφές κατά το μέγιστο. Τρίτο θέμα, η ρευστότητα. Και εδώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν από την Βίκη Φοντ και άλλους, ότι πρέπει να δούμε σε βάθος περαιτέρω τους ορισμούς και προσδιορισμούς ε, των θεμάτων ρευστότητας και coverage rates ε, των ε, ποσοστών κάλυψης. Ξέρω ότι προαναφέρθηκε το θέμα υπάρχει ανοιχτό πνεύμα να προχωρήσουμε δεν καλύπτεται ακόμα από την έκθεση για να σας δώσω όμως ένα σαφές παράδειγμα το να πει κανείς ότι για κάθε καλυπτόμενο ομόλογο το ότι βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και να μην λέει κανείς ότι ε, για κάθε ε, δυνατότητα ασφάλειας όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια πρόκειται για ένα subprime ε, μη ευρισκόμενο στο επαρκές επίπεδο αγαθό Πρέπει να δούμε αυτή τη διαφοροποίηση. Όταν λέμε το ένα είναι καλό, το άλλο είναι κακό και έτσι δεν μπορεί να συμπεριληφθεί, αυτό θα δημιουργήσει, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη. Και δεν είναι νομίζω αυτό το οποίο είναι καλά θεμελιωμένο και τεκμηριωμένο να γίνει. Χρειαζόμαστε όλοι υψηλή ποιότητα αγαθά και, ε, και κτημένα. Και κάτι άλλο, όταν καταλήγουμε σε ένα ίδιο πλαίσιο μπορεί να δημιουργηθεί ένας νέος συστημικός κίνδυνος. Θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω υπέρ της πολυμορφοποίησης με σαφή όμως κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας και αυτό εντάσσεται σε αυτά τα οποία προανέφερε η Βίκη και ο Φιλίπ και ίσως από κοινού με τον εισηγητή μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να τα εξειδικεύσουμε περαιτέρω. Τελευταίο θέμα για την διαχείριση, εταιρική διαχείριση και ε, υπευθυνότητα corporate governance. Συμφωνώ με τα όσα προαναφέρθηκαν. Πρέπει να δούμε οπωσδήποτε σε σχέση και με την πολιτική αμοιβών να ευθυγραμμίζεται με τα μακροπρόθεσμα θεσμικά συμφέροντα ενός θεσμικού οργάνου. Θέλουμε μια μακροπρόθεσμη ε, κερδοφορία και ε, βιωσιμότητα και όχι βραχυπρόθεσμα κέρδη πρέπει να προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε περισσότερο αυτούς τους στόχους. Κάποια κράτη-μέλη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όχι. Όλα αυτά δημιουργούν συνολικά κάποιες συγκεχημένες απόψεις και ένα συγκεχημένο πλαίσιο. Και σε αυτό το πεδίο πρέπει να συνεργαστούμε για τον εναρμονισμό στο ορθό επίπεδο ποιότητας που θα συμφωνηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ώστε να εξειδικευτεί η πολιτική αμοιβών με πιο συγκεκριμένα κριτήρια και μπορεί αυτό να γίνει με μια οδηγία όπως και στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Όλοι Λότβιξεν. Δεν θα μπορέσουν ίσω όλοι να μπορέσουν να παρέμουν σήμερα. Είναι ένα όμω τόσο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που πρέπει να μπορέσουμε να παρέμβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και σήμερα περισσότεροι και μετά να δοθεί συνέχεια ιστερότερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή παρουσίαση από πλευράς του. Έχω και κάποιες δικές μου ξεχωριστές απόψεις, όμως θα ήθελα την αρχή της μέγιστης της να την αμφισβητήσω σε, ε, στη δική μου παρέμβαση. Δεν ανταποκρίνεται σε σχέση με τη Συμφωνία Βασιλείας 2 για τα μέγιστα όρια όσον αφορά την κάλυψη για τις απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων σε σχέση λοιπόν με τη διαδικασία Βασιλείας 2 και επίσης και δεν είναι και καθόλου ο στόχος εξάλλου αυτής της συμφωνίας ε, όσον αφορά την αύξηση της σταθερότητας θα πρέπει λοιπόν να το δούμε ξεχωριστά αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός τραπεζικός τομέας αν ακολουθηθεί μια τέτοια κατεύθυνση θα αποδυναμωθεί, θα αποσταθεροποιηθεί και θα υπάρξουν και μεγάλοι κίνδυνοι για τους φορολογούμενους, μεγάλο βάρος που θα επομίζονται και δεν είναι και το σωστότερο και πρόκειται και για το θέμα της εφαρμογής και υλοποίησης. Με ποιο ρυθμό ταχύτητας ή βραδύτητας θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Εξάλλου, υπάρχουν κάποια άλλα κράτη, κάποια κράτη-μέλη τα οποία προτίθενται ή μπορούν να ακολουθήσουν με ταχύτερους ρυθμούς την πορεία αυτή. Ε, λέει ο εισηγητής ε, ε, και πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να τηρεί τον ρυθμό εκείνο που είναι ε, ε, το, πιο εφικτό να ακολουθηθεί από πλευράς αυτού του κράτους. Να μην επιταχύνονται δια της βίας ή επιβραδύνονται δια της βίας. Αν μπορεί κάτι να γίνει δηλαδή να γίνεται με τον σωστότερο τρόπο. Το όριο λοιπόν της υπερχρέωσης. Υπάρχει εδώ αναγκαιότητα εκ και της προσπάθειας εποπτείας. Όμως μέχρι το 2015 όλα αυτά να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν για παράδειγμα με την τέξια είδαμε ότι το ποσοστό υπερχρέωσης δεν ήταν πάντα το ε, σωστότερο όσον αφορά τα, τις ε, δράσεις ε, ε, αυτού του οργανισμού. Διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι ήταν 60% του ιδίου κεφαλαίου η υπερχρέωση. Ήταν δηλαδή, ας το πω έτσι, πραγματικό πλήγμα αυτό και θα πρέπει σε προημότερο στάδιο, σε προημότερη φάση να μπορούν αυτά να διαπιστώνονται και να προσδιορίζονται. Από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρθηκε ότι πρέπει να ενισχυθεί η τραπεζική εποπτεία. Αντί όμως τώρα να μεταβληθούν ή να αναβληθούν, να επεκταθούν οι προθεσμίες, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να διατεθούν τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη στοχοθέτηση αυτή Έχω όμως την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά της μάλλον διστάζει και είναι επιφυλακτικότερη σε σχέση με την ε, αναγκαιότητα διασφάλισης των αναγκαίων στελεχών για να γίνουν αυτές οι δράσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή λέει η κυρία Μπερές, μας επιτρέπει η πρότασή του να καταλάβουμε καλύτερα την πρόταση ε, και το τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Ε, έχω ένα κατάλογο σημείων και θα αναφέρω τα πιο σημαντικά. Καταρχήν, για το θέμα των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Ε, και βέβαια είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα επί του οποίου θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να λάβουν θέση. Άκουσα τι είπατε, Πρόεδρε, ότι δεν είναι το βασικό θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι το βασικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ε, μπορεί να μιλά συνέχεια για την ανταγωνιστικότητά της χωρίς να θέτει το ερώτημα ε, της ανταγωνιστικότητας στον τραπεζικό τομέα έναντι του υπολείπου κόσμου. Και υπενθυμίζω ότι στην έκθεση για την κρίση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του συμπεράσματος των συμφωνιών τη Βασιλείας 2 για τη μορφή των συνθήκων. Το θέμα της αμοιβαιότητα λοιπόν τίθεται και δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε. Ε, για να έχουμε την ε, αμοιβαιότητα θα πρέπει ε, να ορίσουμε κάποια εντολή για τους επόπτες ούτως ώστε να υπάρχει ένας πίνακας προειδοποίησης κάθε φορά που δεν θα εφαρμόζονται οι συμφωνίες, ιδίως από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι μόνο αμερικανικό βέβαια το πρόβλημα, αλλά έχει προτεραιότητα το αμερικανικό πρόβλημα ε, και μάλιστα διότι έχει επιπτώσεις στις διατλαντικές συναλλαγές. Τώρα για το θέμα του ορισμού της ρευστότητας. Ίσως δεν ε, κατάλαβα ε, καλά αυτό που είπατε. Ε, νομίζω ότι είπατε κύριε Καράς ποια είναι η φιλοσοφία σε σχέση με το νομικό μέσο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει μια συζήτηση ώστε να γνωρίζουμε στο τέλος, μετά την έκθεση και την εκθέταση της κατάστασης, ε, για το αν θα πρέπει να καθορίσουμε τα κριτήρια απαιτούμενη ρευστότητα και αν αυτό θα πρέπει να γίνει με νέο κανονισμό ή αν ε, θα πρέπει να γίνει με ε, νομοθεσία δευτέρου επίπεδου είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε γιατί αυτό το οποίο θα βάλουμε στην πρώτη έκθεση θα είναι διαφορετικό από ότι ε, ε, ε, στις δύο περιπτώσεις αν είναι κανονισμός ή αν είναι δεύτερου επίπεδου. Και επανέρχομαι στο μηδενικό κίνδυνο του δημοσίου χρέους. Άκουσα προσεκτικά αυτό που είπατε σε σχέση με τον κίνδυνο μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων, αλλά εγώ μιλώ για τον κίνδυνο ρευστότητα. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν κατανοώ στην παρούσα κατάσταση. Ο μηδενικό κίνδυνο που δεν είναι μηδενικό κίνδυνο στην αγορά δημοσίου χρέου, νομίζω ότι και ένα δεκάχρονο παιδάκι θα το καταλάβαινε. Αλλά το ότι την 1η Ιουνίου του χρόνου και ελπίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών από μόνη της έχει πει ότι την 1η Ιουνίου του 2012 θα υπολογίζεται η αγοραστική αξία του δημοσίου χρέους και είναι κάτι το αδιανόητο. Για τη ρευστότητα διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται πλήρη ταραχή στις αγορές και δεν μας επιτρέπει η αρμπιτράζ σήμερα και θα προχωρήσουμε όπως κρίνουμε περισσότερο ορθό. Και σε περιπτώσεις ε, αμφιβολίας ε, και ακραίων πιθανότητων θέλουμε να βάλουμε μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ε, για να δούμε πώς θα περάσουμε σε ένα full market risk. Πρέπει να δούμε τι ενδείξεις δίνουμε εμείς στην έκθεση Κάρας. Πιστεύω ότι περισσότερο συνετό θα ήταν να χειριστούμε το θέμα της αποτίμησης του δημοσίου χρέους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και, με το, κριτήριο ρευστότητας. Να γίνεται μια εξέταση για να μπορεί να γίνει το αρμπιτράζ. Ένα τρίτο σημείο, που, τέταρτο μάλλον που θέλω να αναφέρω, είναι το θέμα του διαχωρισμού των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Δεν είναι πια εδώ ο Φιλίπ Λαμπέρ, αλλά συμφωνώ 100% με αυτά τα οποία είπε. Οπουδήποτε μπορούμε να αποφασίσουμε να το βάλουμε, αλλά είμαι βεβαία ότι η έκθεση Κάρας αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για να μπορέσουμε να περάσουμε στο θέμα του διαχωρισμού των ε, τραπεζών καταθέσεων και των ε, επιχειρηματικών τραπεζών, εμπορικών τραπεζών. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, μια σημαντική συνεισφορά του Κοινοβουλίου σε αυτό τον τομέα. Πέμπτο σημείο, το θέμα των οίκων αξιολόγησης. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ε, κάτι που μας πάει πίσω σε σχέση με το Βασιλεία 2. Εγώ διαφωνούσα με τον Αλεξάνδερ Άντβαν όταν είχε αποδεχθεί μια επίσημη ε, δημοσίευση των ε, οίκων αξιολόγησης και μια υπερβολική ε, εξάρτηση από τους οίκους αξιολόγησης. Δεν θα πρέπει να βάλουμε καμία αναφορά στο ρόλο των οίκων αξιολόγηση στην έκθεση Κάρα, στη βασική νομοθεσία υπό αυτή την έννοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παίζουν κανένα ρόλο ή και αξιολόγηση, αλλά δεν θα νομιμοποιούνται, δεν θα τους έχει νομιμοποιήσει ο νομοθέτης. Και υπό αυτή την έννοια θα βρισκόμαστε σε σύμπνοια, σε με αυτό που κάναμε στην έκθεση Λαροζιέρ, όπου αυτό το θέμα ήταν ένα από τα θέματα που εξετάζονταν. Τέλος, για την ε, πλήρη ή μη πλήρη εναρμόνιση, ε, των ορισμών των ιδίων κεφαλαίων. Θα είναι αρκετά δύσκολη αυτή η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα από το Βασιλεία 2 και θυμάστε τις συζητήσεις που κάναμε τότε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε φορέα και ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι ο κόσμος των συνεταιριστικών τραπεζών ε, γνωρίζει τώρα το τι είχαμε αποφασίσει με βάση το Βασιλεία 2, αλλά παραμένουν κάποιες προσαρμογές για τα πιστοποιητικά, παραδείγματο χάρη μου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να αναφέρω όλα τα σημεία. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι διερμηνήσεις θα μας δώσουν άλλα πέντε λεπτά, μας είπαν να ρωτήσω τον εισηγητή. Θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις ή να ακούσουμε μια επόμενη ερώτηση από την Ελίζα Φερέιρα. Ελίζα. Πέντε λεπτά και μετά θα μπορούμε μόνο αγγλικά να συνεχίσουμε, αν συνεχίσεις να μιλάς. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κάποια από τα θέματα τα οποία ήθελα να καλύψω ήδη προαναφέρθηκαν και καλύφθηκαν από άλλους συναδέλφους πριν από μένα. Όμως Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έργο το οποίο επιτελέσατε, διότι πραγματικά είναι σημαντικό για αυτή τη συζήτηση που ανοίγεται με όλους μας, διότι αυτό το θέμα είναι κέρια σημασία, ζωτική σημασία και περίπλοκο ταυτόχρονα. Θα αναφέρω μόνο εξειδικευμένα κάποια θέματα για να υπενθυμίσω αυτό το οποίο προαναφέρθηκε πριν. Το θέμα της αμοιβή είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, πράγματι η πραγματική οικονομία και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε θα καλυφθεί. Το κρατικό χρέος φυσικά είναι ένα άλλο και η ρευστότητα ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα υπό τις, τις πτυχές της ρευστότητας που μέχρι τώρα δεν έχουν επαρκώς ε, καλυφθεί και που υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης ε, για την εξειδίκευση αυτών των προτάσεων για την ρευστότητα. Τώρα, για κάποια άλλα θέματα που θα ήθελα να επικεντρωθώ. Ένα από αυτά είναι ο συσχετισμός του CRD4 και των συστημικών θεσμών και θεσμικών οργάνων και η διαχείριση της κρίσης, αντιμετώπιση της κρίσης μέσα από αυτές τις προτάσεις. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να καλύψω αφορά μια πολύ συγκεκριμένη εξειδικευμένη περίπτωση που όμως έχει τεράστια σημασία για κάποια πρότυπα επιχειρησιακά και αυτό σχετίζεται με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μη λειτουργικού χαρακτήρα εταιρείες και τα θέματα των ε, μειοψηφικών δικαιωμάτων μεριδιούχων. Αυτό σε σχέση με την τροπολογία 40 νομίζω μερικά καλύπτεται, αλλά είναι σημαντικό από την άλλη πλευρά για κάποιες ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η πτυχή, να ενισχυθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοιες εταιρείες που έχουν δικαιώματα μειοψηφιών, μειοψηφία ε, στον τραπεζικό τομέα, σε τραπεζικές τέτοιες δραστηριότητες, που όμως αυτών αυτές οι εταιρείες δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και εξακολουθούν να έχουν την μορφή μη ε, ε, δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων. Υπό αυτό τον όρο απαιτούνται κεφάλαια για αυτές τις εταιρείες. Κεφάλαια τα οποία, για τις εταιρείες που δεν παρεμβαίνουν άμεσα σε αυτές τις τραπεζικές δραστηριότητες. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί και να ρυθμιστεί, διότι η νομοθεσία προετοιμάζεται για εταιρείε, για τραπεζικές ιδιωτικούς ομίλους και επιχειρήσεις που αυτών ασχολούνται με τέτοιες τραπεζικές ε, επιχειρήσεις. Πρέπει όμως να δούμε και το θέμα των προβλημάτων που δημιουργούνται στον τραπεζικό τομέα όταν έχουμε μη καθορισμένες τέτοιες εταιρείες που όμως λόγω μειοψηφικών δικαιωμάτων ε, από πλευράς τραπεζικών ε, επιχειρήσεων, ε, δραστηριοτήτων δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό έχει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα όταν οι τράπεζες βλέπουμε ότι μετεξελίχθηκαν από κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις και έχουμε επιχειρήσεις μεριδιούχων ε, όπου έχουν ε, μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης. Ε, αφ' όμως δεν απαιτείται από πλευράς τους λόγω των ε, διατάξεων και ορισμών να έχουν τα υπαρκή κεφάλαια όπως άλλες τράπεζες, ε, καθαρόεμες τράπεζες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πτυχή των επιχειρήσεων στις οποίες εμπλέκονται και θα ήθελα συγκεκριμένα, εξειδικευμένα να αναφερθεί και να καλυφθεί αυτό το θέμα και να ρυθμιστεί σε σχέση με τα άλλα θέματα με τα οποία ξεκίνησα την παρέμβασή μου θα ήθελα να προσυπογράψω αυτή την κατεύθυνση και να συμφωνήσω με τα προαναφερθέντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας εδώ και τώρα τώρα. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι ε, τον ε, Φεβρουάριο του 2012 ε, οι όσοι θέλουν περαιτέρω να παρέμβουν θα πρέπει να βρεθεί κάποιο χρονικό διάστημα στις εργασίες μας άλλη συνεδρίασης ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και να ακούσουμε και τις απόψεις του εισηγητή επ' αυτών. Σας ευχαριστώ όλους.